Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινούμε τη συνεδρίασή μας. Και χαιρετίζουμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης της ε, Ισπανίας, που όπως ξέρετε έχει το εξάμεινο Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ακούσουμε από το στόμα του τις ε, κατευθυντήρες γραμμές της Ισπανικής Προεδρίας για το τρέχον εξάμεινο. Πρωτού ξεκινήσουμε σε σχέση με το θέμα που συζητήσαμε χθες στη συνάντηση των συντονιστών και που αφορούσε την ε, κατανομή την, ε, μάλλον την απόδοση του, της ηγεσία των φάκελο SWIFT για τη σύνταξη γνωμοδότησης και συμπερασμάτων. Η σοσιαλιστική ομάδα θα αναλάβει αυτό το φάκελο και δίνω το λόγο στην Κίνγκα Κόνς. Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση μονάχα. Κάναμε μια μακρά συζήτηση χθες για το ποιος θα ήταν ο εισηγητής για το SWIFT και η απόφασή μας είναι να αποσύρουμε την αίτησή μας να αναλάβουμε το SWIFT γιατί προτιμούμε να πάρουμε το, την έκθεση για την προστασία των πολιτών όπως συζητήσαμε και χθε Και και αυτό το θέμα εκκρεμεί. Ευχαριστώ κυρία Κάνς. Οπότε περνούμε στο πρώτο σημείο της ημέρας διάταξης που είναι η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Ισπανικής Προεδρίας από τον Υπουργό Δικαιοσύνης της Ισπανίας. Για 15 περίπου λεφτά έχετε το λόγο και στη συνέχεια, όπως χθε θα κάνουμε ένα πρώτο γύρο παρεμβάσεων από τους συντονιστές, ένα συντονιστής από κάθε πολιτική ομάδα και μετά ένα ανοιχτό γύρο ανοιχτό σε όλου του βουλευτέ, οι οποίοι μπορούν να ερωτούν και θα απαντά ομαδικά στι ερωτήσει του ο κύριο Υπουργό. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, καλημέρα σα σε όλου και σε όλου. Έχω την τιμή να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ισπανικής Προεδρίας στον τομέα της δικαιοσύνης και το πράτο με γνώση της φιλοδοξίας που περιέχεται αλλά και της ε, ευθύνης που έχουμε να αναλάβουμε. Είναι η μέρα με την οποία ήδη ε, θυμούμαστε τα θύματα του ολοκαυτώματος. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρισκόμαστε σε μια νέα φάση. Με τη της Λισαβόνας έχουμε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο μας επιποχρεώνει να εργαστούμε έντονα, προσπαθώντας να βρούμε λύσεις προς όφελος των πολιτών, τι κατάλληλε δεσμεύσει, που πιστεύω ότι θα βρουν στην ε, <clears throat> Ισπανική Προεδρία ένα συνομιλητή πάντα διαθέσιμο να ακούσει την άποψή τους. Επίσης, συμπίπτει η ανάληψη της ε, Προεδρίας με ένα νέο <clears throat> Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχουμε νέες μεθόδους εργασίας, έχουμε ένα διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχουμε μόνο ένα νέο κανονιστικό πλαίσιο λόγω της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά επίσης και λόγω της υποχρέωσης να αναπτύξουμε και να εξελίξουμε το πενταετές πρόγραμμα 2009-2014 γνωστό ως πρόγραμμα της Στοχόλμης στον τομέα των εσωτερικών δικαιοσύνης και ελευθερίας. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την απαράγραπτη συνέχεια στη δράση μας και με αυτό το στόχο έχουμε προετοιμάσει την Προεδρία αυτή μαζί με τους εταίρους μας, το Βέλγιο και την Ουγγαρία, που απαρτίζουν την Τρόικα. Έχουμε λοιπόν εξασφαλίσει να έχουμε μια διαδικασία στην οποία θα αποδώσουμε τόση μεγάλη σημασία όσο και στα αποτελέσματα των ενεργειών μας. Θέλουμε λοιπόν καταρχήν η νέα Κομισιόν να μην καθυστερήσει στην παρουσίαση των νομοθετικών της προτάσεων που φυσικά έχουν μείνει ε, εκρεμείς διότι είχαν παρουσιαστεί προηγουμένω με τις προηγούμενε συνθήκες, με την προηγούμενη συνθήκη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θέλουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια με τι συμφωνίε που έχουν επιτευχθεί μέχρι τώρα στο Συμβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα εκμεταλλευτούμε τι συμφωνίε που έχουν επιτευχθεί και να, θα αποφύγουμε με τον τρόπο αυτό η συνθήκη της Λισαβόνα να οδηγήσει σε χρονοτριβή και παράλυση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπορέσουμε λοιπόν να προωθήσουμε θέματα τα οποία την χάνουν ευρεία συνένεση ε, μας ενδιαφέρουν θέματα όπως η μετάφραση και η διερμηνία μέσα στα πλαίσια των διαδικαστικών διαδικασιών στα δικαστήρια και επίσης θέματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλική κακοποίηση των ανηλίκων και την πορνογραφία στο διαδίκτυο. Επίσης θέλουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με το PNR στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι αφιβολίες που έχουν εκφραστεί στο παρελθόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως σε σχέση με την αρχή της αναλογικότητας ό,τι αφορά την ε, χρήση του ΠΕΝΕΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν τώρα η Κομισιόν <clears throat> επανέλθει με την παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας για την οποία έχει ήδη εργαστεί το Συμβούλιο και την έχει επεξεργαστεί, είμαστε εν επιγνώση ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διαβούλευση και αναζήτηση συμφωνίας μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στην απαραίτητη ισορροπία μεταξύ των αναγκαιοτήτων της ασφάλειας που προφανώς υπάρχουν και δικαιολογούν το μέτρο αυτό, αλλά κυρίως και των απαιτήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο προβλέπεται εκφρασμένα στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το οποίο έχει την ίδια νομική ε, <clears throat> ισχύ όπως και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά θα απαιτήσουν πιο έντονη εργασία από την πλευρά μας. Αυτό δεν είναι ποτέ πρόβλημα όμως. Θέλουμε να τονίσουμε ότι είμαστε έτοιμοι να επανέλθουμε σε όλες αυτές τις εκκρεμίες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων θέλω να υπογραμμίσω λόγω της σημασίας της για τους πολίτες την πρωτοβουλία για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών σε ό,τι αφορά την ε, ποινική δικονομία και τις εγγύησεις που συνάπτονται με την ποινική δικονομία. Μετά από τις συζητήσεις του, του, περασμένου έτους, το Συμβούλιο κατέληξε σε ένα φύλλο πορείας για τα θέματα αυτά, ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα, το οποίο δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε. Η Τρόικα Προεδριών και ιδιαίτερα η Ισπανική Προεδρία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα <clears throat> να προχωρήσει προς την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας. Γιατί πιστεύουμε με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών αρχών των κρατών μελών και έτσι να εξασφαλίσουμε να υπάρχει μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή των εργαλείων δικαστικής συνεργασίας που ήδη υπάρχουν στο χώρο ελευθερίας, δικαιοσύνης και ασφάλειας. Το πρώτο λοιπόν από τα μέτρα τα οποία προβλέπουμε σε σχέση με τα δικαιώματα μετάφασης και διερμηνίας στην ποινική δικονομία έχει ήδη ξεκινήσει με βάση μια πρωτοβουλία των κρατών μελών, ξεκινώντας από την πολιτική συμφωνία η οποία επετέφθη τον Οκτώβριο του 2009 στο Συμβούλιο. Ως Ισπανική Προεδρία θεωρούμε ότι είναι εφικτό να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το νομοθέτημα που με τον τρόπο αυτό θα είναι το πρώτο νομοθέτημα το οποίο θα έχει εγκριθεί με την νέα διαδικασία στα πλαίσια της δικαστικής συνεργασίας. Είμαστε δεσμευμένοι λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Πιστεύουμε ότι μια ταχεία συμφωνία για αυτή την οδηγία θα είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε το έργο μας και να υλοποιήσουμε την, τον οδικό χάρτη που ανέφερα προηγουμένως. Η Ισπανική Προεδρία θα επιμείνει ενώπιον της Κομισιόν ώστε η πληροφόρηση των κρατουμένων για τα δικαιώματά τους και η σχετική οδηγία να εγκριθεί μέχρι το τέλος αυτού του εξαμήνου. Όπως είναι γνωστό, η συνθήκη της Λισαβόνας ενισχύει τη λογική αξιολόγηση των πολιτικών στον χώρο της ασφάλειας, δικαιοσύνης και ελευθερίας. Θεωρούμε λοιπόν, όπως έγινε σαφές και στο άτυπο Συμβούλιο του Τολέδου, ότι αυτή η αξιολόγηση δεν πρέπει να γίνει πρόσχημα για την παράλυση της νομοθετικής διαδικασίας, ούτε πρόσχημα για να επικαλύπτεται η προσπάθειά μας με αυτή άλλων θεσμών όπως είναι η Κομισιόν για την η Επιτροπή μάλλον για τα δικαστικά θέματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ούτε επίσης θα πρέπει εμείς να καταδεικνύουμε ποια είναι τα προβλήματα στην κοινή γνώμη, γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αντιπαραγωγικά αποτελέσματα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, ένα από τα βασικά στοιχεία της ταυτότητας της Ισπανίας από την εποχή της εισόδου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η προσήλωσή της για να δημιουργηθεί ένας αυθεντικός χώρος δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας προς το όφελος όλων των πολιτών. Είμαστε πιστοί σε αυτή την πεποίθηση και η Ισπανική Προεδρία είναι αποφασισμένη να προωθήσει όλες τις πρωτοβουλίες οι οποίες εγγράφονται μέσα στο πλαίσιο αυτού του εγχειρήματο, διότι έχουμε και επίγνωση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η Δίκη της και το πρόγραμμα τη Στοχόλμη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι κύριε γραμμέ κατεύθυνσή μα είναι οι εξή. Πρώτα απ' όλα, <clears throat> να ενισχύσουμε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και να διευρύνουμε του διάβλους που είναι ανοιχτοί στου Ευρωπαίου πολίτε, ώστε να ασκήσουν πληρώ τα δικαιώματά του χωρί να πλήττονται από την πολυμορφία των εθνικών πρακτικών και των συστημάτων ένομης τάξης. Δεύτερον, να βελτιώσουμε την απόδοση δικαιοσύνης και την διαχείριση της δικαιοσύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τρίτον, να βελτιώσουμε τα εργαλεία για να μπορέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο να αντιμετωπίσουμε το έγκλημα, την τρομοκρατία και το οργανωμένο ιδίω έγκλημα, πάντα όμως με στα πλαίσια των νομικών και δικαστικών εγγύσεων. Τέλος, να προχωρήσουμε στη δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες. Η δραστηριότητά μας λοιπόν θα υλοποιηθεί στα εξής εγχειρήματα. Πρώτον, να εγκρίνουμε το σχέδιο δράση του προγράμματος Στοκχόλμης. Ώστε να γίνουν πραγματικότητα οι προβλέψει αυτέ, θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο δίδει συγκεκριμένε ημερομηνίε για τις νομοθετικού χαρακτήρα και μη νομοθετικού χαρακτήρα προτάσει που προβλέπονται στο διάστημα 2010-2014. Με αυτό το στόχο θα εργαστούμε επί τη βάση του προσχεδίου της Κομισιόν και είμαστε σε επαφή βέβαια με τις υπηρεσίες της Κομισιόν για το στόχο αυτό και προφανώς θα λάβουμε υπόψη και τις απόψεις των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν το σημαντικό εγχείρημα για όλους είναι να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα εδρεωμένο έγγραφο το οποίο μας οδηγεί σε ρήτρε οι οποίες θα είναι και εφικτές και φιλόδοξες σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Δεύτερον, Θέλουμε να βελτιώσουμε την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσω της ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Σύμβαση της Ρώμης του 1950, όπως αναφέρει το άρθρο 6 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Θέλουμε να γίνει το ταχύτερο δυνατόν αυτή η απαραίτητη νομική, σε νομικό επίπεδο προσχώρησης και περιμένουμε να υπάρξει η δυνατότητα ε, εντολής διαπραγμάτευσης για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Για να προωθήσουμε αυτή τη διαδικασία έχουμε προβλέψει να γίνει ένα σεμινάριο στις 2 και 3 Φεβρουαρίου με παρουσία εκπροσώπων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Συμβούλιο της Ευρώπης, κάτι το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας για ένα θέμα το οποίο έχει και κάποια τεχνική πολυπλοκότητα, όπως γνωρίζετε και εσείς ήδη πολύ καλά. Θα προωθήσουμε επίσης τα εργαλεία τα οποία θα διευκολύνουν την επέκταση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης, ιδιαίτερα στον τομέα της δικαστικής ποινική ε, συνεργασίας. Ένα από τα κύρια στοιχεία της Προεδρίας μας, μαζί με το πρόγραμμα της Στοχόλμης, είναι το να εστιάσουμε την προσοχή μας στην νομική και δικαστική συνεργασία σε σχέση με τα θύματα εγκλημάτων. Θύματα τα οποία πολλές φορές και αδίκως λησμονούνται και των οποίων θα πρέπει να βελτιωθεί η προστασία τους και η αρρωγή που δίνεται σε αυτά τα θύματα. Στην Ευρώπη συνεργαζόμαστε στο ποινικό επίπεδο πάντα από την οπτική γωνία του ενόχου, του, εγκλημα... του Η εναρμόνιση και η συνεργασία και η αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων, αλλά πρέπει συγχρόνως να θέσουμε στο κέντρο αυτής της διαδικασίας και τα θύματα. Κάναμε μόλις στη Μαδρίτη ένα σεμινάριο για τα θέματα αυτά. Εκεί συζητήσαμε επίσης ως μέλη του Συμβουλίου τα ζητήματα αυτά στην πόλη του Τολέδου. Με τον τρόπο αυτό θελήσαμε να προωθήσουμε την παρουσίαση από την Κομισιόν ενός συνολικού νομοθετήματος για τα θύματα των αδικημάτων που ενισχύει το νομικό τους καθεστώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πάνω απ' όλα που βελτιώνει τους μηχανισμούς αποζημίωσης προς τα θύματα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αν σκεφτόμαστε περισσότερο την κατάσταση των θυμάτων και βασιζόμενοι στην πρωτοβουλία που μπορεί να αναπτύξουν τα κράτη-μέλη βάσει της συνθήκης, εμείς με την υποστήριξη άλλων 11 κρατών μελών έχουμε διατυπώσει μια πρόταση <clears throat> ώστε να διευρύνουμε σε όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από μια αρχή εθνική και που έχουν να κάνουν με την προστασία των θυμάτων. Μέσω της ευρωπαϊκής του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Προστασία, θέλουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των θυμάτων σε όλο το ευρωπαϊκό έδαφο και ιδίω να ανταποκριθούμε στην όλο και μεγαλύτερη προσδοκία των θυμάτων ε, οικογενειακής βίας ή ε, κακοποίησης λογοφύλου. <clears throat> Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην αμοιβαία αναγνώριση για να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι αποτελεσματικά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για την προστασία ενός θύματος που θεωρεί ότι βρίσκεται εν απειλή και επέκεινα του, του εδάφους του κράτους μέλους το οποίο διαμένει. Μας φαίνεται λοιπόν ότι αυτό είναι απαραίτητο να, προχω... προωθηθεί γιατί συνδέεται στενά με την έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και φυσικά προσβλέπω και στην υποστήριξη της Επιτροπής σας. Επίσης <clears throat> υποστηρίζουμε ότι πρέπει να προωθηθεί περαιτέρω η αρχή της ε, αμοιβαία αναγνώρισης σε ό,τι αφορά την παροχή αποδεικτικών στοιχείων στις ποινικέ διαδικασίες επί τη βάση μιας, ενός, μιας ευρωπαϊκής τάξης σε ό,τι αφορά <clears throat> τις έρευνες για τέτοιες περιπτώσεις. Θέλουμε να υπάρχει μια πιο φιλόδοξη <clears throat> διαδικασία που δεν επιτρέπει την διπλή απαγγελή κατηγορίας για το ίδιο αδίκημα και που επιτρέπει την αναγνώριση των ε, εντολών που δίδονται για ανακρίσεις σε σχέση με τα θέματα αυτά και προβλέπει ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα για να συμπληρωθούν αυτές οι ενέργειες. Θέλουμε επίσης να μεταρρυθμίσουμε το μοντέλο συμφωνίας για τις κοινέ ανακρίσεις και έρευνες για να προσαρμόσουμε αυτή τη διαδικασία στο φως των εμπειριών που έχουμε συλλέξει τα τελευταία χρόνια. Μια τελευταία προτεραιότητα είναι η βελτιστοποίηση της χρήσης των τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας μέσα στην διαχείριση της δικαιοσύνης. Η Ισπανική Προεδρία ελπίζει ότι θα μπορέσει να εγκαινιάσει το, την δικτυακή πύλη της Ευρώπης για τη δικαιοσύνη Κάτι το οποίο θα φέρει πιο κοντά τη δικαιοσύνη στους πολίτες, αλλά θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε και τις διαδικασίες εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού που εργάζεται στα πλαίσια της ε, απόδοσης δικαιοσύνης. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει επίσης κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας, προβλέπει το αξίωμα ενός Ευρωπαίου εισαγγελέα. Αν και αυτό φαίνεται παράδοξο σε πολλούς, Ακόμα συνεχίζεται η συζήτηση για την υλοποίηση του θέματος αυτού, του αξιώματος αυτού και υπάρχουν πολλαπλές απόψεις σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί. Στην Ισπανία το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έχει συμπεριλάβει μια συγκεκριμένη μνήα για το αξίωμα του Ευρωπαίου Εισαγγελέα και υπό την Προεδρία μας προβλέπουμε να υπάρξει μια πρώτη προβληματική, μια πρώτη διαβούλευση σε σχέση με αυτόν τον νέο θεσμό στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης. Εν τέλει, κυρίες και κύριοι, η εξωτερική διάσταση των πολιτικών ασφάλειας και δικαιοσύνης έχει αποκτήσει, χωρίς καμία αμφιβολία, μια ιδιαίτερη σημασία στον παγκοσμιοποιημένο χώρο στον οποίο ζούμε. <clears throat> Στα θέματα της δικαιοσύνης η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να προάγει το κράτος δικαίου και παράλληλα να προαγάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αντιμετωπίσει τη διαφθορά, να υποστηρίξει την σταθερότητα και επίσης να δώσει ασφάλεια δικαίου στα συστήματα των κρατών μελών για να, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθήσει το εμπόριο και τις ανταλλαγές που είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να συνεχίσουμε την, την δικαστική συνεργασία με τρίτες χώρες και πάντα μέσα στα πλαίσια των εξωτερικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανανέωση της διατλαντικής ατζέντα, όπου τα θέματα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών, όπως γνωρίζετε όλοι, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο τα θέματα αυτά. Η νέα κυβέρνηση Ομπάμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και ένα σημείο καμπής, το οποίο πρέπει να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το εξάμεινο προβλέπεται να γίνουν στην Ισπανία υπουργικέ σύνοδοι τον Απρίλιο των Υπουργών Εσωτερικών και μια διάσκεψη κορυφή με τι ΗΠΑ το Μάιο. Ξεκινώντα λοιπόν από την προηγούμενη σύνοδο του Οκτωβρίου με τι ΗΠΑ, ένα κοινό έγγραφο με τι κατευθυντήρε γραμμέ ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών για τα επόμενα χρόνια, πέντε χρόνια, έχει καταρτιστεί. Και υπάρχει και μια διαδικασία κύρωση των συμφωνιών αμοιβαία αρρωγή και εκρώσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης Με στο πλαίσιο αυτό έντονη συνεργασία είναι απαραίτητο να έχουμε την εντολή η οποία θα μας επιτρέψει να ξεκινήσουμε και τις συζητήσεις που θα οδηγήσουν στο να διερευνήσουμε τη δυνατότητα μιας μελλοντική συνολικής συμφωνίας για την ανταλλαγή πληροφοριών για αστυνομικούς σκοπούς πάντα με ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων, όπως λέει το άρθρο 8 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Ξέρουμε ότι είναι ένα πολύπλοκο και λεπτό θέμα, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι είναι απαραίτητο, ότι είναι εφικτό να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς ασφάλειας χωρίς να υποσκάψουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτή η πεποίθηση επίσης είναι και η πεποίθηση των Αμερικανών φίλων μας όπως είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω στη συνάντηση που είχα με τον Γενικό Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κύριο Έρικ Χόλτερ, καθώς και την ε, Τζάνετ Νοπολιτάνο, την Υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας, στη συνάντησή μας στο Τολέδον. Μας απασχολεί επίσης και η κατάσταση του, της συμφωνίας για την παρακολούθηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Δυστυχώς η Ισπανία ξέρει πολύ καλά τι είναι η τρομοκρατία. Γι' αυτό για να μην δείξουμε καμία δυναμία στο μέτωπο αυτό, θα ήταν απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει, να κυρώσει την προσωρινή συμφωνία των 9 μηνών που επιτύχαμε εργαζόμενοι αγκώνα-αγκώνα στο νομοθετικό αυτό επίπεδο το το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και μπορούμε πια να επιλύσουμε τις τελικές διαφορές που υπάρχουν. Ως Προεδρία ελπίζουμε επίσης να έχουμε την άποψη και του Κοινοβουλίου για τις συμφωνίες του, για το PNR με τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, όπως και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες, κάποιες από τις οποίες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι οποίες δεν είχαν ακόμα ε, δεν είχαν συμπληρωθεί οι διαδικασίε όταν ετέθησε εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Επίση, το εξάμεινό μα προβλέπεται να γίνουν σύνοδοι των Υπουργών Εσωτερικής, Εσωτερικών με, με του ομόλογου του τη Ουκρανία και τη Ρωσία. Θεωρούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συνεργασία στο αστικό και ποινικό δίκαιο με τι χώρε αυτέ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, κλείνω. Αυτές είναι οι βασικές κατευθύνσεις της Ισπανικής Προεδρίας έχουμε προετοιμάσει μαζί με το Βέλγιο και την Ουγγαρία ένα πρόγραμμα δράσης μέσα στα πλαίσια βαθέων και ριζικών αλλαγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα τεθούν σε εφαρμογή επιτυχώς οι νέες διαδικασίες και μέθοδοι εργασίας και θέλουμε από την πρώτη μέρα να έχουμε μια υποδειγματική συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν, γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό είναι ο καλύτερος τρόπος να οικοδομήσουμε την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ, λέει ο Πρόεδρος. Και ακριβώς όπως ε, προείπαμε θα αρχίσει τώρα ένας ε, γύρος παρεμβάσεων έρωτα απαντήσεων, δύο λεπτά για την ερώτηση και δύο λεπτά για την κάθε απάντηση. Συντονιστές, πρώτα-πρώτα των πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια πάλι άλλος γύρος απαντήσεων, τόσο ώστε όσο γίνεται περισσότερο βουλευτές να λάβουν το λόγο. Για το Λαϊκό Κόμμα πρώτα πρώτα. Μπουσούτιλ. Yes, thank you, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Υπουργέ και σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Κύριε Υπουργέ, χθε ε, συναντήσαμε δύο συναδέλφους στην Επιτροπή μας και είχαμε μια πλήρη ανταλλαγή απόψεων μαζί τους. Φυσικά ε, το θέμα της συμφωνίας SWIFT ε, επανήλθε πολλές φορές και μας είπαν ότι θα πρέπει να στραφούμε με την κάνη στραμμένη προς εσάς. Περιμένουμε λοιπόν σήμερα να γίνει μια συζήτηση για το θέμα του SWIFT μαζί σας. Για να ξεκινήσω λοιπόν με αυτό το σημείο και είμαι σίγουρος ότι και άλλοι συνάδελφοι θα συζητήσουν και θα μιλήσουν γι' αυτό. Ξέρετε κύριε Υπουργέ ότι η συμφωνία για τη χρηματοδότηση της δημοκρατίας και το πρόγραμμα ανείχνευσή τους μας εστάλει μόνο αυτή τη βδομάδα. Τώρα αναμένεται εμεί να λάβουμε απόφαση. Ξέρετε ότι για τη διαδικασία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν μεταχειριστήκε σωστά, δεν το αντιμετώπισε σωστά το Συμβούλιο. Ε, πήρε μία απόφαση, καταρχάς, την παραμονή της θέσης ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό δεν είναι μία συμπεριφορά που χαροποίησε το Κοινοβούλιο και εν συνεχεία χρειάστηκαν πολλές εβδομάδες για να μας διαβιβαστεί η ίδια η συμφωνία ε, και τελικά μας ήρθε μόνο αυτή τη εβδομάδα. Και τώρα μας ζητούν να συνενέσουμε σε αυτή τη συμφωνία. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, πραγματικά έχουμε απογοητευτεί από τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο μεταχειρίζεται και αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πόλο δε μάλλον που τώρα τέθηκε σε ισχύ και η συνθήκη τη Λισαβόνα. Τώρα, επί τη ουσία, κύριε Υπουργέ, φυσικά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμεί από πλευρά μα. Θα εξετάσουμε πολύ προσεκτικά αυτή τη συμφωνία. Θα προσπαθήσουμε να μα δοθεί συμβουλή για τη συμφωνία αυτή και θα την ελέγξουμε, θα την εξετάσουμε σε σχέση με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υιοθετήθηκε το περασμένο Σεπτέμβριο του 2009 δηλαδή. Ε, ποια είναι η απάντησή σας στα παραπονά μας για τον τρόπο με τον οποίο το Συμβούλιο αντιμετώπισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια είναι η αποψή σας για την ε, συμφωνία αυτή, αν την συγκρίνουμε με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του περασμένου Σεπτεμβρίου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρία Θα απαντήσει ο Υπουργό. Ε, συνεχεία θα σα δώσουμε τον λόγο εσά για την επόμενη ερώτηση. Γιατί είπαμε πρώτα μία ερώτηση, μετά η απάντηση και ούτω καθεξή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Μπουσούτιλ, είναι μεγάλη μου χαρά να σας απαντώ με ό,τι πληροφορίες έχω στις 30, ενδεκατόταν το Συμβουλίο έλαβε την απόφαση, τότε Θεωρήθηκε ότι έχουμε αυτή την προθεσμία, τόσο ώστε να μπορούμε τώρα να έχουμε μια βάση, ένα θεμέλιο για μια τέτοια νομοθεσία, γιατί όπως ξέρετε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να έχουμε μια τέτοια αναδιάρθρωση της επιχείρησης που έχει αυτά τα δεδομένα, ώστε να μπορούμε να λάβουμε κάποιο μέτρο κάποια στιγμή που ταυτόχρονα με τη θέση ισχύ ορισμένων διατάξεων της ε, συνθήκης Λισαβόνα, να μπορούμε να έχουμε αυτό, αλλά ταυτόχρονα να διατηρηθεί και το status quo το οποίο να παρέχει κάποιες εγγυήσεις ούτω ώστε και το Κοινοβούλιο, το οποίο έχει την τελευταία λέξη, να μπορέσει να λάβει την αντίστοιχη απόφαση. Και αυτός είναι ο βασικός λόγος που στις 30 ενδεκάτου είχαμε το τέλος της εντολής για τις διαπραγματεύσεις. Οπότε, από νομικής πλευράς, επιβαλόταν το Συμβούλιο να λάβει μια απόφαση όντως. Κάθε διαδικασία έχει τα δύσκολα σημεία. Κάθε φορά που ξεκινάει μια καινούργια διαδικασία. Οπότε γι' αυτό και εγώ σας ζητώ να με συμπαθάτε για ό,τι τυχόν προβλήματα σας δημιουργήσαμε. Πάντως εμείς από την πρώτη μέρα προσπαθήσαμε να επιταχύνουμε τους σχετικούς μηχανισμούς τόσο ώστε όλοι αυτοί οι, μηχανισμοί να μπορέσουν να είναι προσβάσιμοι σε όλους τους βουλευτές και επίσης κάναμε ό,τι ήταν δυνατό για να μπορούμε να έχουμε κάποιο είδους διμερείς επαφές με Ένωση και ΕΠΑ σύμφωνα με τα όσα επιτάσσουν οι συνθήκες κάνουμε τα δυνατόν, ώστε να μπορέσουμε να ξαναχτενίσουμε ε, αυτό το κομμάτι της προσωρινής συμφωνίας και να μπορέσουμε να το, να το προσαρμόσουμε στο όσο θα επιτάσσονται στο μέλλον, ώστε να μπορούμε να καλύψουμε αυτόν τον δικαστικό χώρο και έτσι να υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτές τις πληροφορίες. Mm-hmm. Λόπες Αγγελάρ. Και τώρα για τους σοσιαλδημοκράτες η κυρία Γκάντσα. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας και πιστεύω ότι η Ισπανική Προεδρία θα χρησιμοποιήσει τη συνθήκη της Λισαβόνας ε, και θα οργανωθεί με τις επερχόμενες προεδρίες, γιατί τώρα η προεδρία οργανώνεται με τις επόμενες δύο. Δημιουργούν έτσι ένα 18 μήνο προγράμματος. Ε, και θα προωθήσει το πρόγραμμά της. Το SWIFT είναι από τα πιο σημαντικά σημεία. Τις τελευταίες μέρες είναι το σημείο το οποίο ήταν περισσότερο από όλα τα άλλα στα χείλη μας. Θέλω να κάνω ακόμα δύο, υπουργές, ε, δύο ερωτήσεις. Ε, κύριε Υπουργέ, αναφέρατε την προστασία των ανηλίκων και το ότι θέλετε να προωθήσετε αυτό το φάκελο. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα παραπάνω. Ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδια της Ισπανικής Προεδρίας ό,τι αφορά την προστασία των θυμάτων ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ε, την προστασία των ανηλίκων ε, και επίσης για την οριζόντια οδηγία την οποία μελετάει το Συμβούλιο εδώ και πολύ καιρό. Θα θέλαμε να μας πείτε κάποια πράγματα. Έχετε κάποιο σχέδιο για να την προωθήσετε αυτή την οριζόντια οδηγία και με τι χρονοδιάγραμμα σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε Γκέντς για τα καλά σας λόγια και όντως θέλουμε να έχουμε τέτοια στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Τώρα όσον αφορά τα όσα συγκεκριμένα ρωτήσατε. Αναμφίβολα είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία θέσατε για του Ευρωπαίου αλλά και για την ε, πολιτική σε σχέση με τη δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά αυτό το δουλεμπόριο. Ήδη έχουμε προχωρήσει αρκετά, έχουν προχωρήσει διαπραγματεύσει σε πολιτικό επίπεδο στο Συμβούλιο και περιμένουμε κάποια πρόταση τη ε, Κομισιόν η οποία ελπίζουμε να φτάσει τον ε, ρήτρο δυνατόν. Ακόμα πρέπει να γίνουν κάποιε μικρέ ρυθμίσει όσον αφορά το, τη βαρύτητα των ε, ποινών που θα θεσπίσουμε όσον αφορά κάποιες ε, συμπεριφορές, κάποια εγκλήματα, για, γιατί στα κράτη-μέλη υπάρχουν ε, βέβαια διαφορετικές ρυθμίσεις στο καθένα, αλλά θα πρέπει να καταφέρουμε να φτάσουμε σε μια τέτοια συμφωνία, ούτως ώστε να έχουμε κάποιο είδους κοινό τόπο και έτσι το νωρίτερο δυνατόν να μας στείλει και η Κομισιόν την πρότασή της και εμείς να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα στο Συμβούλιο. Επίσης, όσον αφορά την παιδική πορνογραφία και την καταπολέμησή της. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μελετάται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, όπως είπα και πριν για το άλλο ζήτημα, περιμένουμε να στείλουν ό,τι κείμενα χρειάζονται και να προχωρήσουμε σε μια, σε μια οδηγία, να εγκριθεί, να θεσπιστούν κάποιες ε, διατάξεις που να έχουν μια καινούργια διάσταση, διότι για πρώτη φορά να συγκεράσουμε την δίωξη του εγκληματία αλλά και την προστασία του θύματος του εγκλήματος. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι θέλουμε να, να προχωρήσουμε και έτσι να, να δούμε τι πολιτική θα ακολουθήσουμε, την ποινική δικαιοσύνη. Η επόμενη πολιτική ομάδα σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την εισαγωγή σας και εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Μπουσουτήλ και να προσθέσω ότι όχι μόνο το Κοινοβούλιο έτυχε άσχημες μεταχείρισης από το Συμβούλιο, αλλά κατ' επέκταση και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Εμείς πάντα ήμασταν υπέρ της συνεργασίας και παίρνουμε σοβαρά υπόψη μας το θέμα αυτό και τώρα αν βρίσκεσαι σε δύσκολη θέση δεν φταίμε εμείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει ορισμένε προϋποθέσεις για την ψηφοφορία που θα λάβει η χώρα ε, σε δύο εβδομάδες για το SWIFT, κυρίως να έχουμε πρόσβαση σε, όλη τη σχετική, σε όλο το σχετικό υλικό και τις πληροφορίες, γιατί θα πρέπει να μπορέσουμε να ελέγξουμε το θέμα του SWIFT ε, και επομένως θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα πληροφοριακά στοιχεία. Ε, νομίζω ότι η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, που είναι αντίθετη με την συμφωνία όπως έχει ολοκληρωθεί και με την νομική βάση, είναι πάρα πολύ σημαντική για τις συζητήσεις μας. Ε, το Συμβούλιο όμως δεν μας έχει επιτρέψει πρόσβαση σε αυτό το έγγραφο. Και για να σας ενημερώσω, έχω προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτό το σημείο και θα ήθελα να σας πω ότι το Συμβούλιο μας, δεν μας έδωσε πρόσβαση στα στοιχεία, αλλά όχι ομόφωνα, κάποιες χώρες ήταν υπέρ. Για το PNR, όταν πάρουμε απαντήσεις ε, στο ψήφισμά μας, το οποίο εθετήθηκε τον Νοέμβριο του 2008, θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε. Επίσης, καλωσόριζω τα λόγια σας για την προετοιμασία της ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ποια είναι η θέση της Ισπανικής Προεδρίας ε, για δύο χώρες που όχι μόνο αρνούνται να εφαρμόσουν την ομολογία του δικαστηρίου του Στρασβούργου, αλλά αμφισβητούν την αρμοδιότητα και την εξουσία του δικαστηρίου του Στρασβούργου τη στιγμή που είμαστε έτοιμοι να ενταχθούμε. Ε, και το θέμα που είναι ακαθόδες ξέρετε ότι είναι ο διαχωρισμός εκκλησίας και κράτους. Ε, γι' αυτό το λόγο ε, διαφωνούν αυτά τα δύο κράτη. Για το SWIFT έχουμε δύο διαστάσεις. Πρώτα-πρώτα η πιο ουσιαστική, αυτό το οποίο εδώ διακυβεύεται. Ασφάλεια, προστασία δεδομένων υπό συνθήκες, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει πρακτική απειλή η τρομοκρατία της χώρας μας και επίσης από την άλλη μεριά έχουμε και κάποιες θεσμικές ε, σχέσεις που πάλι μας τάσουν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να κινηθούμε. Οπότε και εμείς προσπαθήσαμε να ασκήσουμε τι αρμοδιότητέ μα με υπευθυνότητα για τη λήψη των αποφάσεων. Πρώτα-πρώτα είπαμε να υπάρχει μια προσωρινή συμφωνία η οποία να παραταθεί γιατί κάτι προίσχυε και είπαμε ότι θα έχουν κάποιου συμπειρογνώμονε οι οποίοι θα κάτσουν για να τα ζυγίσουν όλα αυτά και να δούμε πόσο πιο αποτελεσματική η καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Ε, Επίση, λοιπόν, επιβαρόταν να ληφθεί μια τέτοια απόφαση ε, μέσα σε κάποιε κοινέ προθεσμίε επί τη βάση του ισχύοντο δικαίου και του σχέδιου δικαίου ό,τι διατάξει είχαμε. Μακάρι να είχαμε και άλλε καλύτερε. Επομένω, αυτό το οποίο θέλαμε είναι με αυτό το ενιάμι να δοθεί αυτή η παράταση, ούτω ώστε να, είναι, να ανασυνάδει ό,τι, ό,τι αποφασιστεί με τη συνήθεια τη Λισαβόνα. Μια που είναι ένα θέμα που τόσο πολύ καίει του Ευρωπαίου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει προστασία των δεδομένων, αλλά είναι και πολύ σημαντική και η ασφάλεια. Και γι' αυτό είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτή η απόφαση, να είναι έγκαιρη, να καλύψει ό,τι να επί τη βάση για τον όσο θέλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό ήταν ο... ήταν η απότερη ότι απολάβαμε αυτή την απόφαση. Άρα είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια συνεργασία για την κατονίση της τρομοκρατίας να είναι αποτελεσματική και ούτω ώστε να κάνουμε αυτή την παράταση για να μην θεωρηθεί ότι παρελκύουμε την, τη, τη τακτική μας για την κατονίση της τρομοκρατίας Γιατί ξέρουμε ότι μια τέτοια απόφαση δεν θα έχει ούτε ρισκό χαρακτήρα, ούτε είναι δυνατόν ποτέ να ληφθεί εγκρυπτό και απαραίτητο, χωρί να ξέρει το κοινοβούλιο τι γίνεται. Και είπαμε επομένω ότι έχουμε αυτό το εννιάμινο. Σε αυτό το εννιάμινο μπορούμε όλοι μαζί να κάτσουμε και να προβληματιστούμε. Όχι μόνο για το SWIFT, γιατί πάλι θα, δεν θα πειράζει να υπάρχει κάποιο γενικότερη εντολή τη Κομισιόν και να κάτσουμε να, να διαπραγματευτούμε τι θα γίνει για όλα τα αστυνομικά θέματα για τη ΣΥΠΑ. Και έτσι να έχουμε μία, μία άποψη, μία έποψη όλου του, του τοπίου και να ξέρουμε τι γίνεται, πώς θα συγκεράσουμε την προστασία των δεδομένων και ταυτόχρονα και την ασφάλεια. Οπότε αυτό εξηγεί το γιατί η Επιτροπή ο πλευρά της έλαβε την απόφαση που έλαβε. Βέβαια, επειδή ακριβώς πέρασαν μια δικασία στην άλλη, υπήρχαν αυτά τα τα, τα προβληματάκια σε σχέση με το Κοινοβούλιο. Όμω εμείς επαναλαμβάνω προχωρήσαμε προ μια λύση ξέροντα ότι αυτό ε, θα είχε μεταβατικό χαρακτήρα και ότι εν πάση περιπτώσει την τελευταία λέξη θα την είχε το Κοινοβούλιο σα. Συμπληρωματική ερώτηση. Έκανα και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Θα έχουμε πρόσβαση στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Ε, ναι ή όχι. Είναι απλή ερώτηση. Existen, existen una serie de normas que Υπάρχει μια σειρά κανόνων που ρυθμίζουν αυτή τη διαδικασία και ό,τι απόφαση ελήφθη, ελήφθη από τη βάση του κοινωτικού δικαίου, όπως και η τελευταία απόφαση του Πρόεδρου του Συμβουλίου που έστελε αυτήν την επιστολή για τη συνδίκη της Βιέννης κάθε απόφαση που ελήφθη έγινε επί τη βάση αυτών των νομικών βάσεων που θεωρείται ότι ισχύουν. Πράσινη. Ρωμεύω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξεκινήσω με το να σας συγχαρώ κύριε <clears throat> Υπουργέ και έχω να θέσω τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Καταρχήν σε σχέση με την ε, το θέμα της προστασίας των πολιτών. Ποιε είναι οι χώρε οι οποίε έχουν προβλήματα, στι οποίε αναφερθήκατε, για τι οποίε εμεί θα πρέπει να αναφερθούμε τι επόμενε μέρε. Δεύτερο ερώτημα. Συγγνώμη, αλλά το SWIFT παραμένει πρόβλημα. Συζητήσαμε ήδη το διαδικαστικό τμήμα και εγώ υποστηρίζω τα παράπονα που έχουν διατυπώσει ήδη. Για το θέμα της ουσίας, ε, επανέρχομαι στο ερώτημα της κυρίας Ιντφελτ έχετε απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να ζητήσετε τη γνώμη του σε σχέση με το περιεχόμενο αυτού του μέτρου, γιατί παραμένουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα, γιατί είναι μια απόφαση που αφορά τα δεδομένα που πηγαίνουν από την Ευρώπη στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να υπάρχει αντιστάθμισμα από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας μπορεί να υπάρχει μια σύγκρουση. Επομένως, θα ήθελα να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Τρίτο ερώτημα έχει να κάνει <clears throat> με τα άτομα που είναι κρατούμενοι και έρχονται από το Γουαντάναμο στην Ευρώπη. Η Ισπανία και άλλες χώρες όπως ξέρετε έχουν υποδεχθεί αυτά τα άτομα. Κάποια από αυτά τα άτομα υπάρχουν κάποια προβλήματα νομικά που συνάπτονται από αυτά. Συζητήσαμε το πρόβλημα, τα προβλήματα αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις τελευταίες μέρες. Θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση του θέματος αυτού, ποια είναι η διαδικασία που θα γίνει και αν υπάρχει δυνατότητα υποδοχής και άλλων κρατουμένων από το Γουαντάναμο, ο κύριος Υπουργό. Σε σχέση με το πρώτο ερώτημα που διατυπώσατε, το ευρωπαϊκό ένταλμα, η ευρωπαϊκή τάξη προστασίας μάλλον, είναι ένας μηχανισμός αμοιβαίας αναγνώρισης. Ο στόχος είναι να υπάρχει η προστασία των θυμάτων με έναν τρόπο ενιαίο. Γιατί μέχρι τώρα πήκυλε αυτή η προστασία σε σχέση με την εθνική νομοθεσία. Υπήρχαν χώρες όπου υπήρχε μια πολιτική ε, αρχή, ε, μάλλον μια, ένας ε, δικαστής του αστικού δικαίου που προστάτευε τα θύματα οικογενειακής βίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν του ποινικού δικαίου, σε άλλες περιπτώσεις ακόμα και διοικητικού δικαίου αρχές. Είναι απαραίτητο λοιπόν με την αρχή αυτή τη αμοιβαία αναγνώριση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετωπίσαμε <clears throat> για το πλαίσιο αυτό προστασία. Αλλά έχουμε την πλήρη υποστήριξη 12 κρατών μελών και νομίζουμε ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με αποφασιστικό τρόπο σε ένα εργαλείο το οποίο θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για του Ευρωπαίου πολίτε και δεν αφορά μονάχα την τρομοκρατία αλλά αφορά την ε, βία λόγω φύλου και την οικογενειακή βία, θέματα που είναι πολύ σημαντικά για τους Ευρωπαίους πολίτες. <clears throat> Τώρα, για το αν υπήρξε ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με το SWIFT. Πρέπει να σας πω ότι ο χρόνος ανάλυσης, διερεύνησης και προβληματισμού πρέπει να ξεκινήσει τώρα και πρέπει να ξεκινήσει από το ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μέχρι στιγμής το μόνο το οποίο έχει γίνει είναι να πάρουμε μια προσωρινή απόφαση με περιορισμένη χρονική ισχύ, η οποία παρατείνει ένα σύστημα το οποίο υπήρχε στο παρελθόν, συν κάποιες διαδικαστικές εγγύησεις, με στόχο το να μην υπάρξει μία απότομη τομή, μία ασυνέχεια στους μηχανισμούς ασφαλείας, αλλά γνωρίζουμε ότι είναι απαραίτητο να δούμε ποιες θα είναι οι αξιολογήσεις από την πλευρά των νομικών εμπειρογνωμόνων και όχι μονάχα των αστυνομικών εμπειρογνωμόνων, για την αποτελεσματικότητα και την αναλογικότητα του μέτρου αυτού για τα μέτρα ελέγχου τα οποία θα εφαρμοστούν και υπάρχει αυτός ο χρόνος των 9 μηνών για να αναλογιστεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλοι οι εμπλεκόμενοι για την ορθολογικότητα της απόφασης η οποία θα πρέπει να ληφθεί για το μέλλον σε ό,τι αφορά το SWIFT. Τέλος, σε ό,τι αφορά τους κρατούμενους στο Γουαντάναμο, Μπορώ να σας πω πολύ απλά ότι πέραν της συμφωνίας μερικών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υποδεχθούν κάποιους από τους κρατούμενους αυτούς, το θέμα αυτό αντιπο, αντιπετωπίστηκε πάντα στο Συμβούλιο Δικαστικών και Εσωτερικών από τους Υπουργούς Εσωτερικών. Επομένως, εγώ δεν έχω στοιχεία για το ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα ενσωματωθούν μέσα στο ισπανικό νομικό <clears throat> πλαίσιο ή στο ευρωπαϊκό. Η κυρία Βεζάτε βεζατη απο την ΚΟΕ. Κανονικά δεν είμαι εγώ η συντονίστρια, αλλά αντικαθιστώ τον απόντα συντονιστή της ε, ομάδας μου. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θα επανέρχω, στο θέμα της συμφωνίας SWIFT. Ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι όπως και η προηγούμενη α, Σουηδική Προεδρία, υπεκφεύγεται και δεν απαντάτε. Δεν μπορείτε να μας λέτε το δικαίωμα στην ασφάλεια πριν τα ανέβει σε, σχέση με το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Εδώ και πάνω από τρεις μήνες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επαναλαμβάνει τα ίδια ερωτήματα. Εδώ και τρεις μήνες. εδώ έρχονται διάφοροι υπουργοί τη ε, Σουηδικής προεδρία και συνεχεία τη Ισπανική Προεδρία και μα μιλούν για προβλήματα χρονοδιαγράμματος, προθεσμιών κτλ. Αυτό είναι απαράδεκτο. Την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο μα μίλησαν για προβλήματα μετάφραση. Δύο ε, μήνες για να μεταφράσουν μία συμφωνία. Ποιον, κοροϊδεύεται, ποιο κοροϊδεύει ποιον. Ε, πρόκειται για ένα πρώτο πείραμα ε, για την εφαρμογή της συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν μπορείτε να αντιμετωπίζετε το Κοινοβούλιο με αυτόν τον τρόπο. Είναι απαράδεκτο. Είμαστε όλοι πεπισμένοι και όλοι ακούσαμε τον, την Επίτροπο κυρία Ρέντινγκ και την κυρία Μάλστρομ να μας λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει διαφορά μεταχείρισης και ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον, με τον ίδιο τρόπο το θέμα της ασφάλειας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ ε, και εμείς λέμε από πλευρά Κοινοβουλίου εντάξει ε, με το θέμα της ασφάλειας. Ε, συμφωνούμε. Αλλά τι γίνεται με τα προσωπικά δεδομένα. Το Κοινοβούλιο έχει λάβει ένα ψήφισμα το οποίο έχει αγνοηθεί. Κανένα από τα στοιχεία του ψηφίσματος δεν έχουν ληφθεί υπόψη μέσα αυτού του τρει μήνες που έχουν παρέλθει. Είμαστε ακόμα στο ίδιο σημείο, στην ίδια απόφαση μας. Μιλάτε συνέχεια για το χρονοδιάγραμμα. Θα, θα σας θέσω και εγώ μία συγκεκριμένη ερώτηση. Μπορείτε να μας δώσετε μία συγκεκριμένη νομική απάντηση που να εξηγεί γιατί αυτό το χρονοδιάγραμμα είναι έτσι και στις 31, 30 μάλλον Νοεμβρίου θα έπρεπε να πει η ομιλήτρια ε, να πάρει α, απόφαση το Συμβούλιο δεν και καλά εκείνη τη μέρα και να μην περιμένει μια μέρα μετά την 1η Δεκεμβρίου. Είναι λίγο περίεργο, έτσι δεν είναι. Muchas Ευχαριστώ κυρία Βεζιάτ <clears throat> για τις ε, παρατηρήσεις σας. Ο πρώτος που ενδιαφέρεται για να εξασφαλίσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εφαρμογή του άρθρου 8 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, πιστέψτε με, είμαι εγώ. Αλλά για να μπορέσουμε να προασπίσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα, και συγχρόνως να μην θίξουμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, θα πρέπει να εργαστούμε αναζητώντας κοινέ εναλλακτικέ λύσεις. Και αυτό είναι το χρονικό διάστημα που έχουμε τώρα ανοιχτό ενώπιόν μας. Όχι μόνο για το SWIFT, αλλά γενικά για την προστασία των ε, προσωπικών στοιχείων και την ασφάλεια γενικά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Και το PNR και όποια, οποιαδήποτε μορφή ανταλλαγής δεδομένων. Πρέπει να φέρουμε λοιπόν αντιμέτωπα δύο πράγματα και εδώ συμφωνώ μαζί σας. Αναλογικότητα και αποτελεσματικότητα του μέτρου αυτού, διότι άπτεται του θεμελιώδους αυτού δικαίωματος που είναι η προστασία των δεδομένων για τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά παράλληλα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε πώς μπορούμε να διατηρήσουμε κοινέ πολιτικές ασφάλειες με συνεργασία ορισμένων τρίτων κρατών όπως είναι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική. Αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Οι αποφάσει οι οποίε ελήφθησαν είχαν σαν στόχο να μπορέσουμε να καταλήξουμε χωρί να αθίξουμε το πλαίσιο το οποίο ήδη υπάρχει σε μια νέα εναλλακτική λύση. Πρέπει μαζί να δημιουργήσουμε μια νέα αναλλακτική λύση και στις 30 Νοεμβρίου δεν υπήρχε από ό,τι γνωρίζω εγώ κάποια εναλλακτική λύση η οποία να εξασφαλίζει τη σωστή ισορροπία μεταξύ ελευθερίας και προστασίας δεδομένων αφενός και ασφάλειας. Και τα δύο στοιχεία είναι εξίσου σημαντικά. Το πρώτο στοιχείο, η προστασία, είναι θεμελιώδης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να απαρνηθούμε την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό έχουμε ένα πλαίσιο εννέα μηνών χωρί καμία καινοτομία, απλώ παράταση του προηγουμένου καθεστώτο και έχουμε τώρα μια θαυμάσια ευκαιρία να σκεφτούμε και να αναλογιστούμε για τις πάρα πολύ δικαιολογημένες και τεκμηριωμένες αντιρρήσεις της Επιτροπής σας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος των συντηρητικών και αναθεωρητών και θα προχωρήσουμε σε ένα δεύτερο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Ζητώ από αυτούς οι οποίοι θα λάβουν το λόγο να παραμείνουν μέσα σε περιορισμένο χρόνο για να μπορέσουμε να έχουμε ως δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ζήτησαν το λόγο. Σας παρακαλώ και πάλι οι ερωτήσεις σας να περιοριστούν σε ένα λεπτό. Θα γίνουν η μία μετά την άλλη. Θα καταγράψει <clears throat> ο κύριος υπουργό αυτά τα οποία θα πείτε και στη συνέχεια θα κάνει μια τελική παρέμβαση απαντώντας ομαδών. Ο κύριος Βος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. έχετε να αντιμετωπίσετε ένα δύσκολο κληροδότημα σε ό,τι αφορά τα θέματα του SWIFT. Και είναι η, η δεύτερη φορά που πρέπει να αντιμετωπίσετε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το θέμα αυτό. Κατανοώ ότι είναι σημαντικό για το δυτικό κόσμο να υπάρξει μια τέτοια συμφωνία, αλλά γιατί τότε με τόσο ε, τεχνικό τρόπο έχουν λειτουργήσει οι διαδικασίες σε διαθεσμικό επίπεδο. Μιλάτε για μια συνολική συμφωνία. Τότε, αν δεν μπορείτε να έχετε τη συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με ποιο τρόπο θα προωθήσετε μια παγκόσμια συμφωνία. ιδίω σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο αυτής της συμφωνίας. Υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές σε ό,τι αφορά τα πρότυπα και σε ό,τι αφορά και τη νομική κουλτούρα στις διάφορες χώρες του κόσμου. Ίσως είναι απλώς μια θεωρητική ιδέα η συνολική, η παγκόσμια αυτή η συμφωνία που αναφέρατε. Ίσως θέλετε να εξηγήσετε τι ακριβώς εννοούσατε. Ο κύριος Ρομέρο, η κυρία Ρομέρο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα από τα κομβικά θέματα εδώ ήταν ακριβώς η πρόσφατη αυτή διαδικασία όπου ενεπλάκει το Κοινοβούλιο για τα θέματα αυτά. Τώρα βρισκόμαστε στα πλαίσια της ε, συνθήκης της Λισαβόνας και επομένως στα θέματα που ήταν προηγουμένως του τρίτου πυλώνα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Έχουμε δει μια φιλόδοξη θέση από εσά για τα θέματα της αμοιβαίας αναγνώρισης για τις αποφάσεις και τα θέματα προστασίας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρξει αυτό το ξεμπλοκάσμα της κατάστασης με κοινέ αναγνωρίσεις αμοιβέ. Το θέμα είναι όμως με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να δώσετε μια λύση για την προστασία των δεδομένων και την εξισορρόπηση των δικαιωμάτων αυτών με την ασφάλεια. Ποια είναι τα εργαλεία τα οποία θα θέσετε σε λειτουργία ώστε αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε άσχημα να καταλήξει καλά. Ευχαριστώ. Η κυρία Λουτφόρδ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία ερώτηση καταρχήν για το αν ο Υπουργό θα κοιτάξει το θέμα του Ευρωπαϊκού Εντάλματο Σύλληψη. Μιλάει για τα δικονομικά δικαιώματα και το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνία. Ε, νομίζω ότι γίνεται κατάχρηση από κάποια κράτη-μέλη στην εφαρμογή του του Ευρωπαϊκού Εντάλματο ε, Σύλληψη. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται έτσι. Ε, ο κόσμος τελικά ε, μένει στη φυλακή περισσότερο χρόνο, δεν του δίνονται χωρίς να μπορεί να έχει δικαίωμα σε εγγύηση. Έπειτα, για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, θα τους πείτε ότι υπάρχουν κόσμος που κρατούν επαόριστον χωρίς δίκη κτλ. ή θα πρέπει να τους κατηγορήσει ή να τους απελευθερώσει αυτούς κάποιους ανθρώπους γιατί είναι θέμα ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και θα πρέπει να τεθεί αυτό σε αυτό το πλαίσιο. Ο κύριος Ζαπατέρο ε, μας μίλησε την περασμένη εβδομάδα για το SWIFT. Λέει ότι η προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας θα ολοκληρωθεί εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το απορρίψει. Από την άλλη όμως μας λέει ότι νομικά είναι αδύνατο να σταματήσουμε την προσωρινή εφαρμογή. Είναι λίγο δικολαβίστικη αυτή η απάντηση είναι αντιφατική. Ε, μία προσωρινή εφαρμογή μπορεί να ανασταλεί, ναι ή όχι. Για το δεύτερο γύρο, έχεις απόψη, πρέπει να σας πω ότι ο σηκωσνοχικός αν έχει κλείσει τώρα η λίστα των αγορητών, κύριε Μπόζο, έχετε ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λέει ο κύριος Μπρόντς. Με σπέτει για την ενδυνάμωση των θεμελιωδών γεωμάτων, κύριε Υπουργέ. Έχουμε εδώ πέρα δύο συγκεκριμένα έγγραφα. Πρώτα όλα το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αλλά και τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Στην ε, ΑΦΚΟ, την επιτροπή μα την ε, Δευτέρα, ε, για αυτή την αυτοεξαίρεση των τριών χωρών έγινε κουβέντα ε, σε σχέση με τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Επίση, ελέγχθη στη συνεδρίαση τη ΑΦΚΟ ότι κατόπιν του ότι προσυπέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Σύμβαση των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ε, αυτές οι χώρες είπαν ότι θέλουν, αυτές που έχουν αυτό αυτοεξαιρεθεί, θέλουν στο δικαστήριο του Στασβούργου να, να, να, να αυτούς που ε, αυτό αυτοεξαιρέθηκαν να σταματήσουν την, το καθεστώς της αυτοεξαίρεσης μέσω του δικαστήριου. Ελπίζω δεν είναι πάρα πολύ μπερδεμένη η ερώτηση. Και τώρα η κυρία Κίνκα Γκάλ, θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα κύριε Υπουργέ να σου πω άλλο μια ερώτηση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, γιατί με μεγάλη μου χαρά διαπιστώνω ότι υπήρξε πάρα πολύ καλή συνεργασία όσον αφορά την εκπόνηση αυτού του προγράμματος ε, από την Τρόικα, Βελγική, Ουγγρική, Ισπανική Προεδρία. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δουλειά και έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια βήματα πρόοδο όσον αφορά την υλοποίηση της χάρτας των δικαιωμάτων. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε επίσης να προστατεύσουμε τις εθνικές μειονότητες. Έχω συμπορώ την και συγκεκριμένη ερώτηση. Σύντομα γνωρίζουμε ότι πρόκειται να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις, οι συνοήσεις των ειδικών όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εσείς για αυτή την ε, σύμβαση τι μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστώ πρώτα. Υπουργέ. Μας είπατε ότι θα θέλετε κάτι να κάνετε όσον αφορά το δουλεμπόριο θα πρέπει να έχουμε κάποια μέτρα που να προσκοπούν στην πρόληψη. Για πέστε μας, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορεί να κάνει η Προεδρία και έτσι να έχουμε πραγματική πρόληψη. Μπορείτε να κάνετε κάτι ούτως ώστε τα, και στα κράτη-μέλη να υπάρχει λιγότερη ζήτηση από για, για τέτοιου είδου καταστάσεις. Ε, είχαμε κάνει και εμεί κάτι ω Σουηδική Προεδρία, αλλά τελικά δεν καταφέρουμε στο Συμβούλιο. Άρα η Ισπανική Προεδρία θα μπορέσει να καταφέρει κάτι. Προεδρο. Άλμπεχτ. Ευχαριστώ πολύ. Μια παρατήρηση για το SWIFT η οποία συνδέεται με μια ερώτηση. Αν έχω καταλάβει καλά, όταν τα δεδομένα του SWIFT, τα δεδομένα μάλλον δεν θα περνούν στις Ηνωμένε Πολιτείε από την πρώτη, αν δεν περνούσαν από την πρώτη Ιανουαρίου 2010 θα είχαμε ένα νομικό κενό, ένα κενό. Και εγώ θεωρώ ότι θα ήταν δυνατό να καθυστερήσουμε ακόμα περισσότερο την διαδικασία αυτή μέχρι ότου να έχουμε μια απόφαση του Κοινοβουλίου. Δεν, έχουμε, αν, δεν έχετε αναγνωρίσει ακόμα τη σημασία του θέματος αυτού. Δεν υπάρχει κανένα κοινοβούλιο στην Ευρώπη το οποίο έχει εγκρίνει μια τέτοια παρέμβαση στα πολιτικά δικαιώματα. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πολύ σημαντικές συνταγματικές επιπτώσεις. Στην Γερμανία είναι σαφές ότι οποιαδήποτε παραβίαση τέτοιων πολιτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνει χωρίς νομοθεσία από την Γερμανική Βουλή. Επομένως, γι' αυτό εμείς απορρίπτουμε αυτή τη διαδικασία που έχετε αναφέρει. Κύριος Γιακολίνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτά που είπατε για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη, για αυτή την ε, διαδικτυακή πύλη ε, για τα θέματα δικαίου θα ήταν πραγματικά εξυγχρονισμός ε, για τη δικαιοσύνη. Επίσης, ε, πολλές φορές μιλήσατε για το θέμα της συνεργασίας. Συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ατζέντα προβλέπει μια πολύ σημαντική, μια πολύ σημαντική ημερομηνία 10 και 11 Αγκριτζέντο, που είναι και η πόλη μου. Ε, ίσως επειδή η Μεσόγειος είναι πιο κεντρική σημασία από αυτό που αναγνωρίζουμε. Πιστεύετε ότι θα είναι μια καλή χρονική στιγμή αυτή για να καθορίσουμε μια στρατηγική που αφορά και τις επιμέρους ε, διμερείς συμφωνίες με τις τρεις χώρες, αλλά και παράλληλα ε, μιλάει για το προφίλ των μεταναστών. Ε, μιλάει για τους μετανάστες σαν πλούτο και πηγή και θα αναγνωρίσει τη σημασία τους ε, στην ε, ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο Ακτζέντο. Κυρία Μπορσελίνο, ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα κύριε Υπουργέ να σας επιστήσω την προσοχή στο θέμα του οργανωμένου εγκλήματος, ε, μαφιόζικου στυλ, που είναι πολύ πιο ιδιάζων από από το γενικό Γενικώ ας πούμε, γενικός πώς οργανωμένο έγκλημα. Και θα ήθελα να μας πει η Ισπανική Προεδρία αν σκοπεύει να δώσει σημασία και να προτείνει ε, μία νομοθεσία που θα αφορά την κατάσχεση των προσόδων της μαφίας. Ε, στην Ιταλία για αυτό το θέμα υπάρχει νόμος για τη χρησιμοποίηση αυτών των προσόδων για κοινωνικούς σκοπούς. Η υποψήφια επίτροπος, η κυρία Μάλστρομ, είχε σταθεί σε αυτό το σημείο. Ε, θα ήθελα να μου πει η Προεδρία τι άποψη έχει για αυτό το σημείο. Επίση, ένα άλλο σημείο είναι οι μάρτυρε στη δικαιοσύνη. Προβλέπετε κάτι στην Ευρώπη για την προστασία των μαρτύρων. Όχι μόνο για την ασφάλειά του, δεν μιλάω μόνο για την ασφάλειά του, αλλά και για την ίδια την ποιότητα ζωή του. Μιλάω δηλαδή με την ευρύτερη έννοια. Ε, προστασία. Ευχαριστώ κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Κάναμε μια συζήτηση τον προηγούμενο μήνα σε σχέση με την ισορροπία των δικαιωμάτων των πολιτών από τη μία πλευρά και την ασφάλεια από την άλλη μεριά. Εγώ έχω δει τα πράγματα να είναι ότι όταν εμείς θέτουμε κριτικά ερωτήματα σε σχέση με την ασφάλεια των πολιτών και με την, τα δικαιώματα των πολιτών όπως κάναμε με το SWIFT μας λένε ότι ή θα συνενέσετε ή θα συνεχιστούν ή τρομοκρατικές επιθέσεις. Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν ευσταθεί. Εσείς θεωρείτε ότι αν εμείς δεν εγκρίνουμε τη συμφωνία SWIFT θα αποδυναμωθεί η κατάσταση ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι στιγμής το Κοινοβούλιο δεν έχει καμία απολύτως απόδειξη για την αποτελεσματικότητα αυτής της συμφωνίας. Οκτώ χρόνια εφαρμόζεται η συμφωνία του SWIFT. Και είπατε και εσείς ότι σας έχουν επιβεβαιώσει οι επιρρογνώμονες ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ρύθμιση του SWIFT. Λέτε όμως στις απαντήσεις σας ότι τώρα πρέπει να ξεκινήσουμε την αξιολόγηση. Αυτή είναι μια αντίφαση. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω ότι χωρίς πραγματική βάση μας ζητάτε να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία. De Jong. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με όλα όσα, όλα όσα υπόθηκαν για το SWIFT. Κύριε Υπουργέ, δεν μας απαντάτε συγκεκριμένα και νομίζω ότι είναι κρίμα κάτι τέτοιο. Θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή μου σε κάτι άλλο. Εδώ στην Ευρώπη ε, λειτουργούμε στη δικαιοσύνη με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, ό,τι αφορά ας πούμε τις ε, αποδείξεις. Αλλά όμως, σε ό,τι αφορά την ε, επιτήρηση, την εποπτεία για την ε, συγκέντρωση αποδείξεων, δεν κάνουμε πολλά πράγματα. Στην ε, Ολλανδία, ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά νομικά προβλήματα για τον τρόπο που συγκεντρώνται οι αποδείξεις. Νομίζω ότι πρέπει να εποπτεύουμε την εξέλιξη του δικαίου. Και θα πρέπει όμως να μην ξεχνάμε και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ιδίως στις ε, δικαστικές ε, διαδικασίες, νομικές διαδικασίες. Στο, Πρόεδρε, ο πρόεδρος Σαρκοζήλιο και ο Μποργέζιο πολύ πρόσφατα μίλησε για την ε, νέα θέση της γαλλικής κυβέρνησης για το σοβαρό το πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης. Διάφορα ευρωπαϊκά κράτη, όχι όλα, αλλά διάφορα, ε, μιλούν για το αδίκημα της λαφρομετανάστευσης. Η Ισπανική Προεδρία, τι πλεύση θα ακολουθήσει. Πιστεύετε ότι, ότι χρειαζόμαστε μία ευρωπαϊκή στρατηγική για να καταπολεμήσουμε τη λαφρομετανάστευση και σε επίπεδο δικαιοσύνης και σε επίπεδο δικαίου. Και τώρα να δώσουμε το λόγο στον Υπουργό Δικαιοσύνη για να απαντήσει όλε αυτέ τι ερωτήσει που υποβλήθηκαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ του βουλευτέ. Θα προσπαθήσω και εγώ να ομαδοποιήσω τις ε, ερωτήσεις που υποβαλλατε Κάποιε Κάποιες αυτε αυτές είναι λογικά, είναι πάρα πολύ κοντά. Πρώτα-πρώτα, οι ερωτήσεις για το SWIFT να ξεκαθαρίσουμε όσο γίνεται περισσότερο τα πράγματα. Δεν έχει αποφασίσει επί τη ουσία το Συμβούλιο. Για οποιαδήποτε τέτοια απόφαση που θα αφορά τις δημόσιες ελευθερίες, την προστασία των δεδομένων, την προσαρμογή με την πολιτική της ασφάλειας, όλα αυτά δεν θα μπορούσε παρά να αφορούν το Κοινοβούλιο. Βρισκόμαστε σε μια φάση αλλαγής, γιατί πάμε από τη μία συνθήκη στην άλλη. Άρα, θέλουμε να παραταθεί η ισχύ του προηγούμενου καθεστώτος, άπαξ και ο που χειρίζεται τα θέματα αυτά, περνάει τώρα από μια φάση αναδιάρθρωσης. Γιατί είπαμε ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να πάρουμε τα στοιχεία τα οποία θέλουμε από τους Αμερικανούς εκτός αν υπάρχει προηγούμενη έγκριση από την κάθε αρχή η οποία συλλέγει τα σχετικά δεδομένα επομένως δεν είναι δυνατόν να ληφθεί τέτοια απόφαση επί της ουσίας ούτε προτιθέμεθα καμία στιγμή να αποκρύψουμε πληροφορίες, να αποφύγουμε να αποφασίσουμε κάτι που σχετίζεται στην τη κάτι το οποίο είναι θέμα του Κοινοβουλίου σας. Όμως υπάρχουν εδώ πέρα τώρα δύο ζητήματα τα οποία από νομικής πλευράς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτα-πρώτα, στις 30 ενδεκάτου σταματά να ισχύει η νομική βάση για την συνέχιση της ισχύω αυτού του συστήματος. Οπότε ε, πάμε για παράταση ισχύω. Δεν πρόκειται για καμία μεταβολή των όσων ίσχυαν μέχρι τώρα. Επίσης, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, εμείς ως Ευρώπη δεν μπορούμε παρά να αποφύγουμε την μονομερή παράταση της ισχύω της συμφωνίας. Το κοινοβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει. Πρόκειται για ένα από τα πολλά θέματα που εσείς θα πρέπει να ενεργήσετε και εγώ, ως Υπουργός Δικαιοσύνης, θέλω όμως να υπάρχει κάποια ρύθμιση όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ασφάλεια. Και άρα θέλω να υπάρχει ουσιαστικό περιεχόμενο ε, όσον αφορά το άρθρο 8 της Συνθήκης για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. για να ακούμε τι λένε οι πυρογνώμονες, να μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες, να μπορούμε να έχουμε μια ουσιαστική εναλλακτική πρόταση για ένα τέτοιο σημαντικό και περίπλοκο θέμα. Αυτό ε, είναι η πρόθεση που βασίζει τις θεσμικές ενέργειες που έχουμε αναλάβει. Όχι, δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό με την ουσία. Παράταση των όσων ίσχυαν. Παράταση με κάποιες επιπλέον εγγύησεις, περιμένοντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει τις, επί των, ουσίας αποφάσεις. Τώρα, όσον αφορά Ναι, πρέπει να σα πω ότι έχουμε συγκροτήσει κάποιε ομάδε εργασία ψηλού επίπεδου, ε, όπου συμμετέχουν Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Τα, τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών θα γνωστοποιηθούν σύντομα και οι σχετικέ εκθέσει επίση. Και γνωρίζουμε ότι είναι θεμητό να, να προβληματίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με την προστασία των δεδομένων που αφορούν του Ευρωπαίου. πάντω. Κάτσαμε και μελετήσαμε τα όσα λένε οι ειδικοί εμπειρογνώμονε. κάτι το οποίο θα πρέπει και εδώ να συζητηθεί. Εδώ είναι ο σωστός χώρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο. Κάτσουμε και να ζυγίσουμε τι λένε αυτές οι εκθέσεις για τα μέτρα ασφάλειας και τη χρησιμότητά τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Επίσης, υπευλήθη κάποια άλλη ερώτηση και αφορούσε το καθεστώς προστασίας στην Ευρώπη. Έγινε κάποια σχετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσφατα, ήταν θετικά τα αποτελέσματα, παρόλα αυτά όμως έχουμε κάποιες υπερβάσεις εξουσίας, έχουμε κάποιες υπερβολές στην εφαρμογή αυτού του μέσου Μπορούμε να πούμε ότι πρόκειται για κάποιο είδου ε, μεμονωμένα περιστατικά μεμονωμένα περιστατικά παρά το ότι στο σύνολο λειτουργεί καλά η υπόθεση αυτή. Σε όλα τα κράτη-μέλη. Άρα, επιδέχεται βελτιώσεις στο καθεστώς αυτό, το Συμβούλιο έχει λάβει υπόψη αυτά τα προβλήματα και τα επεξεργάζεται. Με την ευκαιρία αυτή πρέπει να πούμε πέραν των ερωτήσεων. Το θέμα, το άλλο, το πάρα πολύ σημαντικό που αφορά την ε, αξιολόγηση και τις εγγυήσει που θα πρέπει να υπάρχουν από πλευρά κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα πρέπει να έχει προτεραιότητα. Θα πρέπει να μπορούμε να δώσουμε στους Ευρωπαίου κάποιε εγγύησει. Να υπάρχει κάποια εναρμόνιση, να προωθούμε του κοινού στόχου και πέραν αυτού θα πρέπει οι εθνικές νομοθεσίες και πέραν της ε, εναρμόνισης να συγκλίνουν στο να υπάρχει κράτος δικαίου, στο να ισχύουν οι βασικές αρχές ενός κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Επομένως είναι πάρα πολύ πολύτιμες οι αξιολογήσεις που γίνονται και το κατά πόσο ξέρουμε τι, τι ισχύει στην πραγματικότητα πέραν της νομοθεσίας. Πώς επομένως λειτουργεί το δικαϊκό σύστημα καθημερινά. Όχι μόνο επομένως τι προβλέπεται, αλλά και το πώς εφαρμόζονται αυτά που προβλέπουν οι νόμοι. Αυτό προβληματίζει το Συμβούλιο, το απασχολεί και οπότε και εμείς ως Προεδρία δεν μπορούμε παρά να ασχοληθούμε και εμείς. Τώρα, όσον αφορά αυτό το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και όσον αφορά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σχετική σύμβαση, εδώ πέρα έχουμε διάφορα ζητήματα που έχουν ανακύψει, πιο πολύ χαρακτήρα, τι θα γίνει όσον αφορά την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα, τα κράτη-μέλη μεμονωμένα, τι φόρμουλα θα, θα βρεθεί, τι διαδικασία θα επινοηθεί. Υπάρχουν θέματα επίσης για το ποιο, ποιος έχει την αυθεντική ερμηνεία, ποιο δικαστήριο, ποιο όργανο πώς θα, ποια, ποια νομολογία θα κατησχύσει. Πάντως, έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρώπη το νωρίτερο δυνατόν να προσχωρήσει αυτή τη σύμβαση επί τη βάση των όσων προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Βεβαίως και έχουμε μια σειρά αριτρών με βατικού χαρακτήρα που αφορούν τα κράτη-μέλη, όμως είμαστε πεπισμένοι ότι σε αυτά τα τεχνικά θέματα υπάρχουν λύσεις τεχνικές και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Άλλο θέμα, το ανέφερε η κυρία Γκάλ, για αυτή την προσχώρηση στην σύνθηκη της Ρώμης. Και εμείς θέλουμε το συντομότερο δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει την εντολή τη διαπραγματευτική για να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Γιατί θεωρούμε ότι είναι κάτι θετικό για την Ευρώπη, θετικό για όλους τους Ευρωπαίους. Επίσης, ανεφέρθηκε για το ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες κάτω κατά των δεσμενών διακρίσεων σε κάποια πολύ συγκεκριμένα θέματα. Συγκεκριμένα έχουμε κατά νου το αστικό δίκαιο ισότητα το οποίο θα πρέπει να αφορά υιοθεσία, γάμο, κληρονομιές, όλα αυτά τα, όλους τους παραδεισιακούς θεσμούς, εκεί θα πρέπει να πρετανεύσει αυτή η αρχή της ισότητας. Κάτι αυτό το οποίο θα πρέπει να εμποτίσει, θα πρέπει να διαπεράσει όλη τη σχετική νομοθεσία για αυτά τα θέματα. Α, το άλλο. Το δουλεμπόριο. Πάρα πολύ σημαντικό για μας. Εντατικά ξεργαζόμαστε το σχετικό έγγραφο της Σουηδικής Προεδρίας. Και είπαμε, το συντομότερο δυνατόν η Κομισιόν να κάνει ό,τι χρειάζεται, να απεμπλακεί το θέμα, γιατί ήδη έχει διαμορφωθεί μια ευρεία συνένεση στο Συμβούλιο για την υπόθεση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσει να γίνει πρωτοπόρα η Ευρώπη σε αυτές όλες τις ε, προσπάθειες καταπολέμησης του φαινόμενου αυτού. Έγκλημα πρέπει να καταπολεμηθεί πάρα πολύ. Επίσης, είχαμε κάποιες άλλες ερωτήσεις που αφορούσαν τη μετανάστευση. Είναι θέματα που αφορούν τους αρμόδιους υπουργούς βέβαια στο Συμβούλιο Βεβαίω και η Ισπανία, όπω και όλε οι χώρε τη Ευρώπη, ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα αυτό, για τη συνεργασία, για τον υπάρχει πολιτική ευρωπαϊκή, το πώ θα ενταχθούν αυτοί οι μετανάστε, πώ θα έχουμε αποτελεσματική πολιτική στα σύνορα, πώ θα μπορέσουμε να ρυθμίσουμε έτσι τον ευρωπαϊκό χώρο. Και προσπαθούμε λοιπόν ως Προεδρία να συντονίσουμε ό,τι δράση χρειάζεται, από ό,τι φορείς χρειάζεται, και να μπορέσουμε να δούμε τι νομοθετικό πλαίσιο θα υπάρχει. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο βγήκε. Τι γίνεται με αυτό τον ευρωπαϊκό μεσογειακό χώρο. Τη συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες Μεσογείου, της εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χρειάζεται, είπαμε, πέραν της δικαστικής και ευρύτερη συνεργασία ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Οργανωμένο έγκλημα. Άλλο θέμα που προέκυψε. Γιατί η τρομοκρατία είναι μόνο μία πλευρά του ζητήματος. Γιατί έχουμε το εργαμένο έγκλημα το οποίο έχει πάρα πολλές μορφές, λειτουργεί σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, πάρα πολλές δυνατότητες έχουν στα χέρια τους κατάσχεση προϊόντων εγκλήματος, προστασία μαρτύρων, όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία τα αντιμετωπίζουμε ε, στην ε, Ισπανία και πιο συγκεκριμένα προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει και με το οργανωμένο έγκλημα σε σχέση με τα ναρκωτικά που σε κάποιες χώρες της Ένωσης έχει τρομερές διαστάσεις. Επομένως, θα πρέπει να δούμε πώς θα υπάρξει η προστασία και των θυμάτων σε σχέση με την προστασία των μαρτύρων. Και είπαμε σε και με άλλα κρατημέλη και σε συζήτηση στο Συμβούλιο να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα προωθηθεί αυτή η προστασία των θυμάτων, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να δουλέψει πάνω σε κάποια συγκεκριμένη ε, πρόταση και να γίνει χωριστή επεξεργασία από το θέμα της προστασίας των ε, μαρτύρων, το οποίο θα συνεχίσει να το προωθεί το Συμβούλιο. Τώρα, όσον αφορά αυτή την κατάσταση του προϊόντων εγκλήματος, σας υπενθυμίζω ότι πολύ πρόσφατα πέρασε αυτή η Ευρωπαϊκή Οδηγία για κάποιους ε, αγαθά, αντικείμενα, τα οποία ήταν προϊόντα εγκλήματος και το τι θα γίνουν, πώς θα κατασχεθούν για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Δεν ξέρω που υπάρχει κάτι το οποίο το παρέλειψα. Συμπάθατε με κάτι το, το, το, το ξέχασα, κάτι δεν το απήντησα. Ευχαρίστω να σας πω. Και έτσι καλώ σας ευχαριστώ όλους για τα καλά σας λόγια. Πάρα πολύ χρήσιμες είναι και οι επικρίσεις τις οποίες έχετε διατυπώσει, γιατί γι' αυτό υπάρχει ένα κοινοβούλιο. Όμως, σας επαναλαμβάνω ότι Πρώτη θέμεθα να συνεργαστούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να αναλύσουμε τα θέματα όλα με σας και αφεντήρια πάντοτε έχουμε το ότι η δική σας Ευρωκοινοβουλευτική Επιτροπή και το Κοινοβούλιο γενικότερα πρέπει να έχει όλα αυτά τα θέματα την τελευταία λέξη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ήταν επικνή, πολύ ενδιαφέρουσα, καρποφόρα συζήτηση και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και όλα τα μέλη της Επιτροπής μας που έλαβαν το λόγο. Μπορούμε λοιπόν να κλείσουμε αυτή την συνάντηση ευχόμενοι στον Υπουργό Δικαιοσύνης τύχη και σωστή πορεία, φυσικά και κάθε επιτυχία στην ε, προσπάθεια του να επιτύχει τους στόχους του Έχουμε λοιπόν μια σειρά από σημαντικά θέματα στην μέση διάταξη. Έχουμε τον Γιλ Ντε Κέρκχοβ, τον συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα κατά πολέμηση τρομοκρατίας και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων. Αλλά προηγουμένως θα ήθελα να αποχαιρετήσω τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Σα ευχαριστώ. pour Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να κάνετε παρακαλώ. Καθίστε λοιπόν παρακαλώ. yes. As we Ξεκινάμε και πάλι με την ημέρησια διάταξή μας και προχωράμε στο επόμενο σημείο και σας είχα ανακοινώσει ότι οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων στην χθεσινή συνάντησή τους σε αυτή καθεαυτή την αίθουσα χθε το βράδυ. Αποφασίσανε οι συντονιστές να διορίσουν τους εξής εισηγητές. Την κυρία Χένις Πλάσσαρτ ως εισηγητρία για το θέμα του SWIFT. Η κυρία Ιντ Φέλτ για το PNR, τα δεδομένα των επιβατών έναντι των ΗΠΑ και της Αυστραλίας και η κυρία Ρόμερο Λόπεθ για το καθεστώς προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν καμία αντίρρηση, θεωρείται ότι επικυρώνεται η απόφαση των συντονιστών. Προχωρούμε τώρα στο επόμενο σημείο που αφορά το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας. Κύριε Μπουσούτιλ, αν μου επιτρέψετε κύριε Πρόεδρε, που προχωρήσουμε μοναχα ένα διαδικαστικό σημείο θέλω να θίξω, σε σχέση με το SWIFT. Θα ήθελα να γνωρίσω αν η Επιτροπή μας έχει αναζητήσει μια γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου σε σχέση με την ουσία της συμφωνίας, με το κείμενο της συμφωνίας. Ίσως η συγγήτρια, την οποία εγώ θέλω να συγχαρώ, μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό αλλά προηγουμένως αυτή τη βδομάδα εγώ έθεσα ένα ερώτημα για το αν είχαμε ζητήσει νομική, μια νομική γνωμοδότηση για την ουσία αυτής της συμφωνίας και θα ήθελα να ξέρω αν έχει υπάρξει κάποια πρόοδο σε σχέση με το θέμα αυτό. Κατά πόσο λοιπόν η δική μας Επιτροπή θα αναζητήσει τη γνώμη εμπειρογνωμόνων σε νομικά θέματα προτού καταλήξει σε μια συνεκτική θέση εν καιρό. Καταγράψαμε αυτή την αίτηση, δεν έχει γίνει ακόμα, θα το κάνουμε θα αποστείλουμε μια επιστολή στην νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώντας κατεπηγόντως τη γνωμοδότησή τους και επίσης θα αναφερθούμε και στον επόπτη προστασίας δεδομένων. Η κυρία Πλάσαρτ, μπορούμε να έχουμε μια καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή γιατί νομίζω ότι ο χρόνος τρέχει. Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θα πρέπει να γίνει με τον πιο κατεπήγον δυνατό τρόπο. Προχωρούμε λοιπόν στο επόμενο σημείο, στο σημείο υπαριθμών 11, Ευρωπαϊκό Κάθεστος Προστασίας, <clears throat> Προστασία των Θυμάτων. Όπως τονίσαμε αυτό είναι μια πολιτική προτεραιότητα στα θύματα ποινικών αδικημάτων έχουν το δικαίωμα στην αποκατάσταση των ζημιών και στην τιμωρία του αδικοπρακτούντος Έχουμε λοιπόν εδώ μια παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας και έχουμε ανακοινώσει ήδη ότι θα αλλάξουμε τη σειρά των σημείων αυτών στην ημερήσια διάταξη. Απλώς πρόκειται για μια ανακοίνωση για το σημείο αυτό. Τόνισαν ότι 12 κράτη-μέλη έχουν καταθέσει μια πρωτοβουλία για μια οδηγία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Καθεστώς Προστασίας. Ο στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι να ενεργοποιηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να μην υπάρξει επανάληψη ενός αδικήματος από τον ίδιο δράστη εναντίον του ίδιου θύματος. Γιατί οι στατιστικές τονίζουν ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ συνηθισμένο φαινόμενο. ιδίω στην περίπτωση βίας που έχει να κάνει με το φύλλο, σεξουαλική ε, εκμετάλλευση, λαθρεμπορία ατόμων. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόζεται αυτό σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το καθεστώς αυτοποστασίας και θα δώσω το λόγο για πέντε λεπτά κατά μέγιστο στον κύριο Χωσέ Μολίνος Κόμπος που είναι εκπρόσωπος της Ισπανικής Προεδρίας και στη συνέχεια θα ακούσουμε την άποψη του κύριου Λεβέντ Αλτάν που θα παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κομισιόν μάλλον για αυτή τη συμφωνία. Κύριε Κόμπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλημέρα κύριε και κύριοι. Μικρόφωνο παρακαλώ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάσω το θέμα αυτό του Ευρωπαϊκού Καθεστώτος Προστασίας. Είναι μια πρωτοβουλία, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής σας, 12 κρατών μελών, παρά το γεγονός ότι είναι μια πρωτοβουλία 12 κρατών μελών προς το παρόν. Έχει τύχει συζήτηση και διαβούλευση με την Κομισιόν από την αρχή και τα γεροφάσκια της πρότασης αυτής και η Κομισιόν μας έχει δώσει από την αρχή την πλήρη υποστήριξή της για να μπορέσουμε να διακπαιρεώσουμε αυτή την πρόταση και εξάλλου η Κομισιόν συμμετέχει ενεργά στη συζητήσεις μας και θέλω να την ευχαριστήσω για το γεγονός αυτό. Ελπίζω θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε και με την υποστήριξη της εισηγήτριας, η οποία μόλις διορίστηκε, που ασχολείται με την πρόταση αυτή. Γιατί παρουσιάζεται τώρα αυτή η πρωτοβουλία από την Ισπανία για ένα πολύ απλό λόγο. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νομικό κενό στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δράστης ή ο υποτιθέμενος δράστης ενός ε, αδικήματος όταν αλλάζει, μια, όταν αλλάζει την κατοικία του και βγαίνει από τα όρια του κράτους μέλους δεν καλύπτεται από τα μέτρα απαγόρευσης ή εποπτείας τα οποία το έχουν επιβληθεί στο κράτος μέλος αυτό. Επίσης όταν υπάρχουν ποινές οι οποίες είναι εναλλακτικές της φυλάκισης ή της κράτησης πρέπει να υπάρχει η εποπτειας τα οποια του εχουν επιβληθει στο κρατος μελος αυτο επισης οταν υπαρχουν πίνες οι οποιες ειναι εναλλακτικες της ε, παρακολούθησης του ατόμου αυτού και εκτός του κράτους μέλους. Αλλά όταν πρόκειται για το θύμα το οποίο βγαίνει από το κράτος μέλος όπου υπήρξε το μέτρο ασφαλείας υπέρ του, πάβει να υπάρχει η προστασία του θύματος. Το μέτρο προστασίας λοιπόν παραμένει μέσα στο εθνικό κράτος όπου έχει γίνει η δικαστική απόφαση. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία είναι απαράδεκτη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί παραβιάζει την ελευθερία διακίνησης που είναι μια από τις βασικές από τις τέσσερις βασικές ελευθερίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχει νόημα με την άσκηση μιας τέτοιας ελευθερίας να χάνει το θύμα το δικαίωμα προστασίας. Ενώ το δικαίωμα αυτό προστασίας θα πρέπει να το συνοδεύει όπου και να βρίσκεται μέσα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς στην περίπτωση της βίας λόγω φύλου δεν έχουμε ακόμα αξιόπιστες στρατηγικές για τα θέματα αυτά. Πολλά κράτη-μέλη δεν έχουν καν στατιστικές για τα θέματα αυτά. Τα κράτη-μέλη που έχουν αυτά τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούν τα ίδια κριτήρια και δεν μπορούμε να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία ομού. Υπάρχει η ισπανική πρόταση για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τη βία λόγω φύλου και θεωρούμε ότι θα μπορέσει να υπάρξει εν καιρό ένα σύνολο στατιστικών αξιοπίστων που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Η Ισπανική Προεδρία Έχουμε κάνει μια προσπάθεια να αποκομίσουμε στοιχεία από τα κράτη-μέλη. Μας, είπανε, μας απαντήσανε 18 κράτη-μέλη από τα 27 και μόνο 13 μας δώσανε στοιχεία. Μέσα στα πλαίσια μιας μελέτης αντικτύπου, εμείς <clears throat> κάναμε την μελέτη για το 2008 και φαίνεται ότι το 2008 υπήρχαν 73.000 περιπτώσεις όπου υπήρξαν αποφάσεις προστασίας έχουμε 118.000 τέτοια μέτρα προστασίας το 2009. Αυτά είναι ένα σημαντικό αριθμός για τα μέτρα προστασίας. Αλλά αν δούμε στατιστικές αποφόρεις όπως ε, το WAY, οι γυναίκες κατά της βίας στην Ευρώπη, είναι ανατριχιαστικά τα στοιχεία τα οποία έχουμε αν δείτε την ιστοσελίδα αυτού του φορέα, βλέπει ότι στην ετήσια έκθεσή του για το 2008 για τη βία κατά των γυναικών φαίνεται ότι είναι πάνω από 348.000 περιπτώσεων βίας κατά των γυναικών. Μόνο σε 15 κράτη-μέλη που είναι αυτά στα οποία δραστηριοποιείται αυτή η οργάνωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι αν στην περίπτωση του 1% των θυμάτων αυτού του είδους βίας υπάρχει μετακίνηση, ήδη έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Επομένω, αυτή είναι η αιτιολόγηση τη πρότασή μα. Θεωρούμε ότι με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τη βοήθεια όλων των κρατών μελών, θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε τι απαραίτητε αποφάσει που θα μα επιτρέψουν να επεκτείνουμε την προστασία και στον τομέα αυτό. Έχουμε επικεντρωθεί στην βία λόγω φύλου, παρά το γεγονός αυτό είναι ένα γενικό μέτρο το οποίο θα πρέπει να καλύψει όλα τα μέτρα προστασίας των θυμάτων. αλλά λόγω της ευαισθησίας αυτού του θέματος καταλαβαίνετε ότι σε μεγαλύτερο στο κύριο, κατά κύριο λόγο θα εφαρμόζεται σε περιπτώσεις βίας λόγω φύλου. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Πρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Σόγκαρ. Ένα λεπτό. Να ακούσουμε τη θέση της Κομισιόν για τη θέση της, για την πρωτοβουλία αυτή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και τώρα θα συνεχίσω στα αγγλικά. Ευχαριστώ που μου δείξατε το λόγο, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα, η Κομισιόν υποστηρίζει πλήρως την πρόταση της Ισπανικής Προεδρίας, τους στόχους της, που είναι να προστατευτούν τα θέματα από τη βία λογοφύλου και συμφωνούμε και με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, δηλαδή να επιτευχθούν αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν και δυνατόν το 2010. Η προστασία των δεδομένων είναι ένα θέμα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε δύο νομοθετήματα, ένα για την, το καθεστώς των θυμάτων στις ποινικέ δίκες από το 2001 και μία οδηγία για την αποζημίωση των θυμάτων ε, μέτρο του 2004, νομοθέτημα του 2004. Ε, πρόσφατα αξιολογήθηκαν ε, από την Κομισιόν το 2009 και το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερο και σε αυτά τα μέτωπα. Ο χαρακτήρας προτεραιότητα τη προστασία των δεδομένων επιβεβαιώθηκε επίση και από την κυρία Ρέντινγκ ε, ενώπιόν σα, την υποψήφια επίτροπο στην πρόσφατη ακρόασή τη τον Ιανουάριο. Και επιβεβαιώθηκε ότι η προστασία των δεδομένων είναι προτεραιότητα και για αυτήν και για την Κομισιόν εν Ετοιμαζόμαστε λοιπόν να συνεργαστούμε με την Ισπανική Προεδρία για το θέμα αυτό. Η Κομισιόν ετοιμάζει μία μελέτη που θα οδηγήσει σε μελέτη αντικτύπου για μια μελλοντική πρόταση που θα αποτελέσει ένα είδος πακέτου και που θα συγχωνεύσει την απόφαση με την οδηγία. Κάποια στιγμή στις αρχές του επόμενου έτους θα γίνει αυτό. Αυτά, Πρόεδρε, και ελπίζω να συνεχίσει καλά η Ισπανική Προεδρία. Ήδη υπάρχουν κάποια ψωμένα χέρια. Το θέμα δεν είναι να γίνει συζήτηση για αυτό το θέμα. Η συζήτηση θα γίνει σύντομα. Θα έλεγα να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Έχουμε καθορίσει έναν εισηγητή, την κυρία Ρομέρο Λόπες. Και σε μια επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ θα ακούσουμε την εισηγήτρια και θα ακούσουμε τις προτάσεις της. Θα περάσουμε σε πιο συγκεκριμένα θέματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουμε μία συζήτηση για τα θέματα αυτά ε, που αποτελούν μεγάλη προτεραιότητα της Ισπανικής Προεδρίας. Και τώρα ας περάσουμε στο επόμενο σημείο που είναι το σημείο 9. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην πολιτική καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Με τους αρωτές σώματος ε, θα μιλήσουμε για την πτήση του Detroit. Θέματα πολύ ενδιαφέροντα για όλους μας. Θα ακούσουμε καταρχήν το συντονιστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της ε, τρομοκρατίας, τον κύριο Ζίλντε Κέρκοφ. Και αμέσως μετά θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, τον κύριο Μπουταρέλη. Και με αυτή την ευκαιρία θα γίνει συζήτηση μετά από αυτές τις παρεμβάσεις και θα διατυπώσουν οι βουλευτές ε, τις ερωτήσεις τους προς τους δύο μιλητές. Ε, καλώς ήρθατε κύριε Ντεκέρκοφ. Θα μπω κατευθείαν στο ζουμί γιατί είσαστε, πιέζεστε και το χρόνο. Καταρχάς, θα ήθελα να σας πω ότι η πτήση του Detroit και τα όσα συνέβησαν ήταν πολύ ενδιαφέροντα για πολλούς λόγους. Καταρχάς επιβεβαιώνει κάτι που ξέραμε, ότι η πολιτική αεροπορία είναι και θα παραμείνει στο στόχαστρο των ε, τρομοκρατών. Ε, καθώς και άλλα μέσα μεταφοράς, ε, θαλάσσια και ισοδρομικά. Δεύτερον, τονίζει ότι πέρα από την σημασία της προστασίας των δεδομένων, της συλλογής των δεδομένων και του επιμερισμού αυτών των στοιχείων, θα πρέπει να βελτιώσουμε την ικανότητά μας να, να ενσωματώσουμε, να αφομοιώσουμε θα έλεγα τα δεδομένα που έρχονται από διάφορες πηγές μυστικές πληροφορίες, ε, αστυνομικά δεδομένα, δεδομένα από τη δικαιοσύνη, από τις θεωρήσεις, από ανοιχτέ πηγές, από τον ιδιωτικό τομέα. Άκουσα πολλά για το SWIFT σήμερα και στοιχεία από το PNR, το Μητρό Ονομάτων Επιβατών κτλ. Αν διαβάσατε την ε, έκθεση του Τζον Brennan, του Συμβούλου του Πρόεδρου Ομπάμα, για το τι συνέβη και το τι πήγε στραβά στην πτήση Detroit, το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπόρεσα να συνδυάσω αυτές τις πληροφορίες στην Αμερική. Τρίτον, και ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχητικό παράλληλα, είναι η, η πρόθεση της Αλκάντα, της Αλ... Αλκάντα να κάνει περιφερειακές υποομάδες. Με franchising όμως. για να επιτεθεί εκτός της ε, περιοχής ε, που λειτουργούσε παραδοσιακά. Αυτή είναι μια νέα εξέλιξη. Η προσπάθεια Σομαλών να σκοτώσουν στη Δανία και η πτήση του Ντιτρόιτ επίσης μας κάνει να σκεφτούμε. Ε, και η χρήση νέων προσώπων, όπως του Αμπτούλ Μουταλά, που είχε την ικανότητα να πάρει θεώρηση για το ταξίδι στις ΗΠΑ. Και κάτι άλλο που θα δείτε στην ε, έκθεση που σας έστειλα, και στις τέσσερις μάλλον πέντε προηγούμενες εκθέσεις, η όλο και μεγαλύτερη σημασία ε, που παίρνει το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης. Ο Μουταλά, ο νέος αυτός, ήταν ε, και πλούσιος ε, και μορφωμένος, είχε σπουδάσει στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, ριζοσπαστικοποιήθηκε σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Γιατί? Πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Κάτι άλλο ενδιαφέρον. Επανέρχομαι στα όσα είπαμε στο Τολέδο την περασμένη φορά με την ε, Αμερικανίδα Υπουργό Ναπολιτάνο. Είναι ότι οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται και περισσότερο για το θέμα της ριζοσπαστικοποίηση. Αν δείτε τις πρόσφατες ε, τα πρόσφατα γεγονότα στις Ηνωμένε Πολιτείε, πάρα πολλοί Σομαλοί, Αμερικανοί πολίτες, ε, μπαίνουν στον αγώνα στη Σομαλία. Αυτό θα μπορούσαμε να το κοιτάξουμε ε, στα πλαίσια της συνεργασίας με τους Αμερικανούς. Επίσης, κάτι άλλο που υπάρχει σε όλες τις εκθέσεις μου και εδώ θα πρέπει να κινητοποιηθεί η Ευρώπη περισσότερο, είναι η Εμένη οι άλλα κράτη τα οποία βρίσκονται ας πούμε στην υποσαχάρια ζώνη ε, που είναι σε φάση που δεν τα κατάφεραν ας πούμε και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ασφαλείς ουρανούς για τους τρομοκράτες. Στην κοινή δήλωση που συμφωνήσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Τολέδο, νομίζω ότι μιλάμε για τις περισσότερες απειλές που ανέφερα. Καταρχάς η ασφάλεια της αεροπορίας. Ε, πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα υπήρχε συνένεση είναι ότι δεν αρκούν ο εξοπλισμός και τα μηχανήματα στα αεροδρόμια. Πρέπει να έχουμε μια προσέγγιση διαστρωματική. Συλλογή δεδομένων, καταρχήν, δεδομένα από το Μητρό Ονομάτων των Επιβατών είναι ένα από αυτά. Ε, πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, αστυνομικές πληροφορίες, παραδείγματος χάρη από τα κλαμέ, κλαπέντα και χαμένα αυτοκίνητα, ε, πληροφορίες ε, για το ποιος έχει πάρει η θεώρηση, ποιος, σε ποιον έχει αρνηθεί η θεώρηση κτλ. Και πληροφορίες για την έξοδο των ατόμων. Ακόμη και αν μοιάζουν αμφιλεγόμενα αυτά που λέω, θα πρέπει να συλλέξουμε δεδομένα, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε πρόθεσμα μια συμφωνία με του Αμερικανού για να μπορέσουμε α, να διασταυρώσουμε τις, ε, τους καταλόγους μας για τα επικίνδυνα πρόσωπα. Αλλά αυτό το καταφέρουμε μόνο αν υπάρχει προϋ... αν έχουμε συνάψει νομικά δεσμευτικές ε, συμφωνίες ε, για αυστηρά προστα... Ε, καθεστώτα προστασίας δεδομένων. Υπάρχει συνένεση στα επίπεδα στις ομάδες του Συμβουλίου για αυτά. Υπάρχουν διάφορα προσκόμματα. αλλά όταν έχει μια νέα εντολή η Κομισιόν θα το ξανασυζητήσουμε. Έπειτα, βιομετρικά στα ταξιδιωτικά έγγραφα, ασφαλή έγγραφα, ε, ο τρόπος ε, διαχείρισης ε, της ταυτότητας. Ε, βεβαίως υπάρχει και το θέμα ε, της διαφθοράς σε πολλές χώρες. Αν πιέσουμε σε πολλές χώρες να υπάρξουν τα βιομετρικά στοιχεία στα διαβατήρια, τότε ε, αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της κλεμμένης ταυτότητας. Ξέρω ότι συζητιέται αυτό το θέμα στην, στο Κοινοβούλιο. Ε, προχωρημένη, προηγμένη τεχνολογία στα αεροδρόμια. Θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε έρευνα για την ασφάλεια. Στο πρόγραμμα ε, πλαίσιο Έχουμε 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ για την έρευνα και έχουμε κρατήσει πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ για το 2010 για αυτή την έρευνα. Και το θέμα βεβαίως των εχνευτών σώματος, των σαρωτών σώματος. Είναι σημαντικό το συντομότερο δυνατόν να προχωρήσουμε. Ε, αυτή τη στιγμή πολλά κρατημέλη δοκιμάζουν τα μηχανήματα αυτά. Και διερωτώ με μήπως πρέπει να εναρμανώσουμε ή να πλησιάσουμε τα μέτρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσουμε και τα σημεία που αναφέρατε εσείς στο ψήφισμά σας. Ούτως ώστε αυτή η νέα γενιά των σαρωτών σώματος, που από ό,τι μου είπαν είναι φιλική για την ιδιωτικότητα του, του ατόμου, είναι ασφαλής και θα, ήταν, θα είχε ανοιχνεύσει αυτά που έφερε πάνω του ο Απτούλ Μουταλάχ. Η ασφάλεια λοιπόν ε, στην πολιτική αεροπορία. Θα θυμάστε ότι είχαμε αξιολογήσει τις διευθετήσεις στα 27 κράτη-μέλη για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία και ένα από τα πρώτα πορίσματα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα κέντρο σε κάθε κράτος μέλος και μόνο 12 με 15 κράτη-μέλη έχουν δημιουργήσει αυτό το κέντρο, ένα κέντρο όπου ε, συλλέγουμε πληροφορίε, όλε αυτέ τι διαφορετικέ πληροφορίε από τι αρνητικέ πηγέ, από την, ε, τον τομέα τη δικαιοσύνη, από την αστυνομία κτλ. Είναι μια προσπάθεια, ε, δεν είναι εύκολο να γίνει. Η Ισπανική Προεδρία την περασμένη εβδομάδα στη Μαδρίτη συγκάλεσε μια συνάντηση αυτών των 12 με 15 κρατών μελών που έχουν τέτοια, κράτη, τέτοια κέντρα συγγνώμη, ε, συζήτησαν για το πώς θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο. Οι Αυστραλοί ήταν παρόντες, οι Καναδοί και η NCTC, από τη ΣΥΠΑ ήταν εκεί. Ε, πρέπει να μάθουμε ένας από τον άλλον, θα πρέπει να δούμε και να καταρτήσουμε εμπειρογνώμονες. Ριζοσπαστικοποίηση. Είναι από τις πρώτες προτεραιότητές μου. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Και αν διάβασα την τελευταία μου έκθεση το Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009 θα καταλάβατε πόσο με ενδιαφέρει να επενδύσουμε και θα επενδύσω εγώ προσωπικά σε αυτό το θέμα. Θα επενδύσω εγώ προσωπικά. Ε, ταξίδια. Μια άλλη ανησυχητική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια είναι ότι όλοι και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί φεύγουν από την πατρίδα τους και προσπαθούν να ταξιδέψουν σε προβληματικές περιοχές. Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ιεμένη, Μαυριτανία, Μαλή, για να πάνε σε στρατόπεδα άσκησης. Θα πρέπει να δούμε με τους Αμερικανούς πώς μπορούμε να μάθουμε περισσότερα για το αμό οπεράντι οπεράντη και τις οδούς που χρησιμοποιούν αυτοί οι επίδοξοι τζιχαντιστές. Και τέλος ε, βοήθεια σε τρίτες χώρες. Πριν από 1,5 χρόνο ξεκίνησα μαζί με την Κομισιόν να προσπαθώντας να κινητοποιήσουμε χρήματα κοινοτικά και των κρατών μελών για να αναπτύξουμε την ικανότητα αυτών των κρατών που δεν τα καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της δημοκρατίας. Όχι μόνο... Κοιτάξτε, όχι να δράσουμε χρονιστέρα, να προβλέψουμε την, ε, και να προλάβουμε τη ριζοστοπαστικοποίηση. Συγγνώμη. Ε, φυσικά, σήμερα το απόγευμα θα γίνει μια συνεδρίαση για το πώς θα αντιμετωπίσει η ΕΜΕΝ το πρόβλημα της ε, τρομοκρατίας συλλογή δεδομένων, κατάθεση αστυνομικών και μυστικών υπηρεσιών. Ε, καλά είναι όλα αυτά, αλλά χρειάζεται και πρόληψη. Πρόληψη. Είναι μια χώρα που έχει τεράστια δημογραφική ανάπτυξη. Έχουν χιλιάδες, χιλιάδων νεαρών ανέργων που κάποια στιγμή μπορεί κάλλιστα να ριζοσπαστικοποιηθούν. Ε, είναι πολύ σημαντικό λοιπόν. Και για να μην μακρηγορήσω, Εγώ ως συντονιστής για την κατα... καταπολέμηση της τρομοκρατίας θέλω να δω πολύ γρήγορα τη μελέτη της Κομισιόν για τους αρωτές σώματος, ούτως ώστε το Συμβούλιο και η Κομισιόν να λάβουν θέση μετά από μια ενδελεχή συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να πάρουμε επίσης ε, προτάσεις με βάση το πνεύμα της Λισαβόνας για το PNR. Η διάθεση των Υπουργών στο Τολέδο την ε, περασμένη εβδομάδα των Υπουργών Εσωτερικών ήταν να συνεχιστεί η συζήτηση γι' αυτό και να ξεκινήσουμε το συντομότερο δυνατό τι διαπραγματεύσει για μια συμφωνία με τους Αμερικανούς για την προστασία των δεδομένων. Όπως ανέφερα, με στο πλαίσιο που ανέφερα. Επίσης θα συνεχίσω τη συνεργασία με του Αμερικανού για τα ταξίδια, για την ε, τη στρατολόγηση, τη ριζοσπαστικοποίηση, την ε, σωμάτωση των δεδομένων και τη βοήθεια στις χώρες, τρίτες χώρες, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την προστασία της πολιτικής αεροπορίας. Ε, Έχω καταγράψει μια σειρά από μέλη τα οποία θέλουν να λάβουν το λόγο για να διατυπώσουν ερωτήματα. <clears throat> Θα ήθελα να προτείνω να ξεχωρίσουμε αυτή τη συζήτηση για την αντιτρομοκρατική στρατηγική από την επόμενη συζήτηση που θα γίνει σε σχέση με τον επόπτη προσωπικών δεδομένων. Πρώτος γύρος λοιπόν για τον κύριο Ντεκέρκ Χόβε και στη συνέχεια ακούσουμε τον κύριο Μπουταρέλη από την Κομισιόν και τον κύριο Φάουλ από την Κομισιόν. λοιπόν, Παρακαλώ να είσαστε σύντομοι στις ερωτήσεις σας. Ένα λεπτό, επομένως, ο κάθε ένας ο οποίος θέτει ερώτημα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, διαδικαστικό ερώτημα. Ένα λεπτό είναι μια φάρσα. Τα θέματα αυτά που μας παρουσιάστηκαν είναι η στρατηγική του υπευθύνου για την ε, αντιτρομοκρατική <clears throat> ατζέντα. Ξέρω ότι έχουμε μια ημέρηση διάταξη. Είχαμε μια μακρά συζήτηση για την Ισπανική Προεδρία. Δεν μπορούμε σε ένα λεπτό να εκφραστούμε πλήρω. Ναι, αλλά είναι το τελευταίο σημείο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν τουλάχιστον 20 μέλη, 2 λεπτά. Αυτό θα καλύψει πάνω από μία ώρα. Αν θέλετε να το κάνουμε έτσι, 2 λεπτά, αλλά νομίζω τότε 2 λεπτά. Γιατί αν είναι πάνω από 2 λεπτά την έχουμε βάψει. Το καθήκον μου είναι λοιπόν να προσπαθήσω να κρατήσω την ημερήσια διάταξη μέσα σε κάποια πλαίσια για να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ατόμων οι οποίοι θα μπορέσουν να λάβουν το λόγο. Ας προχωρήσουμε λοιπόν. Πρώτος, πρώτος, ο κ. Μπουσούτιλ. Πριν ξεκινήσω κύριε Πρόεδρε, και εγώ θέλω να θέσω ένα διαδικαστικό θέμα. Μήπως θα ήταν καλύτερα να ακούσουμε και την άποψη της Κομισιόν και τον, ακούσουμε και από τον κύριο Μπουταρέλη, γιατί θα θέσουν τα ίδια θέματα τα οποία έχουν τεθεί σε συζήτηση από τον κύριο Κέρχοβ. Θα έχουμε μια καλύτερη, πιο εμπεριστατωμένη άποψη για το τι έχουν πει και οι τρεις εκπρόσωποι και τότε μπορούμε να έχουμε και τους τρεις να απαντήσουν στα σχόλιά μας. Έχει νόημα. Έχει νόημα νομίζω να έχουμε χωριστές συζητήσεις να έχουμε χωριστά την στρατηγική κατά της τρομοκρατίας και μετά να ακούσουμε τον κύριο Μπουταρέλ και τον κύριο Τζόναθαν Φάουλ, ο οποίος ε, πιστεύω πρέπει να κάνουμε χωριστές συζητήσεις. Λοιπόν, αν συμφωνείτε κύριε Μπουσούτιλ, να θέσετε ερώτημα παρακαλώ. Εγώ θα μιλήσω για τους αρωτές σώματος, που είναι κάτι το οποίο φυσικά οδηγεί σε ερωτήματα από τους πολίτες μας και ζητούν απαντήσεις. Τα ερωτήματα είναι θεμητά πιστεύω. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα του να πούμε ναι επειδή θέλουμε να προστατεύσουμε την ασφάλεια ή να πούμε όχι γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα των πολιτών. Είναι κάπως πιο πολύπλοκο το θέμα, επομένως πρέπει να προχωρήσουμε πιο πολύ σε βάθος. Οι σαρωτές σώματος είναι μια παρέμβαση στην ιδιωτική ζωή των ανθρώπων. Τίθενται θέματα ιδιωτικότητος και αξιοπρέπειας για τους πολίτες. Κατανοώ επίσης ότι γίνονται αναλύσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν εκθέσεις για τα θέματα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω τι μελετάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν μπορεί να μας ενημερώσει η Επιτροπή για το θέμα αυτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι σε ποιο βαθμό θα είναι αποτελεσματικοί οι σαρωτές σώματος και θα μας δώσουν κάποια απτά αποτελέσματα σε επίπεδο ασφαλείας. Πόσο αποτελεσματική θα είναι σε σχέση με αυτά τα οποία κυκλοφορούν στα αεροδρόμια και τι θα σημαίνει αυτό. Θα περνόμαστε τρεις ώρες πριν φύγει μία πτήση για να μας περάσουν από σαρωτή σώματος. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ποιο βαθμό λοιπόν θα υπάρξει μια, ένας αντίκτυπος επίσης στην υγεία των επιβατών, αλλά κυρίως και των εργαζομένων στα θέματα ασφαλείας στα αεροδρόμια. Και προφανώς τίθεται και το θέμα της ιδιωτικότητα. Και πιο άμεσα. Οι υποτιθέμενοι τρομοκράτες στην πτήση του Ντιτρόιτ θα είχαν εμποδιστεί να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο εάν είχε χρησιμοποιηθεί σαρωτή σώματο. Μπορεί κάποιο να μου δώσει μια σαφή απάντηση, γιατί υπήρξαν διαφορετικέ ερμηνείε σε αυτό το ερώτημα, το οποίο αξίζει μια άμεση απάντηση. Θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε με το συμπέρασμα για το θέμα των σαρωτών σώματο. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα ναι ή με ένα όχι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και περιμένουμε από εσά να πάρουμε μια απάντηση. Σας ξαναλέω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε σχέση με τη χρήση του χρόνου και σας είπα χθε στην αρχή της συνεδρίασής μας Σήμερα το απόγευμα λαμβάνει χώρα μια συνεδρία της Επιτροπής Μεταφορών όπου θα υπάρξει και μια παρουσίαση της Κομισιόν για τους σαρωτές. καλούνται λοιπόν όλα τα μέλη της Επιτροπής μας να συμμετάσχουν σε αυτήν την συνάντηση της Επιτροπής Μεταφορών στις 5 το απόγευμα. Δεν απατώμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν. Ο κύριος Στράσε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιτρομοκρατία είναι σωστό. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το Detroit. Αλλά ήταν ενδιαφέρον το θέμα της πτήσης του Detroit, γιατί διεφάνισε σαφώς ότι εμείς έχουμε αρκετά στοιχεία, αλλά οι μυστικές υπηρεσίες δεν καταφέρνουν να εκτιμήσουν, να σταθμίσουν, να αξιολογήσουν αυτά τα στοιχεία. Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη στοιχείων. Η αστοχία βρέθηκε στο γεγονός ότι δεν υπήρξε η σωστή επεξεργασία των στοιχείων ποια είναι η απάντηση που θέλει να δώσει το Συμβούλιο και η Κομισιόν μετά από τη συνεδρίαση του Τολέντο. Λένε και άλλα στοιχεία. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη λογική καθόλου. Και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό, αυτό το οποίο είπαν οι δύο επίτροποι, Ρέντιν και Μάστρομ, στην ακρόασή τους. Είπαν <clears throat> ότι χρειαζόμαστε βελτιώσεις σε αυτή τη συμφωνία. Το τόνισε η κυρία Ρέντιν ιδιαίτερα για το SWIFT και η κυρία Μάλστομ είπε χρειάζεται καλύτερη αξιολόγηση των στοιχείων που έχουμε συλλέξει και τότε μονάχα θα αποφασίσουμε αν χρειαζόμαστε πρόσθετα στοιχεία. Και κάτι ακόμα. Θέλετε, και αυτό είναι θέμα του Συμβουλίου και της Κομισιόν και φυσικά χρειάζεται υποστήριξη του Κοινοβουλίου, θεωρείτε ότι τα οι ήδη υπάρχοντες, ε, ήδη υπάρχοντες λειτουργούν σωστά. Ο κ. Κύρχοφ, δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να αναφερθώ στο θέμα του θέματος αυτού των σαρωτών σώματος. Μπορεί να είναι θέμα της Επιτροπής ε, Μεταφορών επίσης, αλλά είναι και δικό μας θέμα. Είναι θέμα δημοσίων ελευθεριών. Εγώ ήμουν αρμόδιος για τα θέματα αυτά στο Ηνωμένο Βασίλειο στο παρελθόν. Πρέπει να σας πω ότι Κοιτάσαμε αυτά τα θέματα πριν από πολλά χρόνια. Βέβαια έχει βελτιωθεί η τεχνολογία, αλλά όχι ριζικά. Η τρομοκρατία βεβαίω έχει βελτιωθεί σε σχέση με τις τεχνικές της και δεν μπορεί κανείς ποτέ να προβλέψει τι θα κάνει ένας ε, τρομοκράτης. Είναι απρόβλεπτη η δράση τους και πρέπει να την αντιμετωπίσουν οι δικές μας διοκτικές υπηρεσίες με τρόπους που δεν μπορούμε να τις προβλέψουμε. Δεν είναι απλό να πούμε ότι έχουμε όλοι ένα πολύ καλό σύστημα το οποίο εγκρίνουμε όλοι για τα ανθρώπινα, με λαμβάνοντα υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Αν το δημοσιοποιήσουμε, οι τρομοκράτε θα το εκμεταλλευτούν. Και υπάρχουν και πρακτικά θέματα τα οποία πρέπει να τονίσουμε. <clears throat> θα είμαι παρόν στην Επιτροπή Μεταφορών, αλλά η Επιτροπή Μεταφορών έχει τη δική τη θέση. Για μένα όμω υπάρχει το θέμα του κόστου. Πρέπει να δούμε και τις ε, πολιτικές πρωτοβουλίες που γίνονται με αντανακλαστικό τρόπο ακόμα και από την ε, αγγλική κυβέρνηση σε σχέση με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Δεν πρέπει να προχωρήσουμε έτσι μεμονωμένα, εκτός αν πάμε όλοι μαζί. Δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτός εξοπλισμός σε ένα αεροδρόμιο και όχι σε άλλα. Θα είναι υποχρεωτική ή εθελοντική η χρήση του. Και αν το κάνουμε αυτό, θα φτάσουμε σε μια κατάσταση κατά προφίλ που θέλουμε πολλοί από εμά να το αποφύγουμε και τα δεδομένα, τα δεδομένα που προέρχονται από αυτό τον εξοπλισμό, πώς θα καταστρέφονται στη συνέχεια, πότε θα καταστρέφονται και σε ποια χρήση θα τίθενται. Ξαναγυρίζουμε στη συζήτηση για την κράτηση προσωπικών δεδομένων που είναι θέμα ιδιωτικής ζωής και προστασίας δεδομένων. Δεν πρέπει να θέσουμε περισσότερο βάρος και άχθος στις αεροπορικές συγκοινωνίες <clears throat> όταν οι κυβερνήσεις παίρνουν αποφάσεις οι οποίες δεν έχουν καμία επιστημονική βάση. για τους ρωτές. Τα λέμε και τα ξαναλέμε συνέχεια να κυπεί αυτό το ζήτημα. Και όμως ε, βεβαίως και θέλει να τοποθετηθεί ο κύριος ε, Μπουταρέλη. Thank you, Chairman. Due to the time... πρόεδρε, μια από μας πιέζει ο χρόνος που πρέπει ταχύως να προχωρήσουμε, σας λέω το εξής με συντομία. Ετοιμάσαμε αυτό το έγγραφο συζήτησης για σήμερα. Θα το ανεβάσουμε στο website ε, μετά το μεσημέρι και έτσι θα βρείτε κάποια φρέσκα στοιχεία όσον αφορά την επίσημη τοποθέτηση που συνεχίζει να ισχύει αφού μας ζήτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουμε προς μια διαβούλευση οπότε σε αυτό το χαρτί θα βρείτε και κάποια άλλα στοιχεία καινούργια για το τι προστασία μπορούμε έχουμε για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Και τελικά εξαρτάται από το πότε, πώς, με τι διαδικασίες θα γίνεται αυτή η διαδικασία. Επομένως, Έχουμε εδώ πέρα κάποια μέσα δεύτερη γενιά αλλά έχουμε και προοπτικέ για το μέλλον. Μια που η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίου ρυθμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Πλάσχαρτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Και εγώ θα σα πω ότι θα συζητήσουμε σε Επιτροπή Μεταφορών σήμερα το απόγευμα θα τα ξανασυζητήσουμε. Είναι ένα καινούριο θέμα αυτό. Το 2008 τα ξανασυζητήσαμε. Δεν καταλήξαμε σε καμία δέσμευση. Αλλά είπαμε ότι θα προχωρήσει αυτό το θέμα σε σχέση με την πρόοδο του ζητήματος της προστασίας των δεδομένων και του ιδιωτικού βίου. Το Φεβρουάριο πέρσι ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις Τώρα γίνεται και πάλι αυτή η κουβέντα για τους αρωτές. Είπαμε ότι αυτό θα βοηθήσει για τον νησί της τρομοκρατίας. Υπάρχει πρόβλημα εδώ στο, στο πώς χειριστήκαμε το ζήτημα. Το είπατε ότι ήδη έχουν γίνει κάποια λάθη στη ΣΥΠΑ, ε, τις που απέσπασαν, δεν τι χρησιμοποίησαν όπω έπρεπε. Στην Αμερική ε, η Κομισιόν είχε ένα χρόνο ολόκληρο να κάτσει και να ζυγίσει τα αποτελέσματα διαβούλευση του 2009 και εμεί το ξεκαθαρίσαμε αυτό στο Κοινοβούλιο. Δεν είμαστε κατά των σωρατών, απλώ θέλουμε να πληρούνται κάποιε προποθέσει. Τα είπαμε, τα ξαναείπαμε και τώρα ξαναρχίζουμε από το α. Αφήστε που δεν ξέρουμε κατά πόσο θα σταματάει κάτι τέτοιο του τρομοκράτη. Κύριε Λαμπρινίδη, έχετε το λόγο. Okay. Uh, you mentioned in your presentation 200 million euros will be spent. 200 εκατομμύρια ευρώ είπατε ότι πρόκειται να δαπανηθούν όσον αφορά την έρευνα. Ε, για ασφαλεία. Ποιο αυτά τα διαχειρίζεται, ποιο τα σχεδιάζει. Η, η προστασία του δυτικού βίου τι είναι, είναι μια προπόθεση ε, που θα πρέπει να πληρώνεται τόσο ώστε να ε, εκταμιεύονται να καταβάλουν αυτά τα χρήματα. Μετά. Κάτι που αφορά και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Γιατί πάντοτε, πάντοτε, πάντοτε γίνεται αυτή η κουβέντα στο Συμβούλιο όταν δεν μπορούν να παραστούν τα μέλη της Επιτροπής Φιλικών γιατί είμαστε στο Στρασβούργο. Αυτό είναι παράδειγμα. Επίσης αναφέρεται ότι θα πρέπει να έχουμε ε, ανταλλαγή τη κάθε λίστα που υπάρχει πληροφορίε για του τρομοκράτε με του Αμερικάνου, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ισχύει όμω ή δεν ισχύει το ότι έχουμε αυτέ τι διμερείς συμφωνίε για κατάρριξη τη βίζας που έχουν όμως ως προϋπόθεση το ότι θα πρέπει και τα κρατη να δώσουν στους Αμερικάνους τις δικές τους λίστες για τρομοκράτες. Τι θα γίνει, θα ζητήσουμε να υπάρχει κάποιο είδους αμοιβαιότητα. Θα υπάρχει νομική βάση για τέτοια ανταλλαγή. Excusez-moi, euh, j'ai trois questions très courtes. Euh, Τρεις πάρα πολύ σύντομες ερωτήσεις γιατί είχαμε κάτι πάρα πολύ παράδοξες ε, περιπτώσεις πρόσφατα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την ασφάλεια και δεν αναφέρομαι μόνο στο Detroit κάτι το οποίο ήδη συζητήθηκε αλλά είχαμε τότε εκείνη τη βόμβα στη βαλίτσα ενός Σλοβάκου και στο Μόναχο. Πιο μετά εντοπίστηκαν ίχνη βόμβας στο λάπτοπ ενός ταξιδιώτη που εξαφανίστηκε. Δεν καταλαβαίνουμε. Ποιος τα έκανε αυτά, ποιος ήταν αυτός ο οποίος μετά εξαφανίστηκε. Όλα αυτά μας έχουν πάρα πολύ βαθιά προβληματίσει και θα πρέπει να αναζητηθούν εξηγήσεις. Δεύτερη ερώτηση. Η... Το το πόσο απειλεί η τρομοκρατία την κάθε χώρα στην Ευρώπη. Για πέστε μας. Γιατί πολλές φορές διαβάζουμε πάρα πολύ χάζα πράγματα στον τύπο. Και καταλήγουμε στο ότι μετά από αυτά τα άρθρα ότι δεν υπάρχει απειλή στην Ευρώπη, σε κάποιες χώρες τέλος πάντων, από την τρομοκρατία. Τρίτη ερώτηση. Ποια είναι η σχέση τρομοκρατίας οργανωμένου κλίματος. Για πέστε μας έτσι σε αδρές γραμμές τι συνδέσεις υπάρχουν μεταξύ εργομένου εγκλήματος και τρομοκρατίας. Άλβαρο. Για τους ρώτες. Είναι κάτι που το, έχουμε συζητήσει, το συζητούμε πάρα πολύ συχνά και εμείς ως ε, πολιτικοί προσπαθούμε να θέσουμε ένα πλαίσιο για το τι θα γίνει, ε, πώς θα εφαρμοστεί η τεχνολογία και όχι από τεχνολογία να ξεκινάμε γιατί ε, στην Αμερική έχουν κάποιες τεχνικές στιγμές προδιαγραφές, έχουν και διάφορα άλλα προβλήματα ε, για το πόσο προσβάλλει το εθνικό βίο. Επίσης υπάρχουν θέματα θερμοκρασίας, τι περνάει από το κάθε υλικό. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουμε μόνο αν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις ακμέρους τεχνολογίας. Προσοχή, γιατί δεν πρέπει να φτάνουμε να θεωρούμε τεχνολογία είναι κάτι σαν Ευαγγέλιο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας. Από το 2001 έχουν περάσει 10 χρόνια. Ακόμα δεν έχουν προχωρήσει πολύ, άρα κάτι πάει στραβά συλλογή δεδομένων, ε, ανταλλαγή δεδομένων. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει αφού δεν έχουμε προχωρήσει όσο θέλαμε. Άρα, να κάτσουμε και να σκεφτούμε τι στρατηγική θέλουμε να χαράξουμε και όχι να κολλάμε στα ίδια και στα ίδια. Λοιπόν, ή δεν είναι το μαγικό ραβδί η ανταλλαγή και η συλλογή δεδομένων, ή θα πρέπει να σκεφτούμε πώ θα το χρησιμοποιήσουμε καλύτερα. Μετά, τα προβλήματα αμοιβιότητα με τη ΣΥΠΑ. Αν δίνουμε στοιχεία, θα πρέπει να λαμβάνουμε κιόλα. Άρα, η λέξη κλειδί είναι συνεργασία. Εδώ χρειάζεται συνεργασία και να προχωρήσουμε προς τεχνολογίες που να είμαστε βέβαιοι το πώς θα δουλεύουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για τη χρήση των δεδομένων είναι η πιο σημαντική συζήτηση από όλες που πρέπει να γίνει εδώ. Δεν θέλω να επιμείνω μονάχα στο θέμα των συμπερασμάτων του Detroit. Η συστημική αστοχία που αναγνωρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση είναι σημαντική, αλλά μας ενδιαφέρει πάντα το πρόβλημα της ουσίας, η χρήση αυτών των δεδομένων και γιατί υπάρξει, υπήρξε αυτή η συστημική αποτυχία. Αν εμείς θέλουμε να έχουμε ένα κέντρο για να μαζεύουμε όλα τα στοιχεία για τους τρομοκράτες, όπως αναφέρεται αυτό το γενικό κέντρο όπου συγχωνεύονται όλες οι πληροφορίες. Θα περιλαμβάνει και τις οικονομικές πληροφορίες που βγαίνουν από δικαστικές διαδικασίες με κάποιες εγγύσεις, τότε θα είναι πραγματικά σημαντικές αυτές οι πληροφορίες. Είναι σημαντικές πληροφορίες. Θα είναι τμήμα λοιπόν οικονομικές πληροφορίες. Παραδείγματος χάρη αυτές που έρχονται από το SWIFT μπορούν να έχουν κάποια χρήση σε περιοχές που ενδιαφέρουν την ε, Ευρώπη για χώρες όπως το Μαρόκο που μπορούν να συνεργάζονται ή να δίνουν πληροφορίες στην ε, Αλκάιδα ή άλλες χώρες οι οποίες μπορεί και αυτές να μπορέσουν να μεταβιβάσουν πληροφορίες και οι οποίες θα έχουν άμεση πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές που ε, έχουμε εμείς στη διάθεσή μας. Eh, Και Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τους σαρωτές ε, σώματος. Πριν από δύο εβδομάδες ήμουν στο Σχίπολντ για να ρίξω μια ματιά. Και μετά από δύο χρόνια όπου υπάρχουν εξελίξεις στην τεχνολογία, οι σαρωτές σώματος νομίζω ότι είναι αρκετά καλοί, αρκετά ανεπτυγμένοι το θέμα που μένει να απαντηθεί είναι αν είναι χρήσιμη. Μήπως είναι μια... παίζουμε με όπλα μια μάχη που την έχουμε χάσει εκ των προτέρων. Η συζήτηση για τους αρωτές σώματος είναι τεχνικό θέμα. Μπορούμε να αγοράσουμε ασφάλεια με την τεχνολογία, μπορεί να μην μπορούμε. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι οι σαρωτές σώματος θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για όλες τις πτήσεις και τις ευρωπαϊκές πτήσεις. Νομίζω ότι αυτό θα οδηγήσει σε ένα απίστευτο πολλαπλασιασμό αυτού του, του εξοπλισμού. Και το ερώτημα είναι, θα δουλέψει? Μήπως υπάρχουν άλλα μηχανήματα που μπορούν να είναι εξίσου αποτελεσματικά ή καλύτερα, πιο αποτελεσματικά. Επίσης πρέπει να κοιτάξουμε βεβαίως και τους κινδύνους για την υγεία από τη χρήση αυτών των ε, σαρωτών. Φυσικά, δεν πρόκειται να επιλύσουμε το πρόβλημα μόνο με σαρωτές σώματος. Το θέμα είναι θα βοηθήσουν όμως. Ο κύριος ε, Ντεκέρκοβ μίλησε για μεγαλύτερη προσπάθεια στο επίπεδο της πρόληψης. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Γιατί δεν θα πρέπει να μπλέκουμε την ε, πρόληψη με την καλή κοινωνική συνοχή. Νομίζω θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μηχανήματα έτσι πιο οπτικά για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία. Τώρα, διερωτώ γιατί ανοίγεται αυτό το κουτί της Πανδώρας. Ε, για την καταπολέμηση της δημοκρατίας χρησιμοποιώντας δηλαδή τέτοια μηχανήματα. Ο κύριος Λαμπρινίδης. Δεν έχουμε χρόνο. Το SWIFT είναι τεράστιο θέμα. Παρακαλώ τους συναδέλφου να μην επαναλαμβάνουν αυτά που είπαν άλλοι. Πρέπει να ακούσουμε από τον Τζόναθαν Φολ και τον κύριο Μπουταρέλη και πρέπει να προσέξουμε. Ε, ένα λεπτό. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Ένα λεπτό και να το τηρήσουμε όλοι μας. Εγώ νομίζω το τήρησα. Τι έκανα. Ε, το υπερεύνη κατά 10 δευτερόλεπτα το πολύ. Συμφωνήσαμε ότι έχουμε μια συγκεκριμένη μέθοδο και μια διαδικασία σε αυτή τη συζήτηση. Σας ε, κάνω έκκληση να σεβαστείτε το χρόνο για το καλό και των υπολείπων συναδέλφων. Και για να συζητήσουμε σωστά, αλλά και να δώσουμε, να μπορέσουμε να δώσουμε το λόγο στα περισσότερα δυνατά μέλη της Επιτροπής. Σας κάνω λοιπόν έκκληση να σεβαστείτε τη συμφωνία και τη διαδικασία. Κυρία Λάτφορντ. Δέκα λεπτά το πολύ. Um, Σας σέβομαι κύριε Ντακέρκο προσωπικά αλλά δεν σέβομαι ιδιαίτερα τη θέση ότι ξαφνικά μιλάμε για αυτά τα θέματα, λες και είναι φοβερή ε, καινοτομία ε, και ότι το πρόβλημα με την ε, τρομοκρατία είναι ότι δεν συνδυάζουμε τις πληροφορίες. Εδώ και δέκα χρόνια το λέμε. εδώ και χρόνια εγώ μιλάω για τα μαθήματα από την 11η Σεπτεμβρίου. εδώ και χρόνια μιλάμε για δεδομένα και άλλα δεδομένα και κόντρα δεδομένα. Ποτέ δεν, κάνουμε, δεν τα κοιτάμε όμως, ε, ποτέ δεν, υπάρχει, δεν κοιτάμε αν υπάρχουν διαφορετικές πηγές. Νομίζω ότι χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το δέντρο. Και εγώ, όπως και άλλοι βουλευτές, θέλω να υπάρχουν ε, δεδομένα, επιμερισμός των δεδομένων, ε, με εξασφάλιση της ιδιωτικότητας όμως. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Έρχεστε εδώ πέρα και μας λέτε ξανά και ξανά ότι υπάρχει πρόβλημα και δεν συνδυάζουμε τα δεδομένα πότε θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Πότε θα συνηθου, ε, θα συνειδητοποιήσουμε, ας πούμε, να το ξέρουμε. Πότε θα λάβουμε υπόψη μας μάλλον ότι χρησιμοποιούν νέο αίμα. Ξέρουμε το πρόβλημα της ριζοσπαστικοποίησης. Χθε ακούσαμε υπουργού, ε, δικηγόρους ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο να λένε ότι η εισβολή της, των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ ήταν αντίθετη στο διεθνές δίκαιο. Και όμως ο Τόνι Μπλερ προχώρησε. Επίσης, ε, διαμαρτυρόμαστε για την κράτηση επαόριστον. Τι κάνουμε για όλα αυτά τα θέματα. Κύριος Ντεγιόγκ. Eh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κερκόβ για την παρουσία του. Είπε ότι ήταν απαραίτητο να εργαστούμε πολύ στον τομέα της πρόληψης. Βλέπουμε πράγματι να υπάρχει μια εξέλιξη προς μέτρα κατασταλτικά τα οποία όλο και περισσότερο εφαρμόζονται. Αν θέλουμε να έχουμε μεγαλύτερη καταστολή, θα πρέπει να τα συνδέσουμε με την εξωτερική μας πολιτική, με χώρες οι οποίες βρίσκονται σε αξιοθρύντη κατάσταση, όπως το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η Εμένη. Και θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε εμείς να δημιουργήσουμε τρόπους αντιμετώπισης των τεραστίων προβλημάτων, των δημογραφικών προβλημάτων, παραδείγματος χάρη σε χώρες όπως αυτές που ανέφερα για την περίπτωση της Ιεμένης, είναι εύκολο να κάνετε μία διάσκεψη και νομίζω ότι έχει λύσει το πρόβλημα. Η Ιεμένη είναι πάρα πολύ πολύπλοκη και πολυεδρική. Για να βοηθήσετε την κυβέρνηση στην Ιεμένη θα πρέπει να αντιμετωπίσετε προβλήματα μέσα στον πληθυσμό, προβλήματα διαφθοράς μέσα στην κυβέρνηση. Είναι ένας πολύ πολύ πολύπλοκος χώρος η ΕΜΕΝ. Δεν είναι μονάχα το θέμα της τρομοκρατίας. Και για τα θέματα της πρόληψης θα ήθελα να έχω στοιχεία για κάθε χώρα και να ξέρουμε πώς θα αναλύσουμε τα προβλήματα αυτών των χωρών. Μόνο έτσι θα μπορούσαμε ίσως να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Τέλος, πιστεύω ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει και το πρόβλημα της ε, Μέσης Ανατολής που είναι η πηγή όλων αυτών των προβλημάτων οι άνθρωποι στη Γάζα που είναι αποκομμένοι από οποιαδήποτε βασική υπηρεσία. Έτσι εκτρέφεται η τρομοκρατία αν τα άτομα αυτά δεν έχουν καμία προοπτική για το μέλλον στη ζωή τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει απολύτως τίποτα για αυτά τα θέματα. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για αυτά τα ζητήματα εξάλλου. Ετέθηκε το θέμα του Γουαντάναμο, λέει ο κύριος Κλάες. Ο πρόεδρος Ομπάμα είχε υποσχεθεί ότι θα κλείσει το Γουαντάναμο και θα φέρει τους κρατούμενους ενώπιον τακτικών δικαστηρίων. Και κάποιοι από αυτούς θα είχαν απελευθερωθεί. Κάποιοι επίσης θα μπορούσαν να έχουν έρθει στην Ευρώπη. Και τώρα υπάρχουν αυτοί που λένε ότι ήταν πάρα πολύ βεβαιασμένη η απελευθέρωση αυτών των ανθρώπων όταν τα άτομα αυτά βρισκόντουσαν σε επαφή με τρομοκρατικές ομάδες και είχαν εμπλακεί σε τρομοκρατικές ενέργειες. Και στο Γουαντάναμο υπάρχουν καμιά κοσαρία κρατούμενοι από την Ιεμένη, δεν ξέρω αν είναι ακριβώς σωστά τα στοιχεία αυτά. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τι έγινε στο πλαίσιο αυτό <clears throat> στην πτήση του Ντιτρόιτ. Ο Ομπάμα λοιπόν δεν θα κλείσει το Γουαντάναμο όσο γρήγορα είχε πει λόγω αυτής της υπόθεσης. Η κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, από την περίπτωση του Ντιτρόιτ, εγώ έχω μερικέ απορίε. Ο ίδιο ο πατέρα του δράστη είχε ενημερώσει εγκαίρω τι Αμερικανικέ Αρχέ. Η συμπεριφορά του ιδίου ήταν προφανή. Πώ ήταν δυνατόν ο δράστη να καταφέρει να μεταφέρει εκρηκτικά, αν υπήρχαν σαρωτέ, θα μπορούσαν να είχαν ανοιχνεύσει τα εκρηκτικά. Γιατί απέτυχαν οι μυστικέ υπηρεσίε τη Αμερική με ανταλλαγή πληροφοριών με το αεροδρόμιο να τον εντοπίσουν. Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί πρώτα αποφασιστεί αν πρέπει να μπουν ή όχι οι σαρωτέ. Όσον αφορά του σαρωτέ, διαβάζοντα την τεχνολογία του, θεωρώ ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία. Γιατί υπάρχουν δύο τύποι σαρωτών, οι millimeter wave και οι pack scatters. Ο πρώτο, το πρώτο είδο βομβαρδίζει τα σώματα με ραδιοκύματα και το δεύτερο με ραδιονεργό ακτινοβολία. Σε άτομα που έχουν απεινιδωτέ ή άλλα μηχανήματα προστασία τη καρδία, πιθανόν να υπάρχουν κίνδυνοι. Στέκομαι κυρίω όμω στην παραβίαση τη προσωπική αξιοπρέπεια. Και το ερώτημα μου είναι ακριβώ αυτό που έχει θέσει η κυρία Ρέτινγκ τελικά από το φόβο τη επικράτηση τη τρομοκρατία θα πρέπει να παραβιάζονται προσωπικά δεδομένα, η ιδιωτική ζωή και ο φόβο να καθορίζει αν θα παραβιάζονται ή όχι θεμελιώδη δικαιώματα. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί πρέπει να δουν την εξωτερική του πολιτική για να μην δημιουργούνται προβλήματα, γιατί η τρομοκρατία πολλές φορές ε, υποβόσκει εκεί που υπάρχουν και αλλοπρόσαλες εξωτερικές πολιτικές. Και πρέπει η Αμερική να προσέξει πώ συμπεριφέρεται σε διάφορε χώρε. Δεν αιτιολογώ την τρομοκρατία, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να πανταχθεί η τρομοκρατία, όχι σε βάρο όμω θεμελιωδών ανθρωπινών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Thank you. And Mr. Bonds. Ο κύριος Μποντ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι Ηνωμένες, το, οι του, των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούν ότι η λύση για το πρόβλημα της τρομοκρατίας είναι η στρατιωτική δράση σε μια σειρά μουσουλμανικών κρατών. Αυτό όμως οδηγεί σε περισσότερη ζωσπαστικοποίηση των μουσουλμάνων στη χώρα που γίνεται η δράση και στις χώρες οι οποίες κάνουν αυτή την επέμβαση. Δεν είναι προστασία το να στέλνουμε στους στρατιώτες μας να σκοτωθούν. Η χρήση νέων προσώπων σημαίνει <clears throat> ότι πρέπει να παρακολουθούνται ε, και οι παλιοί και οι καινούργοι τρομοκράτες μέσα σε εισαγωγικά. Τέλος, θα πρέπει να έχουμε μια νέα πολιτική στη Μέση Ανατολή και να αποστασιοποιηθούμε από τη στάση των ΗΠΑ που μονάχα οξύνει την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Τέλος, η κυρία Ιντβέλτ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ολόψυχα υποστηρίζω αυτό που είπαν πολλοί, συνάδελφοι, η Βαρονέσα Λάτφορτ παραδείγματος χάρη, φαίνεται ότι το Συμβούλιο δεν ακούει τίποτα, δεν ακούει καμία επίκριση από καμία πλευρά. Γιατί δεν βλέπω να έχει προκύψει μια νέα αξιολόγηση, κάποια νέα σκέψη για τα θέματα αυτά, απλώς το Συμβούλιο αντιδρά σπασμωδικά. Στις Ηνωμένε Πολιτείες γίνεται τώρα μια πλήρης ανάλυση των αντιτρομοκρατικών μέτρων που επιτρέψει στον εαυτό της να έχει κάποια στοιχεία αυτοκριτικής. Γιατί δεν το κάνει αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν διαμφισβητεί τις μεθόδους που ακολουθούμε. Μέχρι ότου αρχίσει να αναλύει τις μεθόδους στο Συμβούλιο, δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και δεν πρόκειται να αποκομίσουμε τίποτα αυτές τις συζητήσεις. Το ερώτημά μου είναι το εξή. θέλουμε να προχωρήσουμε με νομοθεσία για τις πληροφορίες, πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα κτλ. Αλλά οι αρχές φαίνεται να αποκτούν νόμιμη πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα σε ευρύτατη κλίμακα. Φαίνεται ότι στις ΗΠΑ η FBI είχε πρόσβαση σε στοιχεία που οδήγησαν σε εκβιασμό εταιριών, κυρίως αυτό. Γι' αυτό χρησιμοποίησαν αυτά τα στοιχεία. Όλα αυτά έρχονται ενώπιον δικαστηρίων. Το ερώτημα μου στον κύριο Ντεκέρκοφ είναι το Συμβούλιο θα τα εξετάσει αυτά τα θέματα ή όχι. Κύριε Ντεκέρκοφ, έχετε το λόγο. Καταλαβαίνετε τώρα τη δυσκολία του να έχετε να αντιμετωπίσετε σχεδόν 20 διαφορετικές παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Πρωτού όμως περάσουμε στο επόμενο θέμα και ακούσουμε τον κύριο Μπουτάρελ και τον κύριο Φάουλ. Εμείς θα χαρούμε ιδιαίτερα να ακούσουμε τις συνολικές σας παρατηρήσεις για τα διάφορα θέματα που ακούσατε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να αντιμετωπίσω τα ερωτήματα με τη σειρά που έχουν τεθεί και να είμαι σύντομο γιατί ξέρω ότι έχετε και άλλα σημαντικά θέματα να εξετάσετε. Μια γενική απάντηση καταρχήν για τους σαρωτές σώματος. Θα υπάρξει σήμερα το απόγευμα μια συζήτηση σε βάθος και δεν έχουμε ακόμα δει την έκθεση της Κομισιόν. Είπα και εγώ ο ίδιος όταν μου τέθηκε αυτό το ερώτημα ότι δεν μπορούμε ακόμα να πάρουμε κάποια θέση μέχρι ότου έχουμε τα πορίσματα της Επιτροπής που εξετάζει τα θέματα αυτά και της Επιτροπής για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας και επίσης να ξέρουμε το αντίκτυπο για την υγεία την ανθρώπινη και την αποτελεσματικότητα αυτών των σαρωτών. Αυτά που ξέρουμε από πειράματα στο Ηνωμένο Βασίλειο και από πειράματα στις κάτω χώρες, στο Σχύπχολ είχαν δοκιμάσει σαρωτές της νέας γενιάς στους ε, πιλότους και το προσωπικό καμπίνας στην αρχή ήταν λιγάκι προσεκτική. Αλλά μετά από μια εβδομάδα, ότι όταν είδανε τι υπάρχει στις οθόνες και υπάρχει λογισμικό το οποίο θαμπώνει λιγάκι τις εικόνες που προέρχονται από τους ε, ε σαρωτές, δεν υπάρχει καμία αποθήκευση των στοιχείων αυτών από τους αρωτές λένε και θα ήταν χρήσιμο η Επιτροπή σας να πάει στο Σύπολ και να το ελέγξει αυτό και θα το κάνω και εγώ αλλά περιμένουμε παρόλα αυτά την έκθεση της Κομισιόν. <clears throat> Κύριε Στράσε, ίσως δεν είμαι αρκετά σαφής, τόνισα ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιώσουμε την διασταύρωση των δεδομένων. Δεν είπα όμως τότε ότι δεν πρέπει να συλλέξουμε περισσότερα δεδομένα και υπάρχει μεγάλη έλλειψη ισορροπίας. Εμείς δεν παίρνουμε στοιχεία PNR σε όλα τα κρατη ενώ όλες οι εταιρείε δίνουν στοιχεία στους Αμερικανούς. Πρέπει να κάνουμε και τα δύο λοιπόν. Μιλήσατε για το SIS. Το SIS είναι το καλύτερο αστυνομικό εργαλείο που έχουμε στην Ευρώπη. Είναι σημαντικό συνοδευτικό μέτρο γιατί δεν έχουμε πια τους διαμεθοριακούς ελέγχους. Πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό το εργαλείο. Το VIS επίσης είναι το ίδιο πράγμα. Θα είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Είπατε κύριε Κύρχοφ ότι όσο πιο πολύ δημοσιοποιούμε αυτά που κάνουμε, τόσο πιο πολύ γνωρίζουν οι τρομοκράτες. Φοβάμαι ότι σε αυτή την Επιτροπή θα πρέπει να έχουμε κλειστές συνεδριάσεις μερικές φορές, γιατί πράγματι δεν είναι ιδιαίτερα σόφρον να εξηγούμε πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του SWIFT και τα στοιχεία για τους επιβάτες. Δεν είναι καλό αυτό να το κάνουμε, αλλά μιλάω από τη δική μου πλευρά. Αν δίνετε όλες τις λεπτομέρειες, δίνετε πολλές πληροφορίες στους, στους ε, τρομοκράτες. Αλλά το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται πλήρως η στρατηγική διαχείριση πληροφοριών μπορεί να αναπτυχθεί μονάχα αν υπάρχει μια συνένεση στο Κοινοβούλιο, γιατί υπάρχει μεγάλη αναγκή για κάτι τέτοιο. Οι σαρωτέ σώματο. Τι εμπλέκεται. Το θέμα δεν είναι αν πρέπει να του χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Το θέμα είναι αν πρέπει να του χρησιμοποιήσουμε σαν πρωτογενέ στοιχείο ελέγχου των επιβατών και όχι σαν δευτερεύον στοιχείο ελέγχου. Θα είναι τότε υποχρεωτικό ή εθελοντικό και το χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις περιστάσεις ή σε ορισμένες περιπτώσει και σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία. Αυτό πρέπει να συζητήσετε σήμερα το απόγευμα. Για το ερώτημα του κυρίου Λαμπρινίδη. Θα το απαντήσει νομίζω ο Τζόναθαν Φόλ, ίσως καλύτερα από μένα. Θα έλεγα <clears throat> εγώ. Υπάρχει αυτή η Επιτροπή των Κρατών Μελών που αποφασίζει που πρέπει να υπάρξει επένδυση κονδυλίων. Και αν μας ενδιαφέρει η ιδιωτικότητα, αν διαβάσετε την πρόσφατη ανακοίνωση της Κομισιόν και την έκθεση των εμπειρογνωμών, θα δείτε ότι δεν έχουμε μία καθήλωση με την υψηλή τεχνολογία. Θέλουμε να έχουμε εργαλεία τα οποία είναι φιλικά προς την ιδιωτικότητα και είμαι πεπισμένο ότι όσο περισσότερο αναπτύσσουμε αυτά τα εργαλεία θα πρέπει να τα κάνουμε όλο και πιο προστατευτικά για την ιδιωτική ζωή. Και μία ιδέα ήταν να έχουμε ένα πρότυπο στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να έχει την ετικέτα της φιλικότητας προς την ιδιωτική ζωή, κάτι το οποίο θα επέτρεπε και θα υποχρέωνε και τη βιομηχανία να αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες. Αν το κάνει αυτό η Ευρώπη, <clears throat> πιέζουμε την βιομηχανία μας και θα του βοηθήσουμε να έχουν ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο κόσμο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Σαν τα καθαρά <clears throat> ε, αυτοκίνητα θα έχουμε καθαρού σαρωτές. Θα έχουμε πρωτοπορία σε παγκόσμια τεχνολογία. Δηλαδή να προστατεύουν την ιδιωτική ζωή θα είναι καλό αυτό και θα είναι καλό και για τη βιομηχανία. Είπατε επίση για το θέμα τη αμοιβαιότητα. Μα αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλο και περισσότερο. Με το να έχουμε συμφωνήσει με τι ΗΠΑ για πολλά θέματα αν εμπλέκεται η αρχή της αμοιβαίωτος. Αν δείτε την ενδιάμεση συμφωνία για το SWIFT σε σχέση με την πρώτη, η οποία δεν ήταν μια επίσημη συμφωνία, απλώς μια συμφωνία κυρίων, τι πετύχαμε. Πετύχαμε πιο ενεργή πρόσβαση της Ευρώπης στα δεδομένα που συλλέγονται στις ΗΠΑ και πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη πρόσβαση. Συμμερίζομαι λοιπόν τι απόψει σας για το θέμα αυτό. Κυρία Ανκή, είναι μοναδική αυτή η περίπτωση στη Σλοβακία. Εγώ δεν ξέρω τι λεπτομέρειε δεν θέλω να τη σχολιάσω. Μπορώ να σας πω απλώ και δεν αποκαλύπτω μυστικά. Ο υπουργό Εσωτερικών της Σλοβακία <clears throat> έχει ζητήσει συγγνώμη ενώπιον όλων των ομολόγων του των Υπουργών Εσωτερικών για μια επιχείρηση η οποία δεν ήταν παραδεχτεί. Για την περίπτωση του Μονάχου και εκεί δεν έχω συγκεκριμένες πληροφορίες μέχρι τώρα. Θα το συζητήσω με τον κύριο Ντεμεζιέρ. Είναι πράγματι ένα πρόβλημα. Προφανώς. Αν δούμε κάποιον ο οποίος έχει ίχνη εκρηκτικά στον υπολογιστή του και δεν το συλλαμβάνουμε, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Μας είπατε για την κατάσταση της απειλή. Δεν θα, δεν θα απαντήσω τώρα σε κάποια μεταγενέστερη ευκαιρία μπορώ να το αναφέρω. Σε δύο λεπτά δεν μπορώ να δώσω μια πλήρη απάντηση γιατί ποικίλει από μια χώρα σε μια άλλη. Κάποιες χώρες έχουν μειώσει το επίπεδο ε, επαγρύπνησης ενώ το αύξησε το Ηνωμένο Βασίλειο. <clears throat> Σχέσεις με οργανωμένο έγκλημα και τους τρομοκράτες αρχίζει να γίνει ανησυχητικό. Και υπάρχει τώρα ένα τόξο κρίσης που αναπτύσσεται και φτάνει μέχρι τη Δυτική Αφρική η, τα ναρκωτικά που έρχονται από τη Λατινική Αμερική, το λαθρεμπόριο ανθρωπίνων όντων και όπλων, όλα αυτά είναι δραστηριότητες πολλαπλές που πολλές φορές τις ασκούν οι ίδιες ομάδες και αλληλοενισχύονται. Είναι κάτι για το οποίο αρχίζουμε να εργαζόμαστε πιο ενεργά και υπάρχουν κοινέ πολιτικές τις οποίες πρέπει να αναπτύξουμε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Για το ερώτημα για τις σχέσεις με το βόρειο τμήμα της Αφρικής, το Μαρόκο και τα κέντρα συγκέντρωσης και συγχώρευσης πληροφοριών. Όταν έχουμε ένα τέτοιο συγχώρευση δεδομένων και όταν κάτι μέλη πρέπει να το κάνουμε, θα ήταν καλό από παιδαγωγική άποψη. Είναι η χάρτα που σχεδόν ενεκρίθη την προηγούμενη Παρασκευή στη Μαδρίτη να προβλέψουμε ότι ένας από τους ρόλους αυτού του δικτύου είναι να βοηθήσει άλλες χώρες στο δίκτυο και τρίτες χώρες ακόμα να αναπτύξουν τέτοια κέντρα. Όταν ήμουν στο Πακιστάν πριν από μερικούς μήνες, ένα από τα βασικά <clears throat> σχέδια ήταν η δημιουργία ενός κέντρου όπως το ΣΕΝΣΕΑΚ στην Ισπανία, το ΖΕΤΑΚ στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να υπάρξει η ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών, γιατί δεν είναι εύκολο το να διασταυρώνει κανείς τα στοιχεία. Για το ερώτημα τώρα της αξιολόγησης δεν παρακολούθησα τώρα όλη την ε, ακρόαση κυρία Ιντβέλτ νομίζω ότι οι επίτροποι ήταν παρόντες εκεί και έχουμε διάφορες ε, αξιολογήσεις, την ε, Joint Review για το PNR που αφορά την συμφωνία με τις ΗΠΑ που θα έλθει στο φω σε μία-δύο εβδομάδες. Αυτή είναι μια δυο εβδομάδε. αυτη ειναι μια αξιολογηση τη συμφωνία μας που νομίζω θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Ο δικαστής Μπρίγκερ σε μία εβδομάδα θα, οδηγήσει, θα δώσει μια δεύτερη έκθεση για την συμφωνία με το SWIFT. Θα μάθουμε πολλά πράγματα λοιπόν σε σχέση με την προσθέμενη αξία του συστήματος και η έκθεση αυτή θα είναι στην διάθεσή σας. Ξεκινώντας από τέτοιες εκθέσεις θα πρέπει να αξιολογήσουμε τους μηχανισμούς. Δεν έχω δώσει μια πλήρη σειρά απαντήσεων. Ίσως λυπάμαι αν κάποια ερωτήματα δεν τα έχω διεξέλθει επαρκώς. Αυτά ήθελα να πω όμως. Thank Ευχαριστώ. Όσοι την έλαβαν απαντήσεις, να τις ξαναυποβάλουν εγγράφος και πάρουν εγγραφή απάντηση. Και γραμματεία παρακαλώ να βοηθήσει όσο γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Προσωπικά με εντυπωσίασε αυτό το οποίο είπατε και πρόκειται να γίνει σε δύο εβδομάδες στην μια δεύτερη καινούργια αξιολόγηση του SWIFT. Το PNR, PNR λέει ο... Όχι, όχι το SWIFT, για το SWIFT λέει, λέει κύριε Νετφέλτ. Ορίστηκε ο δικαστή της Μπριγκέρ δεν ξέρω με ποια ακριβώς διαδικασία, ούτως ώστε να εξετάσει το θέμα. Ε, ναι, ήδη την πρώτη σύγκριση και θα υπάρξει και μία δεύτερη την επόμενη εβδομάδα, οπότε μπορείτε όλοι να ενημερωθείτε με πληροφορίες για την προστιθέμενη αξία όσον αφορά την ασφάλεια και το σύστημα. Μα τι αυτό έχει γίνει σαν αναστείο τη Δευτέρα. Θα αρχίσει προσωρινά να ισχύει, όπως είπε η Ισπανική Προεδρία, το SWIFT. Και μας λέτε τώρα ότι εκ των υστέρων αμέσως μετά πρόκειται εμεί να λάβουμε τη δεύτερη έκθεση. Δεν και θυμάμαι με περιορισμένη σύνθεση, τα είχαμε συζητήσει εδώ και τότε συζητήσαμε την προστιθέμενη αξία. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό εκ νέου. Τα συζητήσαμε, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρόκειται για μια διαρκή διαδικασία για την οποία φυσικά και εσείς ε, είχατε υποπτία. Είναι Καλά, φεύγω, φεύγω πρόεδρε μια που ήρθατε. Απλώς σας λέω ότι το timing είναι εκπληκτικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή έχει πέντε εργάσιμες ούτως ώστε να μπορέσει να σκεφτεί για αυτήν την συμφωνία που αρχίζει να ισχύει και κατόπιν θα έχουμε αυτή την έκθεση που είναι τόσο σοβαρή η οποία θα ληφθεί υπόψη. Τι να σας πω, μπορεί να φταίω εγώ, εγώ, εγώ. Κύριε Πρόεδρε, έχετε το λόγο. That's okay. I'm still available. That's okay. We pass on the following point swiftly. But we already started. Okay. Okay, having covered, having covered this point, let's... Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό και πάμε εις το επόμενο. Ο πρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Λέει ο κύριος Fall. Είχα αυτό το έξτρα τεταρτάκι, ούτως ώστε να παρακολουθήσω τι γίνεται και να μπορέσω να ξέρω ότι παρεξηγήσεις θα πρέπει να διευκρινίσουμε. Πάντως, ό,τι ερωτήσει έχετε, ευχαριστώ να απαντήσω. Είχαμε αυτή την βράχη πρόθεσμη προσωρινή συμφωνία με τις ε, ΕΠΑ για το SWIFT, διαβιβάστηκαν τα σχετικά γράφα ή στο Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, περιμένει την συνένεση του Συμβουλίου και ελπίζω ότι και εσείς επομένως θα διαβουλευτείτε και κάτσετε να κάνετε μια πλήρη ανάλυση αυτής της συμφωνίας αλλά και της εκθέσεως του δικαστού Μπριγκέρ που ολοκληρώνει τώρα το έργο του οπότε θα έχετε το σχετικό κείμενο. Τις αμέσως επόμενες μέρες. Και σας τονίζω ότι και τώρα πρόκειται για μια πάρα πολύ σημαντική πτύχη της διαδικασίας ε, σύμφωνης Πού προβλέπει η συνθήκη της εις στο άρθρο 186. Αυτό είναι όμως κάτι το διαφορετικό σε σχέση με την προσωρινή θέση σε ισχύ της συμφωνίας. Σύμφωνα με όσο προβλέπει η Συμφωνία Ένωσης, είπα, αρχίζει αυτή η συμφωνία να ισχύει από την 1η Φεβρουαρίου, όπου και δεν θα έχουμε καθόλου τρόπο κανένα είδου κενό, παραθυράκι για τις σχετικές ε, πληροφορίες που πρέπει να παρέχουμε στις ΕΠΑ. Συμφωνείτε συμφωνία γνώμη, επομένω είναι κάτι το διαφορετικό σχέση με την προσωρινή θέση σε ισχύ τη συμφωνία. Όμω, αν δεν δώσει τη Συμφωνία γνώμη του το Κοινοβούλιο, τότε θα πρέπει να σταματήσει αυτή η προσωρινή εφαρμογή της ε, συμφωνίας. Αυτό είναι σαφές και επομένω ε, και αυτό εσείς θα το λάβετε υπόψη και θα το συζητήσετε όπως πρέπει. Τώρα, προκαταλαμβάνοντας κατά κάποιο τρόπο τη σχετική ερώτηση, το κατά πόσον, όπως ε, είπε προηγουμένως η Βάρνη Λάτφορντ και άλλοι, για το κατά πόσον θα έχουμε μια γενική αναθεώρηση της αντιτρομοκρατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα των μηχανισμών ανταλλαγής πληροφοριών. Η απάντηση είναι καταφατική. Η Σεσίλια Μάστροφη, η υποψηφία επιτρόπος, το υποσχέθηκε αυτό και άλλωστε και εμείς σχετικός ετοιμαζόμαστε τόσο ώστε να μπορέσουμε αυτή την σημαντική ευκαιρία να την έχουμε για την αναθεώρηση αυτών των πρωτοβουλίων. Να μπορέσετε και εσείς να έχετε όλα τα στοιχεία σας και να δείτε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Επομένω αυτό θα είναι αυτού του είδου η κοινή αναθεώρηση τη συμφωνία για τα στοιχεία των επιβατών, κάτι το οποίο θα γίνει σε αμέσως επόμενε εβδομάδες. Ο δικαστή Μπρουγκέρ επίσης, ε, όπως του ζητήθηκε, συντάσσει τώρα αυτή την νέα έκθεση που θα αφορά την ε, λειτουργία του συστήματος SWIFT. Όλα δε αυτά πρόκειται να αποτελέσουν τη βάση για την συζήτηση στο Κοινοβούλιο τώρα. Για τη συμφωνία με τη ΣΥΠΑ. Συμφωνία που συνήφθη τέλη του περασμένου Νοεμβρίου ακριβώς όπως κρίνατε και εσείς ε, πρόκειται για μια ε, σύντομη διάρκεια των 9 μηνών ε, όσον αφορά αυτού του είδους της διατάξης ασφαλείας για το τι θα γίνει εάν δεν υπάρχει άλλη συμφωνία, θα υπάρχουν κάποιοι είδους συμβατικές υποχρεώσεις που θα αναλάβουν και τα δύο μέρη. Όλα αυτά επί τη βάση της ε, απόφασης του Συμβουλίου, της ομόφωνης απόφασης, για αυτή την ροή πληροφοριών που αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την δική μας, για, το, για τη υπό, της δικής ασφάλειας. Γι' αυτό και είναι διαπραγματεύσει και ολοκληρώθηκαν. Και γι' αυτό και είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου προσωρινή ισχύ τη συμφωνία πριν αρχίσει να ισχύει η καινούργια διαδικασία, γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα επιτάσσει η ασφάλειά μα και γι' αυτό και θέλουμε να υπάρχει ένα ούτε παραθυράκι και κενό. Ο δικαστής επομένως ολοκληρώνει τη δεύτερη έκθεσή του και ελπίζουμε στη συνεδρίαση της 4 Φεβρουαρίου να σας κάνουμε τη σχετική παρουσίαση. Να εξασφαλίσουμε ότι το Κοινοβούλιο θα μπορέσουν, το Κοινοβούλιο θα μπορέσει να έχει το, πλήρες κείμενο και επίσης ελπίζουμε ότι από την έκθεση θα αναδειθούν τα εξής δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι οι συνεχίσουν να συμμορφώνονται προς τα όσα έχουν υποσχεθεί για την επεξεργασία των δεδομένων ε, του SWIFT και δεύτερον ελπίζουμε ότι θα προκύψει το ότι η ανάλυση με αυτό το πρόγραμμα αποδίδει πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για πληροφορίες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και αυτό ότι ωφελεί όχι μόνο τη ΣΥΠΑ αλλά και τα κρατη Και τη συζήτηση το Συμβούλιο επίσης αφού προέκυψε πέρσι στη τέλη του χρόνου ότι οι υπηρεσίε πληροφοριών και άλλες διοικητικές αρχές των κρατών μελών πιστεύουν ότι αυτό το πρόγραμμα ενίχνευσης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ακόμα και όταν δεν είναι ακριβώς ε, ε, σαφής η στόχη, είναι κάτι χρήσιμο. Ε, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, βεβαίως και έχετε ακούσει τις ε, εισηγήσεις των Ρέντινγκ και Μάλμστρομ στις σχετικές ακροάσεις τους Περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει το Κοινοβούλιο όσον αφορά την έγκριση της Νέας Επιτροπής. Οπότε... Βεβαίω και βάζετε την επιβάση των απόψεων που ακούσατε και των όσων εσείς είπατε κατά τη διαδικασία των ακροάσεων και έτσι να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τον προγραμματισμό μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ να απαντήσω τις τυχόν ερωτήσεις. Θα ακούσουμε από τα μέλη των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ, ποιος θέλει να μιλήσει. χέρι. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φόλ που είσαστε εδώ μαζί μας για τη συμφωνία SWIFT. Πρέπει να διαχωρίσουμε το περιεχόμενο από τη μορφή του. Εσεί δεν εκπροσωπείτε το Συμβούλιο του ή άλλω και επομένως δεν είσαστε υπεύθυνο για την συμπεριφορά του Συμβουλίου. Επομένως δεν θα τιμωρήσω τον Αγγελιοφόρο. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το περιεχόμενο. Στι 17 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ένα ψήφισμα όπου γράφει ότι ανέμενε από τη Συμφωνία SWIFT. Υπάρχει μια παράγραφο, παράγραφος 2, που λέει ότι η συμφωνία θα πρέπει να αντανακλά την νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία δεδομένων ή να παραπέμψει σε αυτήν την νομοθεσία. Στην παράγραφο 2 υπάρχει και μια υποσημείωση 9 που αναφέρει την νομοθεσία, η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ε, μεταξύ άλλων, είναι η Χάρτα των Θεμελιών Δικαιωμάτων, η Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη 108, η δική μα 95-46 κτλ. Αν δείτε τώρα τα άρθρα της ε, οδηγίας, ε, συμβάσεις, κανονισμοί κτλ. και αν συγκρίνετε όλα αυτά με την συμφωνία SWIFT, θα βρείτε πολλές διαφορές και πολλά σημεία μη συμμόρφωσης. Ένα-δύο έτσι δειγματοληπτικά. Και θα μπορούσα να σας τα μοιράσω αργότερα. Ε, για τα δικαιώματα αυτά δεν συνάδουν με το άρθρο 8 της Χάρτας ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 10, 11, 12 και 14 του 9546, το άρθρο 8 ε, της Σύμβασης 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν συνάδει με το άρθρο 11, 12, 13 και μπορώ να συνεχίσω ΕΣΑΗ e, του κανονισμού 45-2001. Ε, ε, για την περίοδο ε, φύλαξης, για την ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζονται, για την νομική προστασία. Αυτά που δεν, κάποια σημεία που δεν συνάδουν με τη δική μας νομοθεσία. Η συμφωνία συνεχίζει, άρθρα 7, 8 και δεν ξέρω που τελειώνει. Θα βρείτε και εκεί διαφορές τι υπάρχει στη συμφωνία και τι, υπάρχει στο ψήφισμα για την νομική προστασία, την προστασία των δεδομένων κτλ. Απλώς και αν περιοριστούμε στο περιεχόμενο λοιπόν. Ε, και ας ξεπεράσουμε το συνέστημα που έχουμε ότι δεν μας αντιμετωπίζει σωστά το Συμβούλιο. Ε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού αντανακλάται ε, η θέση του Κοινοβουλίου. Ξέρω ότι πέρυσι από τον χρόνο, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για το περιεχόμενο. Έτσι. Ακόμα 20 δευτερόλεπτα το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνει σοβαρή συζήτηση μαζί μας. Γιατί δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το... την προσέγγιση, ας πούμε, του άσπρου μαύρου. Υπάρχει μια εφημερίδα γερμανική που λέει Μπορώ να σας την αναφέρω που λέει, ε, που λέει ε, αναφέρεται σε μια έρευνα ε, ομοσπονδιακή που λέει ότι είναι χρήσιμο το SWIFT. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να εκπλαγείτε με βάση αυτά τα δεδομένα που μπορεί στην ψηφοφορία τα πράγματα να πάνε αλλιώς από ό,τι περιμένετε. Η κυρία Χένις Πλάσχερτ, η συγγήτρια. Ε, δεν θα επαναλάβω τα όσα είπε ο κύριος Άλβαρο. Ε, σωστά είναι αυτά που είπε. Το Κοινοβούλιο ζήτησε, ζητήθηκε μάλλον από το Συμβούλιο να δώσει το Κοινοβούλιο την ε, συνέντευξή του. Θα πρέπει να αναλύσουμε την συμφωνία, έτσι. Εσείς είπατε ότι έχει ασφαλιστικέ δικλείδε για την προστασία των δεδομένων. Ναι, έχει κάποιε για την προστασία των δεδομένων. Κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδε αλλά η... ο ο κ. Άλβαρο δεν υπάρχει νομική προστασία. Υπάρχει πρόβλημα. Το άρθρο 16 δεν υπήρχε, υπήρχε μάλλον σε προηγούμενα σχέδια του SWIFT και τώρα δεν υπάρχει. Και εδώ μιλάμε για δεδομένα Ευρωπαίων ε, πολιτών. Επομένως, θα θέλαμε να εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δικλείδες. Ας πάω τώρα στην ίδια τη συμφωνία. Άρθρο 11.3. Θα ήθελα να μου πείτε τι σημαίνει θα πρέπει... Αν δεν τύχουν σωστή μεταχείριση τα προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη η Αμερικανική νομοθεσία. Τι σημαίνει αυτό για του Ευρωπαίου πολίτε. Θέλω μια εξήγηση. Και θα σταματήσω εδώ, γιατί και πολλοί άλλοι συνάδελφοι θα κάνουν ερωτήσει από το περιεχόμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Μπουσουτήλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είπαμε όλα όσα μπορούσαμε να πούμε για την διαδικασία. Πραγματικά είναι Απαράδεκτοι, δεν, είμαστε δυσαρεστημένοι. Ε, τώρα για την ουσία. Δεν μπορώ να συζητήσω την ουσία εάν δεν μας δοθεί α, πραγματογνωμοσύνη επί τη ουσία. Ε, είμαι κατάπληκτος που ο προηγούμενο ομιλητή ε, έκανε σαφείς δηλώσει ότι υπάρχουν τμήματα της συμφωνίας που δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Εγώ θα ήθελα να μα δοθεί νομική συμβουλή το συντομότερο δυνατόν. Γιατί είναι ο μόνο τρόπο για να μπορέσει αυτή η Επιτροπή να μπει στην ουσία της συμφωνίας με σοβαρότητα, έτσι, και να μην α, συμπεράνει πράγματα επιζήμια. δεν μπορούμε να πούμε ναι ή όχι, χωρίς να έχουμε εξετάσει ενδελεχώς την ουσία. Δεν μ' αρέσουν, δεν είμαι ικανοποιημένο με το βαθμό των πληροφοριών που μας έχει δοθεί. Διάβασα τις πληροφορίες, διάβασα τη συμφωνία. Πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει ε, συμβουλές από εμπειρογνώμονες στο στομό των δυνατών. Ναι, θα υπάρξει μια έκθεση, το σημείωσα, το είπατε, την επόμενη εβδομάδα. Θα τη λάβουμε, αλλά δεν έχουμε χρόνο. Αν θέλετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει σοβαρή απάντηση στο ερώτημα που μας θέτετε, τότε το ελάχιστο που πρέπει να γίνει, και αυτό αφορά όλα τα θεσμικά όργανα, όχι μόνο το δικό μας τελικά, είναι να εξοπλίσετε τους βουλευτές με πληροφορίες, συμβουλές, ούτω ώστε να λάβουν απόφαση με τα λόγω γνώσεως. Ευχαριστώ κύριο Λαμπρινίδης. Συγγνώμη Σταύρο, ξέχασα κάτι. Συγγνώμη, Τζόναθαν. Τζόναθαν Φόλ. Λέτε πάντα ότι υπάρχει ένα χάσμα ασφαλείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, γιατί επί τη βάση των νομικών εργαλείων που έχουμε, έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τις τραπεζικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για αυτές τις έρευνες. Μην ξανασυνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το επιχείρημα για να μας πείσετε να δώσουμε μία άμεση συνένεση, χωρίς πραγματικά να κάνουμε κριτικές ερωτήσεις. Ο Λαμπρινίδης. Ευχαριστώ. Ιωνάθαν, ένα κύκνιο άσμα. Να τελειώνει η καριέρα σας υπερασπιζόμενος εσείς τον κύριο Μπριζιέρ. Καλή τύχη στην επόμενη θέση σας. Λοιπόν, κοιτάξτε. Ο δικαστής Μπριζιέρ υπέβαλε μια έκθεση έκανε, υπέβαλε μια έκθεση πρόσφατα. Έχουμε πολλές εκθέσεις για το πώς εφαρμόζει τη χρήση του PNR οι Ηνωμένε Πολιτείε. Μέσα σε ένα χρόνο, σε λιγότερο από ένα χρόνο, είπατε ότι του ζητήσατε να κάνει μια δεύτερη έκθεση. Ποιο του το ζήτησε αυτό, και το λέω αυτό, Τσόναθα, γιατί πραγματικά είναι εντυπωσιακή η χρονική στιγμή που έγιναν όλα αυτά. Και δίνει την εντύπωση ότι προσπαθούν να μας σπρώξουν με τις εκθέσεις αυτές του κύριου Ρώσια στο να συνενέσουμε σε κάτι που είναι πολύ πολύπλοκο. Ποιος έδωσε και πότε την εντολή στον κύριο Ροζιέρ να κάνει την <clears throat> δεύτερη του έκθεση σε λιγότερο από ένα χρόνο, γιατί την εκδίδει τώρα την έκθεση αυτή. Είχατε πει ότι αυτή η έκθεση θα δοθεί στις 4 Φεβρουαρίου στη δημοσιότητα, αν θυμάμαι καλά. Αλλά είναι 5η-4η Φεβρουαρίου αν τεθεί τότε σε κάποια μυστική αίθουσα στο κοινοβούλιο να τη δούμε, δεν θα προλάβουμε να τη δούμε, γιατί φεύγουμε και μετά είναι η Ολομέλεια και μετά ψηφίζουμε στην Ολομέλεια για το SWIFT. Αυτά λοιπόν δεν στέκονται. Επί της ουσίας, πρώτα απ' όλα θέλω να πω αυτό το οποίο είπε η Ζανίν προηγουμένως. Τι θα γίνει αν το κοινοβούλιο πει όχι σε αυτή τη συμφωνία. Γιατί θα υπάρξει χάσμα ασφάλειας κατά την άποψή σας. Δεύτερον, το άρθρο 3 της συμφωνίας αυτής δεν λέει τίποτα για το SWIFT. Λέει φορείς που έχουν αποφασιστεί από κοινού από τους εμπλεκόμενους φορείς. Δηλαδή φαντάζεστε να χρησιμοποιήσετε και άλλες οντότητες πέραν του SWIFT που θα περιλάβετε σε αυτή την περίπτωση. Όχι, εντάξει, καλό είναι αυτό που μου το λέτε επισήμως. Και ο χρόνος κράτησης των δεδομένων αυτών το άρθρο 5 μη λέει οι πληροφορίες οι οποίες αποκτούνται, <clears throat> οι οποίες ε, εξορίσονται κατά κάποιο τρόπο μέσα από αυτά τα δεδομένα θα υπόκειται σε μία περίοδο φύλαξης που εξαρτάται από την αρμόδια κυβερνητική αρχή. Για τις ΗΠΑ ορισμένες φορές αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι 90 χρόνια για ορισμένες κυβερνητικέ αρχές. Δηλαδή μπορεί να εφαρμοστεί ο χρόνος των ΗΠΑ που μπορεί να φτάσει μέχρι τόσο μεγάλη ε, χρονική διάρκεια. Κύριε Κύρχοφ, κύριε Πρόεδρε, προφανώς το TFTP ισούται με το SWIFT και θα μπορούσε να ισούται και με άλλα θέματα. Αλλά είδατε την επιστολή προς τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, είναι φανερόν ότι αν αυτή η, συμφω... αυτή η επιστολή είναι σωστή, είναι μια προσωρινή συμφωνία η οποία θα επικυρωθεί εν καιρό όταν το Κοινοβούλιο έχει το... την ευκαιρία να τα δει όλα αυτά τα θέματα. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ή βλέποντα την άλλη πλευρά, είναι ένα θέμα όπου μια προσωρινή συμφωνία μπορεί να προχωρήσει χωρί να υπάρχει η έγκριση του Κοινοβουλίου, αλλά αυτό θα πρέπει να επιτρέψει το Κοινοβούλιο να εξετάσει τα θέματα αυτά προσεκτικά και αυτό περιλαμβάνει και την γνώμη των εμπειρογνωμόνων όταν αυτό είναι απαραίτητο και να δώσουμε τη γνώμη μας χωρίς να μας πιέζουν και να μας ζορίζουν. Και ένας μήνας για μετάφραση κύριε Πρόεδρε αυτό είναι αστείο, είναι γελίο. Είναι τελείως παράλογη αυτή η δικαιολογία ακόμα και αν είναι αληθινή. <clears throat> Λοιπόν, δεν μπορείτε να μας πρόχνετε με αυτόν τον τρόπο και να μας πειλατεύετε. Θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να δούμε όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτή τη στιγμή η... δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για την προσωρινή συμφωνία, αλλά χρειαζόμαστε να έχουμε σωστή αντιμετώπιση των δεδομένων για να πάρουμε μια καλή απόφαση. Κύριε Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ. Η νέα αυτή έκθεση του Μπριζιέρ είναι ένα νέο στοιχείο γίνεται όλο και πιο σαφές για μένα γιατί το Συμβούλιο <clears throat> έδρασε με τον τρόπο με τον οποίο έδρασε τις προηγούμενες εβδομάδες. Γιατί μας μένουν ελάχιστες μέρες για να διαβάσουμε αυτές τις εκθέσεις, ουσιαστικά μία μέρα μονάχα. Και εγώ δεν έχω καμία απολύτως εμπιστοσύνη στον τρόπο, στο Συμβούλιο για τον τρόπο που διαχειρίζεται το SWIFT. Και ούτε στον δικαστή Μπριζιέρ έχω καμία εμπιστοσύνη. Γιατί δεν υπήρξε μια συζήτηση για τα θέματα αυτά προηγουμένως. Εγώ διάβασα την έκθεση του δικαστού αυτού και εμένα δεν μου φάνηκε να ήταν ιδιαίτερα αντικειμενική αυτή η έκθεση και απόλυτα τεκμηριωμένη. Και αυτό που είπε ο κύριος Άλβαρο προηγουμένως είναι πράγματι πρόβλημα. Ότι μία από τις υποθέσεις που παρουσίασε σαν παράδειγμα ο δικαστής Μπριζιέρ για τη σημασία του ΣΟΕΦΤ ήταν η περίπτωση Σάουλαντ στη Γερμανία όπου οι ίδιοι οι η ίδια η δικαστική εισαγγελής είπαν ότι δεν ήταν χρήσιμα, δεν ήταν απαραίτητα τα στοιχεία του SWIFT. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί είναι τόσο απαραίτητα τα στοιχεία του SWIFT για να γνωρίσουμε πώς γίνεται η χρηματοδότηση των τρομοκρατών. Και δεν βλέπω ότι έχουμε αρκετά στοιχεία να αποφασίσουμε σε σχέση με αυτό το μέτρο, με τα δεδομένα που μας δίνονται, όπως λέει ο Ισπανός, είπε ο Ισπανός Υπουργός σήμερα το πρωί, παρατείνουμε μια συμφωνία η οποία ισχύει ήδη. Μα σαν να μας κοροϊδεύει το Συμβούλιο, λέει το Κοινοβούλιο. Αυτό κάτι τέτοιο γίνεται. Ο κύριο Σταβάρης. Φτάνουμε σε μια συζήτηση η οποία έχει ήδη μοιαστεί μέσα σε εισαγωγικά από διαθεσμικά προβλήματα. Και αυτά δεν είναι προβλήματα επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να προχωρούμε σε εφημισμούς. Είναι μια απαράδεκτη και ταπεινωτική μεταχείριση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς ζητήσαμε να υπάρχει μια ε, αντιμετώπιση στο πνεύμα της συναπόφασης, στο πνεύμα της Λισαβόνας. Το έχουμε ζητήσει κατά επανάληψη. Υπάρχουν πολλές ασθενείς πτυχές αυτής της συμφωνίας. Αλλά υπάρχουν τα τρία ισχυρά σημεία τα οποία μας παρουσιάζει συνέχεια για το SWIFT. Πρώτον ότι είναι προσωρινή συμφωνία. Όχι, δεν είναι προσωρινή. Τουλάχιστον για πέντε χρόνια θα κρατηθούν αυτά τα στοιχεία. Μέχρι ότου έρθει η επόμενη ε, Αμερικάνικη κυβέρνηση και η οποία μπορεί να μην είναι τόσο προεκτήσεκτική για τα δεδομένα των Ευρωπαίων. Δημιουργεί μια ισορροπία δύναμης και εξουσίας που δεν θα είναι η καλύτερη όταν πρέπει να διαπραγματευτούμε μια νέα συμφωνία. Δεν είναι να διαπραγματευτούμε με τους Αμερικανούς και είναι ακόμα λιγότερο όταν έχουμε ήδη θεσπίσει αρνητικέ πρακτικέ. Λέγεται ότι χρειάζονται αυτά τα στοιχεία επειδή υπάρχει χάσμα ασφάλεια. Το αντιμετώπισε η Ζωανίν Πλάσκετ το θέμα αυτό. Υπάρχει πάντα δικαστική οδό για να αποκομίσει κανεί πληροφορίε για τέτοιε οικονομικέ δόσει όληψίε. Ο αγώνα για την κατάσταση τη τρομοκρατία δεν θα σταματήσει χωρί αυτή τη συμφωνία. Οι εκθέσει του δικαστού Μπρουγκέρ. Εγώ δεν μου αρέσει ο τρόπος που αναφέρθηκαν όλα αυτά. Υποτίθεται ότι είναι μια μυστική έκθεση και παρουσιάζεται σαν να είναι η απόδειξη ότι είναι απαραίτητα τα στοιχεία του SWIFT για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία. Εγώ τη διάβασα αυτήν, θα ήθελα να αναφερθώ σε απόλυτα στοιχεία αυτής της έκθεσης, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι Αμερικανοί θα χρησιμοποιήσουν καλά αυτά τα στοιχεία και δεν υπάρχουν καθόλου εμπειρικά στοιχεία που να παρουσιάζονται ότι ήταν χρήσιμα αυτά τα στοιχεία. Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι τα στοιχεία αυτά ήταν ε, απα, απαραίτητα. Είναι μια σαθρή η πρώτη έκθεση Μπρουγκέρα και η δεύτερη έκθεση υποτίθεται ότι θα αποδείξει κάτι το οποίο δεν απέδειξε η πρώτη έκθεση. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τυφλά και ασθενή στοιχεία. Παρακαλώ κλείστε. Όχι, για αυτά είναι σημαντικά κύριε Πρόεδρε. Ναι, φυσικά είναι σημαντικά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν έρευνε για τι τρομοκρατίες. Αλλά εδώ έχουμε πληροφορίες οι οποίες αφορούν κατά 90% Ευρωπαίους πολίτες και επιχειρήσεις που δεν είναι τρομοκράτε. Και η Επίτροπος Ρέντινγκ μας είπε πώς θέλει να διαπραγματευτεί. Μας έδωσε τις γενικές γραμμές και νομίζω ότι είναι θετικό αυτό. Μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη συμφωνία και ίσως αν το Κοινοβούλιο απορρίψει αυτή τη συμφωνία θα κάνει για μια χάρη σε όλους. Όλοι κατανοείτε ότι η διαχείριση του χρόνου δεν έχει καμία σχέση με τη σημασία του θέματος αυτού. Απλώς προσπαθώ να σεβαστώ την ημέρησια διάταξη και το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό δεν έχει τίποτα να κάνει με το ζήτημα το συγκεκριμένο. Βίβα. <coughs> Νομίζω ότι κάνουμε περιγέλαστο και πάλι το, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν ακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση, θα πρέπει να συμμετάσχουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να φτάσουμε σε μία σοβαρή συζήτηση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως έχουν πάει τα πράγματα μέχρι στιγμής. Και μία σοβαρή συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μονάχα γύρω από τα διαδικαστικά θέματα. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία με τις ΗΠΑ και είναι ζωτική για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και θα πρέπει να υπάρξει η εξέταση σε επίπεδο περιεχομένου. Δύο ερωτήματα. Το κενό, το χάσμα αυτό ασφαλείας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ακόμα σήμερα, χωρίς συμφωνία για το SWIFT, εξακολουθεί να υπάρχει η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών. Αν δεν εκριθεί αυτή η συμφωνία θα σταματήσει η συνεργασία. Και το δεύτερο κεντρικό θέμα. Αν μιλάμε για την μελλοντική, την οριστική ε, συμφωνία που θα πρέπει να τύχει διαπραγμάτευσης, θεωρείτε ότι αν πούμε εμείς ναι στην προσωρινή συμφωνία ότι υπάρχει μια δυνατότητα η προστασία των Ευρωπαίων πολιτών να βελτιωθεί σε μια μακροχρόνια συμφωνία. Ή θα πούν οι Αμερικάνοι αφού είπατε ναι στην τωρινή συμφωνία δεν χρειάζεται να διαπραγματευτούμε κάτι άλλο. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε μια μακροπρόθεσμα, μια συμφωνία που θα είναι καλύτερη για τους Ευρωπαίους πολίτες. κυρία Ιντβελτ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπε ο κύριο Βέμπερ, όχι όλα. Δεν είναι διαδικαστικά αυτά τα πράγματα που συζητούμε. Είναι ουσιώδη. Έχουν να κάνουν με το δημοκρατικό έλεγχο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ελέγξει τις εξουσίες του, του δημοκρατικού ελέγχου πλήρως, εάν έχει πρόσβαση σε όλε τι πληροφορίε. Και υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θέλω να τονίσω εδώ. Πρώτον, ότι χρειαζόμαστε πρόσβαση στη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Είναι ένα κεφαλαιόδε στοιχείο για την εξέταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χωρίς αυτή την έκθεση εγώ δεν μπορώ να ασκήσω κοινοβουλευτικό έλεγχο πλήρως. Δεύτερον, η δεύτερη έκθεση Blue εγώ είμαι εμβρόντιτη γιατί μιλάμε για το SWIFT εδώ και έξι μήνες από τον προηγούμενο Ιούλιο και ποτέ δεν μας είπαν ότι προετοιμαζόταν μια νέα έκθεση. Εγώ εντυπωσιάζομαι από το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Κομισιόν και το Συμβούλιο κράτησαν σιγή ηχθείως και τέλος μια φιλοσοφική παρατήρηση αν μου επιτρέπετε. Η Ευρώπη είναι ένα ιδιότυπο σου γένερης οικοδόμημα. Αλλά πρέπει να πω ότι εδώ βλέπω να υπάρχουν κάποιες παραλληλίες και ομοιότητες με εθνική πολιτική αν μια κυβέρνηση αρνηθεί ή αποτύχει να πληροφορήσει το Εθνικό της Κοινοβούλιο σε τέτοιο επίπεδο, θα είχε εκδιωχθεί. Εγώ λοιπόν βρίσκω απαράδεκτο αυτό το οποίο γίνεται. Κύριε Στράσε. Πάρα πολύ σύντομα και εμφαντικά να πω στον ε, Γενικό Διευθυντή και τους συνεργάτες τους ότι έχω κριτικές παρατηρήσεις λόγω της πολιτικής ουσίας του θέματος αυτό ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου έχει ζητήσει από το Συμβούλιο και την Κομισιόν να, εξασφαλίσει, να εξασφαλίσουν το ότι η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει στο Κοινοβούλιο να κάνει μια σοβαρή και πλήρη εξέταση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι αυτή η απόλυτα θεμητή αίτηση του Κοινοβουλίου να μην τύχει ανταπόκριση από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Δεύτερο, για το κενό ασφάλειας. Εάν υπήρχε ένα τέτοιο κενό ασφαλείας, αυτή είναι η στιγμή που το έχετε. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Ιανουαρίου τουλάχιστον. Και αν υπήρχε ένα τέτοιο κενό, να, τώρα γίνεται αυτό το πράγμα. Και παρόλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν. Πού ακριβώς είναι το πρόβλημα λοιπόν. Τρίτον, για το περιεχόμενο. Εμείς, τα μέλη της Επιτροπής πολιτικών ελευθεριών, δεν είμαστε σίγουροι αν έχουμε ακόμα το πλήρες κείμενο στα χέρια μας. Θα το ξέρουμε αυτό μόνο την τελευταία στιγμή να ξέρουμε αν έχουμε πράγματι όλο το κείμενο, όλα τα παρατήματα, όλες τις ε, σχολιάσεις, αν έχουμε όλα τα νομικά στοιχεία στο τέλος. Το Κοινοβούλιο όμως έχει το δικαίωμα, εφόσον συναποφασίζει, να έχει τις πλήρες πληροφορίες για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση και η δική μου βάση για μια απόφαση σε αυτή τη συμφωνία είναι καταρχήν το ψήφισμα του Κοινοβουλίου στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2009. Αυτό είναι, αυτός είναι ο γνώμονας για την στάθμιση θέση από μας. Και τρίτον, όλα αυτά τα οποία ακούμε εμείς ανεπίσημα δείχνουν ότι τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στην αρχή των διαπραγματεύσεων έχουν ξεπεραστεί. Αυτό είναι θετικό και θα χαρώ αν μπορέσουν να ξεπεραστούν και άλλα στη συνέχεια. Μας είπανε. Το σύστημα διαρμηνίας συνένεσε σε 10 λεπτά ακόμα για την Επιτροπή μας να καλύψουμε το θέμα αυτό το οποίο συζητούμε. Σας παρακαλώ και πάλι να κάνετε καλή χρήση αυτού του πρόσθετου χρόνου 10 λεπτών. Ο κύριος Μπουταρέλη θα πρέπει να λάβει το λόγο τώρα για 5 λεπτά για να συνοψίσει την νομική γνωμοδότηση η οποία έχει δοθεί σε όλα τα μέλη της Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι τεχνική και νομική πληροφόρηση που έχει ζητηθεί για μια σειρά από τα θέματα αυτά. Θα ακούσουμε λοιπόν ε, τον κύριο Μπουταρέλη και θα έχουμε την τελική απάντηση του Τζόναθαν Φόουλ από την Κομισιόν. Κύριε Μπουταρέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε. Πέραν κάποιων διαδικαστικών, τα οποία τώρα δεν θα με απασχολήσουν, τα περισσότερα από όσα ακούσαμε σήμερα αναφέρονται στην προστασία του ιδιωτικού βίου και της ασφάλειας σωστά. Όλα αυτά θεωρούνται από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ως σημαντικά και έχω να σας πω ότι όλα αυτά με μεγάλη προσοχή έχουν ληφθεί υπόψη ένα προς ένα σε αυτό το έγγραφο το οποίο πριν από λίγες μέρες σας διαβιβάστηκε. Αυτό το έγγραφο το οποίο έχει να κάνει σε ένα συμπέρασμα σύντομο αλλά σαφές. Επίσης όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχετε λάβει και το EDPS αναδεικνύει κάποια στοιχεία τα οποία δικαιολογούν το ότι θα πρέπει να συναυθεί μια τέτοια συμφωνία. Έχουμε εδώ εν μέρει επικάλυψη με τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, υπάρχουν κάποια θέματα αυτής της συμφωνίας τα οποία ακόμα δεν έχουν περικαραδοκωθεί αρκετά ούτως ώστε να έχει ξεχαθαστεί τελείω το ποια δεδομένα διαβάζονται τη ΣΥΠΑ. Οπότε, εάν αρθούν αυτές όλες οι ασάφειες, θα έχουμε βελτίωση της προοπτικής για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία. Όμως είναι πάρα πολλά τα σχετικά σημεία αυτά. 16 τουλάχιστον μπορεί κανείς να επισημάνει τέτοια σημεία σε σχέση με άλλα κείμενα σχετικά που αφορούν δηλαδή τον εντοπισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων της τρομοκρατίας, οικονομικής υποστήριξης, όπως ας πούμε τα νομοθετήματα που έχουμε για το ξέβλημα χρήματος. Ούτε θεωρούμε ότι υπάρχει κάποιο είδου ε, συσχετισμό μεταξύ αυτών των ε, δεδομένων που ε, επεξεργαζόμαστε. Γιατί τα συλλέγουμε σε εδώ τα δεδομένα και τα διαβάζουμε στους Αμερικανούς. Οπότε, σε αυτό το έγγραφο τονίζουμε το θέμα της ποιότητα των δεδομένων και του σκοπού τον οποίο χρησιμοποιούνται. Και είπαμε ότι υπάρχουν κάποιε δυσκολίε εφαρμογή του άρθρου 4 τη ενδιάμεση προσωρινή συμφωνία σε σχέση με το άρθρο 8 τη Συμφωνία Αμοιβαία Αρρωγή που έχουμε συνάψει με τι ΗΠΑ. Και θέλουμε να υπάρχει κάποιο του δικαστικό έλεγχο. Επίσης, άρθρο 4 παράγραφος 6 θα πρέπει και εδώ να σταθούμε σε σχέση με τη διαβίωση των δεδομένων. Επίσης, στο άρθρο 2 είναι ευρύτερος ο ορισμός, ευρύτερος του άρθρου 1 της απόφασης του 2002 για κατά της τρομοκρατίας. Επίσης, φύλαξη επί πέντε χρόνια κάποιων δεδομένων και είπαμε ότι δεν δικαιολογείται ε, το, το, επί τόσο χρόνο κράτηση, φύλαξη, αποθήκευση των δεδομένων γιατί προκύπτει ότι ό,τι δεδομένα δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν για δίωξη δημοκρατία, να εξαλείφονται, να καταστρέφονται και επίση θα πρέπει να υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων και με τρίτες χώρες. Τώρα, όσον αφορά το άρθρο 11, κάτι το οποίο τόνισε ο συγκητής, έχουμε εδώ τουλάχιστον τρεις δυσκολίες όσον αφορά την εφαρμογή της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου. Γιατί η παράγραφος 1 του άρθρου 11 δεν παρέχει εγγύησεις και στις ΗΠΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, με αυτή τη διάταξη έχουμε ενδεχόμενους περιορισμούς ε, ούτως ώστε να μπορούν οι αρχές να κάνουν αυτούς τους ελέγχους γιατί ε, εδώ πέρα η... είναι δυσνόητο το άρθρο, δεν προκύπτει κάποια λογική δομή του και είναι κάτι που δεν έχει και προηγούμενος αρρύθμιση. Διόδος πληροφοριών, αποζημίωση για παράνομη εξασία δεδομένων. Εδώ πάλι απουσιάζει συγκεκριμένος τρόπος εφαρμογής της διάταξης. Και άρα βλέπουμε ότι θα πρέπει Και πάλι τονίζουμε το ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί υπάρχει αυτή η μνήμα στο άρθρο 16 σαν νομική βάση. Να απαλληφθεί λέμε. Επίσης, και θα πρέπει είπαμε, να ληφθούν υπόψη και, άλλες, και, και, άλλα, και άλλες συμφωνίες για το Μητρό Πληροφοριών των Επιβατών. Thank you so much, Mr. Butarelli, for the information that you've just shared with all of us. Σα Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Ο κύριος Τζόναθαν Φόλ. Ευχαριστώ. Ζητώ που θα απογοητεύσω το Σταύρο Λαμπρινίδα. Δεν θα, μάλλον δεν θα είναι τελευταία μου εμφάνιση στην Επιτροπή σας. Δεν ξέρω πότε θα πάω το νέο μου πόστο. Αλλά μπορεί να μην γίνει όσον νούπο. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το τέλος τώρα. Και να αναφέρω κάτι που είπε ο κ. Βέμπερ και άλλοι. Θα συνάψουμε καλύτερη συμφωνία στο μέλλον. Το ελπίζω. Πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτή την βραχυπρόθεσμη διάταξη με μία πιο πλήρη και πιο μακροπρόθεσμη συμφωνία με βάση τις διατάξεις της νέας συνθήκης, της Συνθήκης Λισαβόνας. Αυτό όμως θα το διαπραγματευτεί η Κομισιόν με βάση τις νέες διατάξεις με την πλήρη υποστήριξη, ελπίζω, του Κοινοβουλίου και θα προκύψει ε, μια συμφωνία που το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποδεχτούν. Δεν θα είναι εύκολο. Όσοι έχουμε εμπλακεί και ειδικά οι Σουηδοί φίλοι μου στις διαπραγματεύσεις ε, με τους Αμερικανούς στις περσινές διαπραγματεύσεις ξέρουν πόσο δύσκολο είναι, αλλά θα γίνει. Και όλοι όσοι μίλησαν για αυτό το θέμα, και ο Μπουταρέλη και άλλοι, Όλα αυτά τα σημεία που ανέφεραν θα ληφθούν υπόψη. Ελπίζω λοιπόν, εγώ δεν θα είμαι αυτός που θα συνεχίσει σε αυτό το πόστο, αλλά η νέα Επιτροπή με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου ελπίζω ότι θα φτάσουν σε μια καλύτερη συμφωνία. Και του Συμβουλίου βεβαίω, να μην το ξεχνάμε, και το Συμβούλιο. Αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί σήμερα. Σήμερα μιλάμε για την παλιά συμφωνία της 30ης Νοεμβρίου. Ε, που είναι μια προσωρινή συμφωνία έτσι για να καλυφθεί το κενό. Ε, για αυτήν θέλουμε να συνενέσετε. Θα ισχύσει για 9 μήνες και κατά τη διάρκεια αυτών των 9 μηνών θα πρέπει να ξεκινήσουμε τις προετοιμασίες για τη νέα συμφωνία. Τώρα, έρχομαι στα φιλεγόμενα θέματα που θίξατε. Ε, ξέρω δεν έχω χρόνο. Δέκα λεφτά, το πολύ. Θα κάνω την μπορώ μέσα σε 10 λεπτά. Γι' αυτά που είπε ο κύριος Άλβαρο. Ειλικρινά σας λέω, δεν συμφωνούμε. Το Συμβούλιο δεν συμφωνεί ότι η συμφωνία δεν συνάδει με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αλλιώς δεν θα είχε συναυθεί αυτή η συμφωνία, το Συμβούλιο δεν θα την είχε συνάψει και δεν θα την είχαμε βάλει σε εσά για να μας δώσετε τη συνένεσή σας. Αλλά αυτό είναι θέμα εντάξει, νομικής γνωμοδότησης. Αυτή πάντως είναι η άποψη της Κομισιόν. Γιατί η Κομισιόν δεν αντιτάχθηκε στο να φτάσει σε αυτή τη συμφωνία το Συμβούλιο ομόφωνο, όπως ξέρετε. Η άποψη της Κομισιόν μάλιστα ήταν ότι συνάδει αυτή η συμφωνία με όλα τα εφαρμοστέα μέτρα του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί δεν θα υπήρχε αυτή η συμφωνία ενώπιό σα. Μπορεί να έχετε διαφορετική γνώμη, θα δούμε πώς ε, θα, προχωρήσουν τα πράγματα, αλλά αναμφίβολα η Κομισιόν θα έκρινε κάτι και ελπίζω και το Συμβούλιο να μην έκρινε κάτι το οποίο δεν ε, συμμορφωνόταν με το ευρωπαϊκό δίκαιο και ιδιαιτέρως με τα ευρωπαϊκά θεμελιώδη δικαιώματα. Το άρθρο 16 που ανέφεραν πάρα πολύ. Αυτό ελπίζω να μπορώ να σας το διεκπαιρεώσω σύντομα. Ήρθαμε σε επαφή με τους δικηγόρους μας, κοιτάξαμε όλο το θέμα της νομικής βάσης που είναι δύσκολο ε, σε αυτόν τον τομέα. Ξέρουμε το ιστορικό, ξέρουμε το... την κόδρα Κοινοβουλίου Συμβουλίου για το... την νομική βάση του PNR ε, και στον τομέα της εφαρμογής του δικαίου. Μία συμφωνία για την ανταλλαγή δεδομένων είναι τι είναι, ε, ασφάλεια, ε, τρομοκρατία κτλ. Στο, στα παλιά δεδομένα ήμασταν στον τρίτο πυλώνα. Με τα νέα δεδομένα τώρα, λένε οι δικηγόροι μας, πιστικά νομίζω, ότι η κατάλληλη νομική βάση είναι στα άρθρα 82 και 87 τζάι στις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 16 είναι μια συγκεκριμένη νομική βάση για συγκεκριμένα θέματα προστασίας των δεδομένων. Είναι και θα είναι η νομική βάση εν ευθέτω χρόνο για τη γενική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που η Βίβια Ρέντινγκ, η υποψήφια αντιπρόεδρος και επίτροπος, σας είπε ότι θα είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κομισιόν στο εγγύς μέλλον. Δηλαδή μια αναθεώρηση όλων των νομοθετημάτων της προστασίας δεδομένων. Άρθρο, λοιπόν, αυτό το άρθρο 16 είναι η κατάλληλη νομική βάση. Αυτή είναι η άποψη των νομικών μας και του Συμβουλίου. Και ακριβώς γι' αυτό, αλλά μην δίνετε πολιτική σημασία σε αυτό, γι' αυτό νομίζω, λέγω, επελέγει, ε, δεν συμπεριληφθήκε η νομική βάση του 16. Τώρα, το κενό ασφάλειας. Ορισμένοι είπαν ότι χρειάζεται πραγματογνωμοσύνη. Θέμα δικό σας θέμα δικό σας, πώς θα ενημερωθείτε από εμπειρογνώμονες και τα λοιπά στην Επιτροπή σας. Εγώ όταν μίλησα για το κενό δικαίου, ε, κοινό ασφάλειας μάλλον, εννοούσα το εξής, ότι αυτό το θέμα και το θέμα της ε, ε, οικονομικής, του οικονομικού εντοπισμού τρομοκρατών είναι απαραίτητο για την ασφάλεια. Ε, αυτό είναι το προήμιο από το οποίο ξεκινάμε, ότι χρειάζεται για την ασφάλεια. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία χρονική περίοδος, μακρά ή όχι, ε, κατά την οποία δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα. Τώρα, τι θα γίνει αν το κοινοβούλιο πει όχι. Αν το κοινοβούλιο πει όχι, φαντάζομαι ότι το Συμβούλιο θα ενημερώσει τη ΣΥΠΑ ότι δεν ισχύει συμφωνία. Δεν θα τεθεί α, σε ισχύ. Ε, καμιά φορά και η Γερουσία, η Αμερικανική, αποφασίζει τέτοια πράγματα. Έχει ξαναγίνει. Επομένω δεν θα, δεν ισχύσει συμφωνία. Πολύ ωραία θα ισχύει συμφωνία. Τι θα έχει συμβεί στην πράξη, και εδώ η, η κατολόγω. Μπορώ να φανταστώ ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε επειδή πιστεύουν, όπως και εγώ, ότι αυτό είναι σημαντικό θέμα για την ασφάλειά τους, θα συνεχίζουν να αναζητούν αυτές τις πληροφορίες. Επομένως, θα χρησιμοποιούν τους συνήθεις μηχανισμούς αμοιβαία νομικής αρρωγής, ε, τη δυνατότητα κλήτευσης που προβλέπει το Αμερικανικό Δίκαιο για να αναζητήσουν πληροφορίες από το SWIFT. Θα, θα εξηγήσω γιατί, λέμε, ε, γιατί το λέμε SWIFT Δεν το αναφέρουμε αυτό συμφωνία. Θα βρουν άλλους τρόπους να βρουν αυτές τι πληροφορίε. Αυτό σημαίνει κλήτευση. Θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν την αρχή της κλήτευσης ε, στα, σε κράτη-μέλη που συνδέονται με τέτοια θέματα και το ευρωπαϊκό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων θα ισχύσει. Αυτό που δεν θα ισχύσει είναι οι συγκεκριμένες διατάξεις προστασίας των δεδομένων που οι Ηνωμένε Πολιτείε αναδεσμεύτηκαν ε, ότι θα σεβαστούν στη ΣΥΠΑ. Αυτό δεν θα υπάρχει. Θα εξαφανιστεί. Θα εκλείψει. Όλες οι διατάξεις που έχουμε συμπεριλάβει στη συμφωνία για αυτή την περίοδο δεν θα ισχύσουν. Επομένως, θα υπάρξει ένα κενό ασφαλείας ή ένα κενό προστασία των δεδομένων. Αλλά αποκλείεται να έχετε την πλήρη κάλυψη που εξασφαλίζει η συμφωνία. Για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Γιατί αναφέρεται το SWIFT. Γιατί δεν θέλουμε να αναφέρεται. Το SWIFT δεν θέλει, δεν είναι καλό να δημοσιοποιείται, να υπάρχει διαφήμιση γύρω από αυτό <coughs> και προτιμήσαμε και οι Αμερικάνοι το δέχτηκαν να χρησιμοποιήσουμε μια διαφορετική ονομασία, έτσι, να το παρακάμψουμε, να μην αναφέρουμε το SWIFT. Αναφέρουμε άλλους φορείς και τα λοιπά, αντί για το SWIFT. Αλλά το SWIFT είναι το κυρίαρχο, ας πούμε, πλαίσιο δεν μπορώ να σας μιλήσω για τις διαδικασίες, ε, το πόσο χρόνο χρειάζονται οι μεταφράσεις. Ξέρω από τη δική μου τη δουλειά, το ξέρετε κι εσείς, ότι είναι δύσκολη η ιστορία οι μεταφράσεις και παρά την προσπάθεια των μεταφραστών να δουλέψουν πιο γρήγορα, ε, έχουν κάποια όρια. Ε, δεν υπάρχει συνωμοσία πάντως. Κανένας δεν θέλει να ταπεινώσει κανέναν. Είναι λεπτό θεσμικό θέμα ανάμεσα τρία θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαβαίνουν όλοι ότι ήμασταν σε μια λεπτή χρονική στιγμή, η Λισαβόνα, λεπτή στιγμή στις διατλαντικέ σχέσεις. Εσείς καταλαβαίνετε, είσαστε πολιτικοί, εγώ δεν είμαι. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε πολύ. Γίνεται και μια, ένας διάλογος εκτός μικροφώνου. Ούτε σε εγώ δεν είμαι πολιτικό, δεν με έχει επικυρώσει κανένα εκλογικό σώμα, έτσι. Αλλά νομίζω ότι απόκειται σε όλους μας, ο καθένας με τον τρόπο του, να βρούμε λογικούς τρόπους για να προχωρήσουμε. Χωρίς να δημιουργήσουμε ε, ούτε εσωτερική ούτε διεθνή κρίση. Α, για τον δικαστή Μπρουγκέρ. Ε, είχε ένα συμβόλαιο δύο χρόνια για την έκθεση. Το ήξερε το Κοινοβούλιο. Αυτή η σύμβαση νομίζω λύγει τον Απρίλιο του 2010. Επομένως, λογικό είναι. Και κανένας δεν έκανε καμία... Κάτι το απρεπές εδώ. Ε, σωστό είναι να κάνει μια, ένα δεύτερο γύρο πούμε, ερευνών για να καταλήξει μια δεύτερη έκθεση και νομίζω θα τη βρείτε χρήσιμη κι εσείς για να μπορέσετε να καταλήξετε στη συνένεση που σας ζητούμε για τη συμφωνία. Και για να προβληματιστείτε εν γέννη για το, την οριστική συμφωνία SWIFT που θα την διαπραγματευτούμε αργότερα. Προσπάθησα να είμαι λακωνικός. Ξέρω δεν απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και άρα απογοήτευσα κάποιους. Αλλά είναι μια συμφωνία που διαπραγματεύθηκε ε, καλή την πίστη μετά το ψήφισμά σας του 2009, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που κάνατε στο ψήφισμα. Η άποψη του Κοινοβουλίου τώρα είναι ότι και τις συμμερίζεται η Κομισιόν. Ότι συνάδει με το ευρωπαϊκό δίκαιο και με τις υψηλές αξίες και πρότυπα ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα βελτιωθεί την επόμενη φορά. Ας προσπαθήσουμε να την κάνουμε καλύτερη αυτή η συμφωνία την επόμενη φορά. Ούτως ή άλλως θεσμικά ε, είμαστε πιο έτοιμοι τώρα, καλύτερα υψοπλισμένοι για κάτι τέτοιο. Πάντω τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ε, και η ΕΠΑ θεώρησαν ότι αυτή η προσωρινή εννιάμινη συμφωνία ήταν σημαντική. Και πιστεύουμε και εμεί, από πλευρά Κομισιόν ότι πρέπει να προχωρήσει. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για όλη τη δουλειά, όλη την προσπάθεια που κάνετε για να ολοκληρώσετε για, μέσα σε δέκα λεπτά. Ο κ. Μπουταρέλη, μισό λεπτό. Συμφωνώ απόλυτα ότι αν δεν το δεχτεί το Κοινοβούλιο, οι ρήτρε προστασίας δεδομένων και οι εγγυήσει μπορούν να εξαφανιστούν. Όπως είπατε όμως, οποιαδήποτε μεταφορά δεδομένων σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να καλύπτεται και να ρυθμίζεται από, τις εθνικές, από τους εθνικούς κανόνες προστασίας δεδομένων που εδώ πρέπει να είναι πολύ πιο αστηροί από αυτούς που συζητούμε τώρα. Είναι διάφορα τέτοια στοιχεία που θα βοηθήσουν να αξιολόγησή σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο μας. Κάναμε πολλή εργασία. Θέλουμε να σα ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία σα για να τα κάνουμε όλα αυτά να λειτουργήσουμε.